Okay, suggest we, um, we start today's session. Welcome. Συνάδελφοι, προτείνω να ξεκινήσουμε. Είναι η ακρόαση για την ηλεκτρονική παρακολούθηση. Θα ακούσουμε ε, δύο ομάδες ομιλητών. Όπως ξέρετε, η πρώτη με δύο ομιλητές και η δεύτερη με θέμα το whistleblowers, τους, τις διαρροές πληροφοριών, απόρριτων πληροφοριών. Θα έχουμε διάφορους εκπροσώπους αμερικανικών οργανώσεων για την προστασία των ε, δημόσιων ελευθεριών. Θα δώσω το λόγο καταρχήν στον Μάρκ Ρότενμπεργκ, ο οποίος δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται εδώ στο Κοινοβούλιο και παίρνει το λόγο, καθόπιν η Κάθριν Κραμπ από την ε, Αμερικανική Ένωση Ελευθεριών και φυσικά κατόπιν θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, μέλη της Επιτροπής, ε, φίλοι και προσκεκλημένοι και εσείς από την Εθνική Υπηρεσία ε, Ασφάλειας, την NSA της Αμερικής που μπορεί να διαβάζετε το ε, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και γνωρίζετε ότι είμαι εδώ. Εμείς είμαστε ένας ερευνητικό οργανισμός ο οποίος δεν έχει καμία πολιτική συνάφεια στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν δεχόμαστε χρηματοδότηση από καμία ε, κυβερνητική υπηρεσία και ούτε και από καμία ιδιωτική επιχείρηση. Προσπαθούμε να εκπροσωπήσουμε τις απόψεις των χρηστών ε, του διαδικτύου σε θέματα ε, προσωπικών δεδομένων και πολιτικών ελευθεριών. Συνεργαζόμαστε βέβαια με οργανώσεις ε, ε, οι οποίοι προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα και ασχολούνται με τα θέματα της πολιτικής ε, ε, ελευθερίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και με πανευρωπαϊκούς οργανισμούς που ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε μια πολύ σχηματική διάσκεψη στη Βαρσοβία στην Πολωνία με τίτλο «Τα δεδομένα μας, τα στοιχεία μας, οι ζωές μας». Και αυτό ήταν η προστασία της ιδιωτικής ζωής στο σύγχρονο κόσμο. Μου ζητήσετε να σας εκφράσω τις απόψεις των ε, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στις Ηνωμένε Πολιτείες. Θα κάνω κάποιες παρατηρήσεις για να σας πω τι έχουμε επιτύχει, τι θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει περαιτέρω και κατόπιν να σας ε, ζητήσω να αναλάβετε συγκεκριμένες δράσεις. Καταρχάς να σας πω ότι από την 11η Σεπτεμβρίου και μετά οι οργανώσεις ε, των πολιτικών ελευθεριών στις Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάστηκαν προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη λογοδοσία και έλεγχος για τις ε, εποπτικές αρχές οι οποίες έχουν ε, συσταθεί με νομοθεσία όπως το Patriot Act, ε, νέα συστήματα και βιομετρικά δεδομένα και άλλα αντίστοιχα νομοθετήματα και άλλες μορφές παρακολούθησης και εντοπισμού ατόμων εντός των ΗΠΑ. Είχαμε κάποιες επιτυχίες, βέβαια είχαμε και κάποιες αποτυχίες. Κάποιες διατάξεις του νόμου Patriot τροποποιήθηκαν χάρη ε, στην παρέμβασή μας και κάποια πράγματα όμως επεκτάθηκαν σε πράγματα τα οποία δεν ε, θεωρούμε ότι ήταν σωστά. Μας υπογοήτευσε ιδιαίτερα το γεγονός ότι το Κογκρέσο αποφάσισε να επεκτείνει αυτή την νομοθεσία η οποία στόχο είχε αρχικώς να επικεντρωθεί στο ε, θέμα της παρακολούθησης ε, ξένων κατασκόπων που δραστηριοποιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτό διευρύθηκε σε μια πολύ ευρύτερη κατηγορία συλλογής ε, στοιχείων από ό,τι θεωρούμε ότι θα έπρεπε να επιτρέπεται. Παρά τις καθυστερήσεις μας λοιπόν και από κάποιες επιτυχίες που είχαμε, Τίποτα δεν μας είχε προετοιμάσει για το έγγραφο το οποίο αποκαλύφθηκε στις αρχές ε, του καλοκαιριού από τον κύριο Σνόντεν. Ήταν μια διαταγή την οποία είχε εκδώσει το Εποπτικό Συμβούλιο στις ΗΠΑ που υποχρέωνε την τηλεφωνική επιχείρηση Verizon να δώσει όλα τα τηλεφωνικά αρχεία, όλα τα στοιχεία για όλους τους πελάτες της σε συνεχή βάση χωρίς καμία εξαίρεση απλώς και μόνο για τις επικοινωνίες εσωτερικού. Εγώ ασχολούμαι με θέματα προσωπικών δεδομένων και ιδιωτική ζωής εδώ και 20 χρόνια. Ποτέ δεν έχω δει ένταλμα το οποίο να δίνει τόσο μεγάλες εξουσίες. Και το γεγονός ότι ήταν ε, όλα αυτά απόρριτα και δεν υπήρχε δυνατότητα να αμφισβητήσει κανείς ε, το ένταλμα και να ζητήσει κάποια αιτιολόγηση ε, έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου στις οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών. Ε, είχε ξεκινήσει μια πολύ σημαντική διαμάχη που έφτασε και στο ανώτατο δικαστήριο το προηγούμενο χρόνο και αναγνώριζε, όπως και εμείς, ότι το συγκεκριμένο ένταλμα ήταν παράνομο. Ε, έγιναν ενστάσεις ε, από πλευράς τους ε, στο δικαστήριο στη Νέα Υόρκη. Εμείς πήγαμε κατευθείαν στο ανώτατο δικαστήριο. Κάποιοι μας είπαν για ποιο λόγο υποβάλλεται αγωγή. Μπορεί κάλλιστα ένα δικαστήριο να εκδώσει εντάλματα για να συλλόξει στοιχεία. Ναι, αλλά θα πρέπει να έχει εξουσιοδότηση και αυτό να βασίζεται σε μια συγκεκριμένη νομική βάση. Όταν αναζητούν τόσο μεγάλο εύρος στοιχείων ε, και θεωρούν ότι έχουν αυτή την εξουσιοδότηση, το δικαστήριο ε, θα πρέπει να έχει ε, κάποια νομική βάση να το στηρίξει. Πολλοί καθηγητές νομικής, ακόμα και η δικαιοδοσία ίδια του ανωτά του δικαστηρίου υπέβαλαν ε, στοιχεία και εκθέσεις στηρίζοντας την αγωγή μας και λένε ότι θα πρέπει πραγματικά να δοθεί ε, μία μάχη, να υπάρξει δίκη γιατί το ένταλμα αυτό είναι παράνομο και πρέπει ε, να απαγορευτεί. Υπάρχουν πολλοί τρόποι στις Ηνωμένες Πολιτείες ε, για να ανταποκριθεί στο γεγονός ότι όλοι γνωρίζουν ε, πλέον πόσο σημαντικές είναι αυτές οι παρακολουθήσεις. Ακόμα και μετά από την 11η Σεπτεμβρίου θα ήταν αδιανόητο να υπάρχουν όλες αυτές οι δυνατότητες παρακολούθησης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε ότι όλα ε, η κίνηση στο διαδίκτυο, όλη η ροή δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων που εδρεύουν στις Ηνωμένε Πολιτείε, θα μπορούσε να είναι στοιχεία στα οποία έχει έχει πρόσβαση η NSA. Και ενώ είχα φτάσει στο σημείο να αντιλαμβάνομαι ποιος ήταν ο στόχος και να προετοιμαστώ και για τις ε, παρατηρήσεις που θα έκανα σήμερα στην παρέμβασή μου εδώ, το Σαββατοκυριακό οι New York Times μας έδωσαν ε, μία ακόμα πολύ συναρπαστική έρευνα, διότι σύμφωνα με τους New York Times η NSA μπορεί να αυξήσει τα στοιχεία τα οποία λαμβάνει με υλικό από διάφορες πηγές που περιλαμβάνει και τραπεζικούς λογαριασμούς, ε, προφίλ στο facebook, ε, ε, ε, ποιος εγγράφεται για να ψηφίσει στους εκλογικούς καταλόγους, καθώς επίσης και μία σειρά από φορολογικά στοιχεία βάσει των εγγράφων τα οποία δημοσιεύθηκαν αυτό το Σαββατοκύριακο. Αυτό σημαίνει ότι το να διαθέτει ένα τέτοιο προφίλ ε, ένας αμερικανικός οργανισμός παραβιάζουν την νομοθεσία περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής και πέραν της παρούσας έρευνας που γίνεται για την ε, ε, νομοθεσία για τις ξένες παρακολουθήσεις και τις μυστικές υπηρεσίες θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Βέβαια ξέρω ότι δεν σας έχω πει τίποτα το οποίο να διασκεδάζει τις ανησυχίες σας από όσο γνωρίζω. Και το θέμα είναι τι μπορούμε να πούμε για την παρακολούθηση από πλευρά Ηνωμένων Πολιτειών Ευρωπαίων πολιτών. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να σας πω καταρχάς δύο απλά πράγματα. Πραγματικά πιστεύω ότι όλες οι κυβερνήσεις είναι υποχρεωμένες να προστατεύουν τους πολίτες τους και να φροντίζουν να είναι ασφαλείς. Και επίσης θεωρώ ότι όλες οι κυβερνήσεις έχουν δικαίωμα να προσπαθήσουν να εντοπίσουν ποιες είναι οι απειλές κατά της χώρας τους. Για αυτά τα βασικά στοιχεία νομίζω ότι κανείς από εμά ε, δεν θα μπορούσε να διαφωνήσει. Το ερώτημα είναι πώς μια δημοκρατική κυβέρνηση κάνει διάκριση μεταξύ φίλων και εχθρών και συμμάχων και πραγματικών απειλών. Στην αρχική νομοθεσία για τις ε, παρακολουθήσεις στο εξωτερικό θεωρήθηκε ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στις πραγματικές απειλές στις Ηνωμένες Πολιτείες και όλα αυτά επί τη βάση της νομοθεσίας για να δημιουργήσουμε μία βάση για να ξεκινήσει η ηλεκτρονική παρακολούθηση. Σήμερα πλέον έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο ώστε έχουμε απομακρυνθεί τόσο πολύ από τη θεμελιώδη αρχή για την ηλεκτρονική παρακολούθηση, που φαίνεται ότι ακόμα και οι αρχές του δικαίου έχουν αναστραφεί τελείως. Η NSA ανα πάσα στιγμή καθοδηγείται από την επιθυμία της να αποκρύψει, να αποφύγει, να παρακάμψει, να παρερμηνεύσει και να αγνοήσει τις νομικές αρχές για να μπορέσει να επεκτείνει τις πρακτικές μέσω των οποίων συλλέγει στοιχεία. Όσοι ασχολούνται με την ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά δεδομένα και τις πολιτικές ελευθερίες, είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να ανησυχούν ε, για το θέμα αυτό. Τι μπορούμε να κάνουμε. Τρεις σύντομες συστάσεις. Οι κυβερνήσεις ε, επικοινωνούν για μία σειρά από θέματα. Οι κυβερνήσεις ε, συνεννοούνται για την προώθηση του εμπορίου και ε, προς όφελος των επιχειρήσεών τους και των καταναλωτών τους. Μιλώ όμως εξ ονόματος οργανώσεων καταναλωτών και στις Ηνωμένε Πολιτείες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σας προτείνω ότι καλό θα ήταν από ευρωπαϊκή σκοπιά τουλάχιστον να ανασταλούν οι εμπορικές διαπραγματεύσεις εν αναμονή της ε, απόφασης για τις ε, έρευνες ε, για τις παρακολουθήσεις. Διότι οποιοδήποτε άφιλος μπορεί να προκύψει από το περαιτέρω εμπόριο θα είναι εις βάρος του κάθε ανθρώπου όταν τα προσωπικά τους δεδομένα ταξιδεύουν σε διεθνή σύνορα. Κανείς δεν θα μπορεί να είναι σίγουρος ότι προστατεύεται η ιδιωτική του ζωή και ε, προστατεύεται όπως θα έπρεπε και στη χώρα τους. Δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να προχωρήσουν οι νέες εμπορικές συμφωνίες εάν δεν υπάρχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αντίστοιχα, θα ήθελα να σας προτείνω να επανεξετάσετε και το παρόν πλαίσιο για τη μεταφορά των στοιχείων PNR και των στοιχείων SWIFT, τα μητρώα των ε, επιβατών και τα τραπεζικά στοιχεία. Και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού θα πρέπει κανονικά να καθοριστεί ένα πλαίσιο το οποίο θα μας επιτρέψει να εντοπίσουμε ποιες είναι οι πραγματικές απειλές για την ασφάλεια και των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και της Ευρώπης. Και εδώ δεν ε, προτείνω να αλλάξει τίποτα. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι από την ευρωπαϊκή πλευρά όταν τα δεδομένα σας πηγαίνουν στις Ηνωμένε Πολιτείε, δεν είναι ασφαλή όπως θα ήταν εάν ε, ήσασταν ε, πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών βάσει της νομοθεσίας για την ιδιωτική ζωή. Για ιστερικούς λόγους, το 1974 όταν εγκρίθηκε η σχετική νομοθεσία, ελάχιστοι νομοθέτες είχαν θεωρήσει ότι θα έφτανε κάποια ημέρα που οι εθνικές υπηρεσίες θα συνέλεγαν ε, καθημερινά στοιχεία άλλων κυβερνήσεων. Και ίσως ε, γι' αυτό το λόγο ε, οι νομοθέτες της συγκεκριμένου, της συγκεκριμένου νομοθετήματος είχαν πολύ υψηλή προστασία για τους Αμερικάνους πολίτες αλλά έχουμε περάσει πολλά χρόνια από εκείνη την ημέρα και σήμερα πλέον στην Ευρώπη μας τα χρηματοοικονομικά σας δεδομένα, τα ταξιδιωτικά σας δεδομένα, ε, πληροφορίες οι οποίες είναι διαθέσιμες δημοσίως για οποιοδήποτε ε, στοιχείο θα μπορούσε να βρίσκεται σε ψηφιακή μορφή στο διαδίκτυο, μπορεί να διαβιβαστεί σε εθνικές υπηρεσίες πληροφοριών. Και ίσως για κάποιο λόγο θα μπορούσε κάποιος να συλλέξει αυτά τα δεδομένα, αλλά δεν ξέρω βάσει ποιας λογικής μπορεί κάποιος να πει ότι ναι, μπορείτε να συλλέξετε αυτά τα δεδομένα και δεν υπάρχουν και ταυτόχρονα δικλείδες ασφαλείας όπως αυτές που υπάρχουν στην νομοθεσία περί ιδιωτικής ζωής των ΗΠΑ. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς πυρηνικός επιστήμονας για να αντιληφθεί αυτό το επιχείρημα. Ε. Ε, θα πρέπει να υπάρχουν οι αρχές της αμοιβαιότητας, οι οποίες είναι σαφώς καθορισμένες στο διεθνές δίκαιο. Και αν οι Ηνωμένε Πολιτείε θέλουν να λαμβάνουν αυτά τα στοιχεία για τους Ευρωπαίους πολίτες, θα πρέπει να παρέχονται οι ίδιες δικλείδες ασφαλείας όπως παρέχονται και στους Αμερικανούς. Τέλος, να σας πω ότι είναι κατεπήγον να υπάρξει ένα διεθνές πλαίσιο για την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Γνωρίζω ότι πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο ανησυχεί ιδιαίτερα εσάς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γνωρίζω ότι πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο ε, ανησυχεί την Επίτροπο Ρέντινγκ και στο οποίο έχει αναφερθεί και η Επίτροπος και άλλοι. Υπάρξουν και κυβερνητικέ οργανώσεις οι οποίες προσέγγισαν τις ΗΠΑ που ζητούν να κυρώσει ε, να κυρώσουν οι ΗΠΑ τη συγκεκριμένη ε, σύμβαση για την ιδιωτική ζωή, διότι θεωρούμε ότι αυτό παρέχει τι κατάλληλε δικλείδες ασφαλεία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αλλά επίσης γνωρίζουμε ότι υπάρχει και ένα κίνημα το οποίο ε, είναι συνεχώς αυξανόμενο και θέλει να εξεταστούν τα πολιτικά και αστικά δικαιώματα, κυρίως το άρθρο 17, το οποίο αναφέρεται στην προστασία της ιδιωτικής ζωής. Ε, κάτι το οποίο έχει κυρώσει και, έχουν κυρώσει και οι Ηνωμένε Πολιτείες και πολλές άλλες χώρες και το ενέκριναν και οι Επίτροποι Προστασίας Δεδομένων στην συνεδρίασή τους στη Βαρσοβία. Ίσως λοιπόν με αυτό θα μπορούσα να ολοκληρώσω την παρέμβασή μου και θα μπορούσα να αποτελέσει και την αφετερία για το πώ θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα τη προστασία των προσωπικών δεδομένων στο σύγχρονο κόσμο. Στην ε, Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το 1948 των ΗΠΑ ε, αναφέρεται αυτό και θα ήθελα να σα το διαβάσω. Κανεί δεν θα πρέπει να υπόκειται σε αυθαίρετη ή παράνομη παρέμβαση τη ιδιωτική του ζωή, τη οικογένειά του, τη οικία του ή τη αλληλογραφέα του και ε, θα πρέπει να γίνονται σεβαστοί οι μνήμοι του καθενό. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να προστατεύεται κατά τέτοιων πράξεων και αυτά ε, θεωρώ ότι είναι το ίδιο επίκαιρα σήμερα όπως και τότε που εγγράφησαν το 1948 περιγράφουν πώς θα πρέπει κανονικά να λειτουργούν οι δημοκρατικές κυβερνήσεις οι οποίες θέλουν να προστατεύσουν την ιδιωτική ζωή των πολιτών τους. Ελπίζω αυτό να είναι κοινή μέρημνα για όλους, ε, για τις κυβερνήσεις από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι θα δώσουμε το λόγο τώρα στη δεύτερη ομιλήτρια. Thanks. I'm obviously new here. I appreciate the help. On behalf of the American... Ευχαριστώ εκ μέλου τη Ένωση για τι Πολιτικέ Ελευθερίε των ΗΠΑ. Ήθελα να σα ευχαριστήσω για την ευκαιρία να σα μιλήσω εδώ για τα θέματα τη ηλεκτρονική παρακολούθηση. Η ACIU είναι μια εθνική ένωση στι ΗΠΑ με πάνω από 4.000 μέλη που ασχολείται με τι αρχέ τη ελευθερία και τη ισότητα όπω διατυπώνονται στο Αμερικανικό Σύνταγμα και στους ομοσπονδιακούς μας νόμους. Καταλαβαίνω ότι σκοπό αυτή τη ακρόαση είναι να κοιτάξουμε πώς εξετάζονται οι κατηγορίες όπως παρουσιάζονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το τι γίνεται με την αναλογικότητα και την ε, νομιμότητα της παρακολούθησης των προσωπικών δεδομένων. Σήμερα θα ήθελα να επικεντρωθώ στο τι κάνει ακριβώς η δική μας ένωση αλλά και άλλες εθνικές μας ενώσεις στις ΗΠΑ. Ήθελα να περιγράψω το τι είδους προσπάθειες έχουμε καταβάλει ως τώρα προκειμένου να συνδυάσουμε τις ε, προσπάθειές μας. Ελπίζω ότι περιγράφοντας την, ε, το έργο τέτοιων ενώσεων θα μπορέσετε κι εσείς να σκεφτείτε καλύτερα πώς θα καθορίσετε την πορεία σας. Χάρη σε πολλούς από τους υπεύθυνου για να καταγράφουν τα δεδομένα μας, αυτή τη στιγμή έχουμε την ε, μεγάλη εμβέλεια παρακολούθηση δεδομένων όπως έπρεπε να έχει γίνει από καιρό στις ΗΠΑ. Η εθνική μας υπηρεσία έχει κάποιες φορές παρακολούθηση τηλεφωνικών συνομιλιών, ηλεκτρονικών ε, επικοινωνιών, όχι μόνο στις ΗΠΑ αλλά και ανά τον ε, κόσμο. Στο άρθρο 215 του Patriot Act καθορίζεται ότι μπορούν όλα τα μεταδεδομένα τηλεφωνικών επικοινωνιών να καταγράφονται εκτός και εντός πολιτεών. Στον αναθεωρημένο νόμο 702 του 2008 λέγεται ότι όλες οι τηλεφωνικές επικοινωνίες ανά τον κόσμο μπορούν να παρακολουθούνται προκειμένου να συγκεντρώνονται τα απαραίτητα στοιχεία. Αυτά είναι προγράμματα που έχουν συζητηθεί εντατικά αλλά και άλλα υπάρχουν. Με το πρόγραμμα Χένες, ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε βελτίωσε την πρόσβαση, ε, κάμπτοντας τα εντάλματα, χωρίς δικαστική δηλαδή έγκριση, και μπορεί να καταγράψει τηλεφωνικά στοιχεία από το 1997. Το πρόγραμμα αυτό φαίνεται ότι στόχο έχει τις εγχώριες βέβαια εξελίξεις και έρευνες, όμως και η Ευρώπη με τα εθνικά της προγράμματα δεν θα περιοριστεί σε θέματα μόνο εθνικής παρακολούθησης. Ε, η Ένωση λοιπόν σκοπό είχε να παρακολουθήσει τους ε, στη χώρα, τραπεζικά συστήματα, ε, ηλεκτρονικές ανταλλαγές, email, chat στο ίντερνετ, τηλεφωνήματα και βεβαίως οι ερευνητές θεώρησαν ότι εφόσον η Ένωση μας μπορεί να έχει καλύτερη πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να φτάσει πιο εύκολα και σε εξωτερικούς ε, εχθρούς ή σε ενδιαφερόμενες εταιρείες. Το περιεχόμενο των ε, επικοινωνιών στο διαδίκτυο τώρα είναι ένα συγκεκριμένο θέμα, διότι ως τώρα είχαμε κράσει ανησυχίε για, την, ε, για τον αναθεωρητικό νόμο 702, και τα όσα προβλέπει για τα προγράμματα upstream και την παρακολούθησή τους. Παραμένουν ερωτήματα για, την, για το πεδίο ακριβώς ε, του προγράμματος αυτού. Και οι ιδιώτες, οι πολίτες ανά τον κόσμο, δεν πρέπει να ξεχνάνε ότι καλό είναι να μην περνάνε οι κυβερνήσεις τους σε εντατική συγκέντρωση δεδομένων, σε μαζική συγκέντρωση δεδομένων που να τους αφορούν γιατί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολλαπλούς σκοπούς. Η Αμερικανική κυβέρνηση θεώρησε ότι οι Αμερικανοί δεν θα πρέπει να ανησυχούν με τη συλλογή δεδομένων. Το επιχείρημα όμως αυτό δεν είναι ακριβώς σωστό. Πρώτον, διότι δεν είμαστε αφελείς για τις διάφορες μυστικές υπηρεσίες ανά τον κόσμο, όποιου κράτους και αν είναι, και για τους σκοπούς τους. Η παρακολούθηση και από άλλες κυβερνήσεις αφορά ε, ξένους πληθυσμούς εκτός από τον Αμερικανικό. Και υπάρχουν χώρε όπου δεν υπάρχει νόμο που να απαγορεύει την παρακολούθηση των ε, επικοινωνιών των πολιτών. Αυτό δεν σημαίνει όμω ότι μια κυβέρνηση θα πρέπει να το πραγματοποιεί αυτό. Υπάρχουν πρακτικέ που ελπίζουμε να καταγγελθούν από του πολίτε ε, στι διάφορε χώρε όπου λαμβάνουν χώρα. Οι μόνιμε αντιπροσωπείε των ΗΠΑ ε, καταγράφουν χώρε όπου στοιχεία για του Αμερικανού καταγράφονται όντω και παρακολουθούνται. Αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει να σκεφτούμε και τι γίνεται με τους αλλοδαπούς που είναι στόχος του εξωτερικού. Η ΕΠΙΚ υπέβαλε μήνυση για αυτήν ακριβώς τη διάταξη και την υλοποίησή της. Στη μήνυση αυτή η Amnesty International, κατά κλάπερ δηλαδή, δημιουργήθηκε μια μεγάλη ομάδα δικηγόρων, ακτιβιστών, εκπροσώπων των δημοσιογράφων, των ε, πολιτών όπου η έρευνα αυτή αφορούσε και συναδέλφους εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, ανθρώπους που ήταν θύματα εγκλημάτων μίσους, συναδέλφους πολλές φορές. Η Amnesty International, η Human Rights Watch και η Ένωση που υπερασπίζεται, οι Ενώσεις που τους πολίτες σε διάφορες χώρες συμμετείχαν στην όλη προσπάθεια, όμως το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ την ε, απέρριψε. Δεν ήταν αρκετά τεκμηριωμένο το επιχείρημα ότι παρακολουθούνται οι τηλεπικοινωνίες. Δεν μπορεί να μην διερωτάται κανός, κανείς σήμερα πώς τέτοια θέματα που είχαν ανακύψει από το παρελθόν ε, θα μπορούσαν να είχαν λάβει διαφορετική τροπή εάν ίσχυαν τα σημερινά νομοθετικά δεδομένα. Τώρα, για το πρόγραμμα μαζικών καταγραφών τηλεπικοινωνιών. Το πρόγραμμα αυτό το αποκάλυψε στις στις 5 Ιουνίου η Guardian λέγοντας ότι κάθε τηλεφωνική συνομιλία εντός και εκτός των ΗΠΑ καταγράφονται από, την εθνική μυστική, από τις εθνικές μυστικές υπηρεσίες σε καθημερινή βάση. Όπως πολλοί σημείωσαν, το πρόγραμμα αυτό ως προς το πεδίο του είναι πραγματικά τεράστιες εμβέλειες. Αλλά μπορεί πραγματικά ο κάθε Αμερικανός να, ξε, είναι βέβαιος ότι ακόμα και ο κατάλογος με τις ε, επαφές του είναι γνωστός στις μυστικές υπηρεσίες. Μιλάμε για πραγματικά συλλογική καταγραφή δεδομένων από όλες τις μεγάλες τηλεφωνικές εταιρείες και τουλάχιστον για μια επταετία πίσω. Η Ένωσή μας λοιπόν ξαφνιάστηκε με το θέμα αυτό της Guardian και την υπόθεση της Horizon, διότι και εμείς είμαστε πελάτες της Horizon. Οπότε, μια εβδομάδα μετά την δημοσίευση του άρθρου, εμείς μηνύσαμε στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο και ε, η μήνυση αυτή στράφηκε κατά του προγράμματος που παραβιάζει και το πρώτο νόμο για το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου και το τέταρτο για την απαγόρευση της παρέμβασης της κυβέρνησης στη ζωή των πολιτών. Το τέταρτο άρθρο του Συντάγματος των ΗΠΑ προστατεύει τους πολίτες. Ο πρόεδρος Ομπάμα και άλλα μέλη της κυβέρνησης δυσκολεύτηκαν και έρθαν ε, σε δύσκολη θέση και αναγκάστηκαν να τονίζουν ότι το πρόγραμμα αυτό καταγράφεται με τα δεδομένα των τηλεφωνικών επικοινωνιών και όχι όλο το περιεχόμενο. Όμω το τέταρτο άρθρο θεωρεί την τοποθέτηση αυτή, κάνει μάλλον την τοποθέτηση αυτή ανεφινοήματος. Πώς καθορίζει κανείς ποιο είναι το περιεχόμενο και ποια τα μεταδεδομένα. Εφόσον όλα τα τηλεφωνήματα αποκαλύπτονται ακόμη και αν ας πούμε κάποιος τηλεφωνεί σε μια κόκκινη γραμμή, γραμμή επιγόντων για την ε, οικογενειακή βία μια, ένα απλό τηλεφώνημα, μπορεί να είναι γνωστό. Αυτό θα έπρεπε να απορρίπτεται ακόμα και βάσει του πρώτου άρθρου, διότι καταπατάτε η ελευθερία του λόγου και του... και του συνασπίζεστε. Εδώ λοιπόν η Ένωση καταγράφει και γνωρίζεται ότι τα τηλεφώνηματα τους καταγράφονται από τους whistleblowers σε καθημερινή βάση αλλά εδώ οι υπηρεσίες μπορούν να καθορίσουν μια συμπεριφορά ως ε, παράνομη ή όχι αυθαίρετα. Συζητήσαμε λοιπόν το θέμα αυτό για να επηρεάσουμε και μέλη του Κογκρέσου και να μπορέσουμε και με τη συνεργασία άλλων ενώσεων να επικαλεστούμε το τμήμα 317 όπου βάση της διάταξης αυτής είναι σαφές ότι οι στόχοι της καταγραφής ήταν ε, να χρησιμοποιηθούν στον αγώνα κατά της θερμοκρατίας. Ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκλησή σας και πραγματικά ανυπομονώ να ακούσω τις ερωτήσεις σας. Okay, thank you very much. Ευχαριστώ και στους δύο ομιλητές. τον πρώτο γύρο των ερωτήσεων και φυσικά θα ζητήσω κατόπιν από τους δύο μιλητές να απαντήσουν. Αν έχουμε αρκετό χρόνο μπορούμε να κάνουμε και ένα δεύτερο γύρο ερωτήσεων και απαντήσεων. Αλλά παρακαλώ να είστε σύντομοι, συγκεκριμένοι, έτσι ώστε να μπορέσουν όλοι να πάρουν το λόγο. Ο εισηγητής όμως έχει το λόγο πρώτος. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και τους δύο μιλητές. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές ερωτήσεις, γι' αυτό και είμαι πολύ σύντομος. Στον Μάρκ Ρότενμπεργκ θα ήθελα να πω ότι πραγματικά ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η ομιλία σας. Ιδιαίτερα όταν γίνεται αναφορά στο άρθρο 17, και στις ε, πολιτικές ελευθερίες. Νομίζω πραγματικά ότι το θέμα της προστασίας είναι πολύ σημαντικό, όπως ε, είπες. Η ερώτησή μου λοιπόν καταρχήν είναι τι θα κάνει αυτή τη βδομάδα το Κογκρέσο όσον αφορά τη νομοθεσία, πώς έχει προχωρήσει η πρόταση και θα θέλαμε να ξέρουμε τι ε, προστασία πρόκειται να μας παρέχει από εδώ και πέρα η νομοθεσία των ΗΠΑ και τι πρέπει να κάνουμε εμείς μόνοι μας για να προστατευτούμε. Αναφέρθηκε στις εμπορικέ συμφωνίες και στα δεδομένα SWIFT, τα τραπεζικά δεδομένα αλλά και τα δεδομένα των επιβατών Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω ποια είναι η κατεύθυνση, ποιος είναι ο προσανατολισμός του Αμερικανού νομοθέτη προς αυτή την κατεύθυνση, τι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Αυτή η ερώτηση απευθύνεται και στην κυρία Κραμπ. Δεν ξέρω τι έχετε να μας πείτε όσον αφορά αυτό το θέμα. Πρόεδρος να γίνουν πρώτα οι ερωτήσεις και μετά να απαντήσετε. Ωραία. Οι σκιώδεις εισηγητές. Για το ΕΛΚ πρώτα. Ναι, και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους δύο ομιλητές. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους δύο μιλητές. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι παρουσιάσεις τους. Από αμερικανικής απόψεως πήραμε πολλές πληροφορίες. Έχω λοιπόν ερωτήσεις, ιδιαίτερα ακούγοντας τον κύριο Ρότενμπερ και τις συστάσεις του. Με ακούτε? Ναι. Με ακούτε? Όσον αφορά τις συστάσεις ε, του κυρίου Ρότενμπεργκ, θα ήθελα να σας πω ότι όσον αφορά την συμφωνία την εμπορική, τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη συμφωνία για να θέσουμε ένα επίπεδο ασφάλειας όσον αφορά τα δεδομένα. Μπορούμε δηλαδή να συμπεριλάβουμε στις διαπραγματεύσεις μας και τα προσωπικά δεδομένα και την προστασία τους. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο, έχω την εντύπωση ότι εδώ πρόκειται για δύο διαφορετικές διαδικασίες. Από τη μία είναι η νόμιμη οδός και από την άλλη η μη νόμιμη οδός κατά κάποιο τρόπο μέσω της NSA. Το θέμα είναι να κοιτάξουμε το νόμιμο κομμάτι, τι μπορούμε να κάνουμε μέσα σε μια συμφωνία ή ε, δημόσια αν θέλετε ή να δούμε πώς μπορούμε να καταργηθεί το παράνομο κομμάτι. Γιατί αν θέλουμε να προστατευτούν τα δεδομένα εμείς σαν Ευρωπαίοι, είτε θα προσεγγίσουμε το θέμα από τη δική μας πλευρά, είτε θα πούμε ότι είτε πρόκειται για ευρωπαϊκό επίπεδο προστασίας, είτε για αμερικανικό, είτε για κινέζικο, είτε για ρώσικο, θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το επίπεδο προστασίας στην κάθε χώρα, στην κάθε ήπειρο και να προσπαθήσουμε να βρούμε κάποια διεθνή ε, δεδομένα προστασίας, αν αυτά υπάρχουν. Πρόεδρος, είμαι εισηγήτρια για την Άλντε, αλλά θα μιλήσω τελευταία. Εξ ονόματος των Πρασίνων Άλμπρεχτ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ μαζί μας. Και ε, οι προτάσεις σας είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Θα σας ρωτήσω λοιπόν το εξής. Τι έχετε να πείτε για τις περιπτώσεις παρακολουθήσεων που γίνονται εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή από την NSA αλλά σε ε, άλλες χώρες και με βάση τρίτες χώρες. Δηλαδή δεν πρόκειται για παρακολουθήσεις οι οποίες εμπίπτουν στον νόμο, στην νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχουν τόσες πολλές υπηρεσίες που βεβαίως εδρεύουν στην ε, Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε αυτή την περίπτωση έχουμε πρόβλημα εμείς ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Υπάρχει λοιπόν από τη μία η συζήτηση που λαμβάνει η χώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και των ε, ελευθεριών των πολιτών των Ηνωμένων Πολιτειών και από την άλλη υπάρχει η παρακολούθηση εκτός από τρίτες χώρες. Μιλάμε λοιπόν εδώ για διπλά στάνταρτ και φυσικά ε, κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει η Αμερικανική κυβέρνηση να συνειδητοποιήσει ότι και για τους μη Αμερικανούς πολίτες θα πρέπει κάτι να γίνει ε, όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα και όσον αφορά το Privacy Act και την ενδεχόμενη μεταρρύθμιση του. Θα ήθελα επίσης να μου πείτε πώς βλέπετε το θέμα της διαφάνειας, της πρόσβασης από μέρους ε, και άλλων αρχών, άλλων κυβερνήσεων Υπάρχει, όπως ξέρετε, και ένα αίτημα των Ηνωμένων Εθνών για περισσότερη διαφάνεια και πρόσβαση και βεβαίως σήμερα θα ήθελα να ξέρω αν υπάρχουν κινήματα για περισσότερη διαφάνεια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, ε, από τη στιγμή που θα διαπιστωθεί ότι υπάρχει παραβίαση ε, ποιος μπορεί να προσφύγει. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχει κανείς από μέρος της ΕΣΥΑΡ, αλλά θα δώσω το λόγο αμέσως στην ΓΚΟΕ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν σας ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ. Είναι μια πολύ ζωντανή συζήτηση. Είναι πολύ ενδιαφέρον για μας που μπορούμε να έχουμε τέτοιες ε, ανταλλαγές απόψεων και σε μια τέτοια περίπτωση που μας ε, φαινόταν ε, χωρίς δυνατότητες διαλόγου είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον που μπορούμε να έχουμε τέτοιους συνομιλητές σαν και εσάς. Θα ήθελα να μου πείτε λοιπόν τι είναι αυτό που εμποδίζει περισσότερο την αλλαγή, το να προχωρήσουμε και να αλλάξουμε κάτι σε αυτή την κατάσταση. Και δεν εννοώ μόνο νομοθετικά, αλλά ουσιαστικά τι πρέπει να κάνουμε, πού βλέπετε να υπάρχουν τα σημαντικότερα εμπόδια. Γιατί όπως ξέρετε μπορεί να αλλάξει ο νόμος πολλές φορές, το πρόβλημα όμως να παραμένει. Και εδώ μιλάμε πολύ για ένα διεθνές πλαίσιο, για διεθνή πρότυπα. Η ερώτησή μου όμως είναι πώς θα αρχίσουμε να σεβόμαστε οι μεν τους δε, να διαπιστώσουμε που υπάρχουν πραγματικές ανάγκες. Κάτι πρέπει να γίνει ως προς την ουσία κατά την άποψή μου. Επίσης, όσον αφορά την Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου. Είπατε ότι είναι σημαντικό να γίνει κάτι στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας. Αλλά πείτε μας πολύ συγκεκριμένα θα χρησιμοποιήσουμε αυτήν την συμφωνία για να προστατεύσουμε ικανοποιητικά τα προσωπικά δεδομένα. Πείτε μας ακριβώς τι εννοείτε. Τρίτη ερώτηση. Από τη στιγμή που υπάρχει παρακολούθηση και Αμερικάνων πολιτών, πείτε μου ποια είναι εδώ η νομική βάση και πώς αντιδρούν οι πολίτες Υπάρχουν κινήματα στην Αμερική όπως σε εμά εδώ στην Ευρώπη που αντιδρούν. Υπάρχουν απομονωμένες, μεμονωμένες αντιδράσεις, υπάρχουν μαζικές αντιδράσεις. Ε, εδώ δεν αναφέρομαι στους Ευρωπαίους, αναφέρομαι στους Αμερικανούς πολίτες. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Και τώρα θα θέσω κι εγώ κάποιες ερωτήσεις εξ ονόματος των φιλελευθέρων. Πολύ σύντομα, διότι είναι πολλές ερωτήσει που θέλω να θέσω. Καταρχά. ποια είναι η άποψή σα για την αποτελεσματικότητα τη ε, βόρεια ως ε, αντίβαρο σε αυτές τι παρακολουθήσει. Εγώ πραγματικά θεωρώ ότι είναι πολύ πιο αποτελεσματική από τον ε, κανονισμό για τη διαφάνεια που έχουμε εμεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν όρια. Όλα αυτά τα προγράμματα μαζικών παρακολουθήσεων πάντα αιτιολογούνται για, με την ανάγκη για ασφάλεια. Όλοι θέλουμε ασφάλεια, ε, όπως είπαν και άλλοι, αλλά τι αποδείξεις υπάρχουν ότι πραγματικά είμαστε ασφαλείς. Υπάρχουν ενδείξεις για αποτελέσματα. Ε, υπάρχει τρόπος μέσω των ε, μηχανισμών ελέγχου, να ελέγξουμε ότι όντως είμαστε ασφαλείς. Και το αντίθετο, υπάρχουν αποδείξεις ότι τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για σκοπούς που δεν έχουν καμία σχέση με την ασφάλεια. Μα δίνεται εντύπωση ότι χρησιμοποιούνται όντως για άλλους σκοπούς. δεν υπάρχουν άλλα νομικά μέσα. Νομίζω ότι ο Μάρκ Ρότεμπερκ ε, αναφέρθηκε ε, λίγο σε αυτό. Υπάρχουν και άλλες δυνατότητες νομικής συνδρομής. Γιατί δεν ζητούν πληροφορίες οι Αμερικανοί από εμά αντί να ε, απλώνουν τα πλοκάμια τους στις βάσεις δεδομένων μας. Ε, αναφερθήκατε στους συμμάχους σας και πάντα με εντυπωσιάζουν αυτά που κάνουν οι οργανώσεις της ε, κοινωνίας των πολιτών και για την προστασία της πολιτικής ελευθερίας στις ΗΠΑ. Ποιοι είναι οι εταίροι σας, με ποιους συνομιλείτε, ε, και θεωρώ ότι είναι κατεπίγουσα η ανάγκη να έχουμε και έναν αντίστοιχο ευρωπαϊκό οργανισμό. Συνεργάζεστε με ευρωπαϊκούς οργανισμούς, είναι χρήσιμο και τι συμμάχους έχετε σε άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα τη Βραζιλία, η οποία καθόλου δεν ικανοποιήθηκε από το γεγονός ότι παρακολουθούσαν τον πρόεδρό τους για τις τηλεφωνικές τους συνδιαλέξεις στις ΗΠΑ. Θα ήθελα λοιπόν να απαντήσετε στις ερωτήσεις οι οποίες ετέθησαν και θα κάνουμε και ένα γύρο ε, υπαριθμών 2, διότι έχουμε άλλα πέντε άτομα που ζήτησαν το λόγο. Καταρχάς όμως να απαντήσετε σε ερωτήσει. Ο Μάρκ πρώτα. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Κύριε τα κάνατε κάποιες ερωτήσεις και είναι πολύ σημαντικό να σας πω ότι ναι, βεβαίως η Αμερικανική κυβέρνηση σήμερα δεν έχει μια ενιαία θέση και άποψη, αλλά όσον αφορά την συλλογή δεδομένων υπάρχει μια μεγάλη συμφωνία όλων των πολιτικών τάσεων ότι θα πρέπει αυτό το πρόγραμμα PRISM να σταματήσει και μάλιστα έγινε μια ψηφοφορία όσον αφορά δηλαδή και τους Ρεπουμπλικάνους και τους Δημοκράτες υποστήριξαν ε, τον πολύ σημαντικό περιορισμό αυτών των δραστηριοτήτων και μάλιστα για πέντε ψήφους δεν πέρασε η πρόταση να σταματήσει τελείως η χρηματοδότηση του προγράμματος για την NSA όσον αφορά την συλλογή ε, δεδομένων και πληροφοριών. Αυτές οι αλλαγές που έχουν σημαντικές επιπτώσεις όσον αφορά την παρακολούθηση στην Ευρώπη ε, θα πρέπει να εντοπίσετε αυτές που πραγματικά θα έχουν αποτελέσματα. Σε αυτό πρέπει εσείς στην Ευρώπη να είστε πολύ προσεκτικοί, να μην γίνουν κάποιες αλλαγές οι οποίες δεν θα έχουν επιπτώσεις. Γιατί ουσιαστικά αυτά που αποφασίζονται στι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν επιπτώσεις και δεν επηρεάσουν καθόλου τη δραστηριότητα των Αμερικανικών υπηρεσιών εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό λοιπόν είναι ενδιαφέρον για σας και αυτό θα πρέπει να εστιάσετε. Γι' αυτό και σας μίλησα για τις εκρεμείς εμπορικές συζητήσεις για την Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου. Και έχω την εντύπωση ότι αν κάνετε κάποια αιτήματα με σκοπό και να προστατευθούν τα προσωπικά δεδομένα αλλά και να προχωρήσει και να υπογραφεί η Συμφωνία Εμπορικών Συναλλαγών μπορείτε να ζητήσετε από τις Ηνωμένε Πολιτείες να ε, δημιουργηθούν, να καθοριστούν ασφαλιστικές δικλίδες προστασίας για τους Ευρωπαίους πολίτες. Τίποτα άλλο. Είναι πολύ απλό και με αυτόν τον τρόπο θα θεσπιστούν και θα δημιουργηθούν νομικές εγγυήσεις έτσι ώστε να υπάρξει πραγματική προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί κανείς να σας το αρνηθεί, πρέπει όμως οπωσδήποτε να το ζητήσετε και έχω την εντύπωση ότι και ο κύριος Όλμπρεκτ και όλοι οι συνάδελφοι μπορούν να κάνουν προτάσεις προς αυτήν την κατεύθυνση. Εμείς έχουμε ένα πολύ ωραίο πλαίσιο στις Ηνωμένε Πολιτείε όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αυτό έχει ανακοινωθεί και είναι γνωστό και έχει δημοσιευθεί πριν από ένα χρόνο. Από εκεί και πέρα και έχω την εντύπωση ότι αν υπάρξει και μεγαλύτερη πίεση μπορεί να αυξηθεί ακόμα περισσότερο το επίπεδο προστασίας όπως έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη και έτσι να επωφεληθούν οι Ευρωπαίοι πολίτες από αυτή την προστασία. Είπατε επίσης ότι θα θέλατε να ξέρετε ποια είναι τα νομικά εμπόδια. Κοιτάξτε, αν υπάρχει μία συμφωνία η οποία υπάρχει και ισχύει, θα πρέπει να είσαστε σε θέση να διαπιστώσετε αν και στην ουσία, στην πράξη, αυτά που έχετε συμφωνήσει και υπογράψει εμφαρμόζονται. Επαναλαμβάνω ότι το πρώτο βήμα θα ήταν η υπογραφή μιας συμφωνίας, δεύτερον όμως να δείτε αν στην πράξη υλοποιούνται αυτά. Κύριε Όλμπρεχτ, είπατε επίσης ότι θα θέλατε να ξέρετε ποιοι είναι οι σωστοί μηχανισμοί για την προστασία των δεδομένων. Έχω την εντύπωση ότι το πρώτο και το πιο σημαντικό είναι να ξέρει κάποιος ποια είναι τα δεδομένα που τον αφορούν τα οποία κατέχει μια υπηρεσία. Εγώ λοιπόν νομίζω ότι μπορείτε να κάνετε το ερώτημα τι πληροφορίες έχετε για μένα, για το πρόσωπό μου, πού τις βρήκατε, πού τις φυλάτε και για ποιο σκοπό τις έχετε συλλάξει και πώς μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε. Και πολύ ε, φοβάμαι ότι και οι ιδιωτικές και οι δημόσιες ε, επιχειρήσεις που ε, έχουν συλλέξει τέτοια δεδομένα που σας αφορούν θα αρνηθούν να απαντήσουν με διαφάνεια. Οι συγκεκριμένες λοιπόν συστάσεις που μπορώ να σας δώσω είναι ότι πραγματικά στην Αμερική το Privacy Act οδήγησε σε μια πραγματική αλλαγή της κατάστασης. Το διεθνές πλαίσιο για την προστασία της προσωπικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων άλλαξε πραγματικά τα πράγματα. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι η συνέχεια είναι κάτι που θα ενδυναμώσει το επίπεδο προστασίας στις Ηνωμένε Πολιτείες, στις συναντήσεις που είχαμε με τους συμβούλους του Προέδρου, με τον Πρόεδρο, από τη στιγμή που προετοιμάσαμε και μία γνωμοδότηση νομική, έχουμε συναντήσει όλες τις νομικές υπηρεσίες και αυτό θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό. Θα χρησιμοποιήσουμε επίσης όλα αυτά τα δεδομένα έτσι ώστε ένας ε, όμπουτσμαν ένα συνήγορος του πολίτη να μπορέσει να αναλάβει αυτό το θέμα και να εγείρει όλες τις περιπτώσεις αυτές κατά της Αμερικανικής κυβέρνησης. Θεωρούμε ότι όλα αυτά, χωρίς να αλλάξουν βεβαίως την κατάσταση στην Ευρώπη όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων Ευρωπαίων πολιτών, σίγουρα είναι ευίωνα στοιχεία εάν εσείς θελήσετε να αναλάβετε δράση για την προστασία των πολιτών στην Ευρώπη. Όσον αφορά όλα αυτά είμαι σίγουρος ότι η πίεση που προέρχεται από τις αποκαλύψεις του κυρίου Σνόντεν σίγουρα ε, θα οδηγήσει την Αμερικανική κυβέρνηση σε μια περαιτέρω αλλαγή της τάσης της και της συμπεριφοράς της. Ευχαριστώ πολύ. Ε, αστείο να λέτε ότι κάποιος θα λέει στο, ε, στις οργανώσεις ε, τι στοιχεία έχουν. Όταν ρώτησα εγώ, σε καμία περίπτωση δεν ήταν διατεθειμένοι να μου πούνε, ακόμα και μετά από μια δημοσιογραφική υπόθεση. Κυρία Κράμπ, ευχαριστώ. Θα προσθέσω να μην επαναλάβω τα όσα είπε ο κύριος Ρότεμπερκ, θα προσθέσω κι εγώ ένα-δυο σχόλια. Μία ερώτηση ήταν τι θα γίνει αν και άλλες χώρες ε, έκαναν ε, στην NSA ό,τι κάνει ε, η NSA στην Google και στη Yahoo. Οι αποκαλύψεις του Snowden στην πραγματικότητα μας έδειξαν αυτό που ε, φαίνεται ότι είναι μεγάλο σφάλμα. Δεν θα πρέπει να εξαρτώμαστε τόσο πολύ από το διαδίκτυο μιας άλλης χώρας. Και αυτό ε, σημαίνει ότι φοβούνται ότι θα αλλάξουν τα πράγματα και θα μειωθούν οι δυνατότητες που έχουν. Αυτά τα κινήματα για τη διαφάνεια καλά μεν, αλλά νομίζω ότι όλα αυτά θα γίνουν κατόπιν εορτής και δεν θα υπάρχει κανένα ε, ε, νόημα. Δείτε για παράδειγμα το άνταλμα για τη Verizon. Η Verizon ε, αν δείτε πόσα εντάλματα έχουν συλλεχθεί είναι 12 ή 6, αλλά αν αυτό το μετρήσετε με τον αριθμό των ατόμων ε, τα οποία παρακολουθήθηκαν, έχουμε εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους. Και το άλλο το οποίο με κάνει αποφαλεκτικό για αυτή την έκθεση για τη διαφάνεια είναι Πού ήταν κρυμμένοι όλοι αυτοί τόσα χρόνια. Κάποιε από τους παρόχους ε, διαδικτυακών υπηρεσιών, η ε, Yahoo, η Google, δεν ήταν καλύτερες από τις ε, τηλεπικοινωνιών. Εγώ εδώ και χρόνια προσπαθούσα να πείσω τις τηλεφωνικές επιχειρήσεις να απαντήσουν στα βασικά ερώτημα του πόσο καιρό αποθηκεύονται τα δεδομένα των πελατών. Πόσο καιρό, για παράδειγμα, αποθηκεύονται τα μηνύματα τα οποία στέλνονται μέσω κινητού τηλεφώνου. Επίσης, τα αρχεία του ποιου ποιος τηλεφώνησε και σε ποιον τηλεφώνησαν. Και τελικώς σε μία μικρή πόλη στο Χίκερινό ε, στην Βόρεια Καρολίνα δόθηκαν ε, ε, στοιχεία μέσω ενός εγγράφου που σε μία σελίδα μας εξηγούσαν για πόσο ακριβώς καιρό αποθηκεύονται τα στοιχεία αυτά από τις επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών. Δεν ήταν τόσο δύσκολο τελικώς να συντάξει κάποιος σε μια σελίδα, αλλά εδώ και χρόνια δεν το έλεγαν στους Αμερικανούς και χαίρομαι ιδιαίτερα διότι ε, γίνεται με ε, κάποια κίνηση προς τη διαφάνεια πλέον, αλλά νομίζω ότι το κίνητρο είναι μάλλον ε, η ανησυχία για τα επιχειρηματικά συμφέροντα και το γεγονό ότι ο κόσμος στο εξωτερικό κυρίω πιστεύει ότι παραβιάζεται τα προσωπικά του δεδομένα και όχι από κάποια ανάγκη για πραγματική διαφάνεια. Ε, για το Foiler, ναι, θα μπορούσε να είναι και χρήσιμο εργαλείο αλλά και χρήσιμο παιχνίδι. Νομίζω ότι αυτό το οποίο απέδειξε είναι ότι υπάρχει μεγάλη ανεπάρκεια και ε, ε, αν μάθαμε κάτι από τον Έντουαρτ ε, Snowden τους τελευταίους τρεις μήνες είναι ότι άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε τις παρακολουθήσεις που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όλοι ζήτησαν πληροφορίες για τις αρχές οι οποίες είναι αρμόδιες ε, για τα θέματα αυτά και τελικά χρειάστηκε ένας να μας δώσει πληροφορίες, ένας whistleblower για να μας παρουσιάσει όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία ζητούσαμε τόσα χρόνια. Και για να συνεχίσω και από κάτι που ανέφερε ο κύριος Ρότεμπεργκ, συμφωνώ απολύτως ότι μάλλον είναι απίθανο ε, οποιαδήποτε από τις ε, ε, οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών που, προστατεύει τα πολιτικά, που ασχολείται με την προστασία των πολιτικών ελευθεριών στην ΗΠΑ θα πετύχει κάτι. Δεν έχουμε αρκετά εργαλεία διότι το Αμερικανικό Δίκαιο κυρίως προστατεύει τους Αμερικανούς πολίτες και θα πρέπει να ασχοληθούμε με αυτά που έχουμε και επομένω δεν έχουμε πολλά πράγματα στη διάθεσή μας για την προστασία των αλλοδαπών. Ευχαριστώ. Φτάνουμε με αυτό στο δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Έχουμε πέντε άτομα που έχουν ζητήσει το λόγο. Θα ήθελα να σας ζητήσω όταν θα απαντήσετε στο δεύτερο γύρο ερωτήσεων να επανέλθετε και λίγο σε αυτό που ανέφερα εγώ για τις αποδείξεις για αποτελέσματα ή για κατάχρηση των δεδομένων. Η κυρία Μορβάη και οι υπόλοιποι που άκουσαν το όνομά τους είναι στον κατάλογο. Θέλει κάποιος άλλος το λόγο. Αν όχι, η κυρία Μορβάη έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω την ερώτησή μου καθότι θεωρώ ότι εδώ υπάρχει μία, μη, ένας μη ανταγωνισμός. Βλέπουμε από τη μία τις Ηνωμένες Πολιτείες να παραβιάζουν τα δικαιώματα των πολιτών της Ευρώπης. Παραδείγματος χάρη ε, στην ε, Ουγγαρία. Ο κύριος Σοταβάρες ο ίδιος, ο οποίος δεν είναι σήμερα εδώ, ενώ είναι μεγάλος υπερασπιστής ε, των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ε, ελευθεριών. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη έλλειψη ενδιαφέροντος, ενώ αυτές οι περιπτώσεις είναι καθαρά παραβιάσεις της νομιμότητας, πρόκειται για παραβιάσεις και παράνομες πράξεις από μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών. Μου θυμίζει εδώ το 1984 του Orwell. Γιατί υπάρχουν αυτές οι υπηρεσίες οι οποίες συγκεντρώνουν αδιάκριτα πληροφορίες ηλεκτρονικές για την ιδιωτική ζωή των Ευρωπαίων. Παρακολουθούνται ε, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, μας λένε ότι αυτές δεν έχουν ενδιαφέρον άμεσο, ενώ ξέρουμε ότι αυτό βεβαίως ε, είναι ψέμα. Γνωρίζουμε σήμερα ότι για να παρακολουθήσουν τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις του, της Προέδρου της Βραζιλίας ή του Μεξικό, αυτό δεν μπορεί να έχει σαν σκοπό να προστατεύσουν τους πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τρομοκρατικών επιθέσεων. Ποιος είναι λοιπόν ο σκοπός, για ποιο λόγο συλλέγουν αυτές τις πληροφορίες και αυτά τα δεδομένα και τι θα τα κάνουν. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί μη κυβερνητικοί οργανισμοί οι οποίοι θέλουν να αντιδράσουν και να βοηθήσουν να προστατεύσουν τον κύριο Σνόντεν. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι ποιος και πώς θα προστατευθεί ο κύριος Σνόντεν στις Ηνωμένε Πολιτείες. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σίβολ για δύο λεπτά. Η κυρία πολύ συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομη. Άκουσα ότι στις Ηνωμένε Πολιτείες υπάρχει σήμερα μία πολύ σημαντική συζήτηση όσον αφορά αυτήν την συλλογή δεδομένων. Βεβαίω, σήμερα είναι πολύ αργά μετά από αυτό που συνέβη στις 11, την 11η Σεπτεμβρίου και τουλάχιστον θα πρέπει να δούμε ότι στην Αμερική μετά από τις πρόσφατες αποκαλύψεις έχουν γίνει κάποιες ε, βελτιώσεις όσον αφορά την νομοθεσία ή την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τουλάχιστον στην Αμερική. Αυτό που μας λέτε λοιπόν είναι ότι όντως έγιναν βελτιώσεις ή απλώς γίνονται κάποιες ανακοινώσεις καθησυχαστικές για να σταματήσει η συζήτηση που έχει ξεκινήσει. Επίσης πείτε μας κάτι παραπάνω πώς ε, θα πρέπει να μεθοδευτεί αυτή η συζήτηση μεταξύ Ευρωπαίων και Αμερικανών. Συμφωνώ με τον Μάρκ Ρότενμπεργκ ότι αν χρησιμοποιήσουμε εδώ τις εμπορικές διαπραγματεύσεις μπορούμε να πετύχουμε κάτι στις Ηνωμένε Πολιτείες μπορεί να σταματήσει η παρακολούθηση των Αμερικανών πολιτών, αλλά όλοι αδιαφορούν στις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά την συνέχιση των παρακολουθήσεων Ευρωπαίων πολιτών. Συμφωνώ λοιπόν με τον κύριο Ρόδενμπερκ ότι κάτι πρέπει να κάνουμε με την Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου, γιατί με αυτόν τον τρόπο πιέζουμε όχι μόνο τις Ηνωμένε Πολιτείες, αλλά και τις Ευρωπαϊκές Αρχές να κάνουν κάτι. Θα πρέπει λοιπόν ίσως να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας και πείτε μας πώς μεταξύ Ευρωπαίων, Αμερικανών και μη κυβερνητικών οργανισμών. Πώς αποσπά η NSA τις σωστές πληροφορίες από αυτήν την τεράστια βάση δεδομένων. Δεν θέλω να υποβεβάσω το έργο σας, αλλά υπάρχει κατάλογος προσώπων ή οργανισμών που σας ενδιαφέρουν περισσότερο Πώς εντοπίζετε τους ανθρώπους που εμπλέκονται σε όλα αυτά και σε ποιο βαθμό οι Αμερικανοί ε, ζημιώνονται από τέτοιου είδους μη πολιτικές ε, επαφές από τις ενέργειες της NSA. Πώς χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες επίσης, τις καταγράφετε ως πληροφορίες ή μπορεί να αναλυφθεί και νομική δράση. Επίσης, η συζήτηση αυτή πώς γίνεται, πώς οργανώνεται στις ΗΠΑ, ποιος πιέζει για να προχωρήσει η παρακολούθηση, ποιον τα συμφέροντα και ποιον οι ομάδες πίεσης ε, παρεμβαίνουν στον ιδιωτικό βίο των πολιτών. Υπάρχουν ε, διασυνδέσεις με άλλα τρίτα κράτη και μεταφέρονται ποτέ τα δεδομένα αυτά σε ξένες χώρες. Ακούσαμε κάτι πολύ ενδιαφέρον την περασμένη εβδομάδα. Ο κύριο Ομπάμα είπε ότι το πρόβλημα της παρακολούθησης δεν είναι μόνο η, κακή χρήση, αλλά ότι η ίδια η επίγνωση ότι κάποιος παρακολουθείται μπορεί να οδηγήσει σε ακτιβισμό ή κάποιοι να αναπτύξουν δράσεις σε ιστότοπου χωρίς να ήταν αρχικά ο σκοπό του. Εάν λοιπόν, σωστά το αντιλαμβάνομαι, οι μυστικέ υπηρεσίε δεν θεωρούν ότι δεσμεύονται από του νόμου περί ιδιωτικού βίου, όπω εμεί οι κοινήθνητοι. Η συνέπεια είναι ότι όποια νομοθεσία και αν εγκριθεί, τελικά δεν θα περιορίζονται. Και μια τελευταία παρατήρηση, και επειδή εδώ υπάρχει μεγάλη προσέλευση, νομίζω η προσέλευση θα ήταν μεγαλύτερη εάν μπορούσαμε την ε, συνεδρίαση της Πέμπτης και τη σημερινή να τις είχαμε συνδυάσει στην ίδια μέρα. Πρόεδρος, δυστυχώς δεν είμαι εγώ υπεύθυνη γι' αυτά. Δεν νομίζω όμως ότι επαναλήψαν οι συνεδριάσεις. Ευχαριστώ. Να σας ευχαριστήσω για τις α, πολύ πλούσιες Παρουσιάσει σας και τις πληροφορίες που μας δώσατε. Αναφερθήκατε στις διάφορες συνομιλίες ε, μεταξύ οργανώσεων προστασίας των ε, ελευθεριών και αρχών των Ηνωμένων Πολιτειών και των πιθανών επιπτώσεων για την Ευρώπη. Εγώ πιστεύω ότι η συνεργασία μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής πρέπει να συσφιχθεί, πρέπει να γίνει εντενότερη και καταρχήν στο επίπεδο των ε, βουλευτών αυτό πρέπει να το κάνουμε εμείς. Πείστε μας τι άλλο πρέπει κατά την άποψή σας να κάνουμε, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε και ενδεχομένως να αυξήσουμε τη συνεργασία σε κάποια επίπεδα που να υπάρξει αποτέλεσμα θετικό για την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Λάτφορντ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήθελα να ευχαριστήσω και την Κάθριν και τον Έντμα για, την, για τις παρουσιάσεις τους. Έχουμε λάβει μεγάλη βοήθεια από την ΕΠΗ και την και αυτός είναι και βασικός λόγος που Δεν θέλουμε να αποκόψουμε την Ευρώπη από τις Ηνωμένε Πολιτείε. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά κοινά ενδιαφέροντα και συμφέροντα. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι η Ευρώπη έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά το τι συμβαίνει γενικότερα σε επίπεδο κράτους, ενό μεγάλου κράτου όπως οι Ηνωμένε Πολιτείε και γενικά με την παρακολούθηση. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να πιέσουμε με τρόπο ευθύ και τις κυβερνήσεις και την, ε, τις εταιρείες. Δεν είναι μόνο η NSA το θέμα. Το τελευταίο τρίμηνο, αν θυμηθούμε τι έγινε, είναι και η Βρετανική DCHQ και οι Γάλλοι το ίδιο, να μην είμαστε βεποκριτές. Οπότε υπάρχει πρόβλημα και εντός Ευρώπης ένα θέμα υπερβολικής παρακολούθησης από τις μυστικές υπηρεσίες. Είναι δύσκολο να χειριστούμε την όλη διαδικασία. Πώς θα ασκηθεί πίεση με σωστό τρόπο χωρίς να βάλουμε τρικλοποδιά στον εαυτό μας. Νομίζω ότι η αναστολή ε, των εμπορικών διαπραγματεύσεων είναι μάλλον... Ε, ε, θα έχει μάλλον το αντίθετο αποτέλεσμα. Ο σκοπός εδώ είναι να έρθουμε πιο κοντά και να βρούμε έξυπνους τρόπους προστατεύοντα και τον ε, επιχειρηματικό αυτό κλάδο και τα εμπορικά του συμφέροντα, βρίσκοντα λύσει που ε, να συμπεριλαμβάνουν και το να απιστή το Κογκρέσο. Πολλοί ε, συνάδελφοι, μεταξύ των οποίων και εγώ, είχαν εμπειρία και πείρα. Εγώ υπήρξα πρόεδρος της Επιτροπής για τις μυστικές υπηρεσίες και τις πληροφορίες της γερουσίας και εδώ θα πρέπει να συνδυάσουμε τις δυνάμεις μας, αλλιώς δεν βλέπω να βρίσκεται λύση. Είπατε ότι το Κογκρέσο θα απαιτήσει νομικές διασφαλίσεις και για τους Ευρωπαίους. Αυτό πώς θα εξυπηρετήσει όμως του Αμερικανού ε, στα πλαίσια του NSA. Ο νόμος για τον ιδιωτικό βίο δεν έχει βοηθήσει για, το, για την ώρα του ίδιου του Αμερικανού. Πρόεδρος, αυτές ήταν οι ερωτήσεις. Ίσως να απαντήσουμε αντίστροφα και να απαντήσει πρώτα η κυρία Κράμπ. So Πολλές ερωτήσεις. Θα τις ε, πιάσω από τα μαλλιά και θα αρχίσω να απαντάω στην κύκη. Έγινε ερώτηση για τον Σνόντεν. Και αν υπάρχουν προετοιμασίες για την υπόθεσή του. Τι κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά. Έχουμε ήδη δηλώσει ότι είμαστε ευγνώμονες για τη δική του συνεισφορά στην εκπόνηση των προγραμμάτων μας και εφόσον χρειαστεί υπεράσπιση θα την έχει εάν φτάσει στις ΗΠΑ. Ακούστηκε και μια σειρά από ερωτήσεις για το πώς αποσπώμε τα σωστά δεδομένα μεταξύ των όλων πληροφοριών που έχουμε. Υπάρχουν κάποια προγράμματα που συμπεριλαμβάνουν την μαζική συλλογή, την ευρεία συλλογή δεδομένων, αδιακρίτως. Κάποια όμως κάνουν επιλακτική συλλογή δεδομένων, αναχώρα, αναπεριφέρεια. Είναι δύσκολο να σας δώσω μια συνολική απάντηση εδώ. Πάντως, με τις επερχόμενες αποκαλύψεις του κυρίου Σνόντεν, και επειδή το συζητούν όλο και περισσότερο στην κυβέρνηση, πιστεύουμε ότι σύντομα θα έχουμε τις κατάλληλες, περισσότερες και ευστοχότερες πληροφορίες. Τώρα, ο νόμος για την παρακολούθηση είναι και η βάση της νομικής μας αυτής προσφυγής κατά της κυβέρνησης. Δηλαδή, Υπάρχουν πολίτες που θέλουν να συζητήσουν με οργανώσεις όπως η CLU αν, αν θεωρήσουν ότι οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περάσουν και στα χέρια της κυβέρνησης. Αλλά από την ιδιότητά μου ε, στην νέα μιλώ με πολύ κόσμο. Ουδέποτε στο παρελθόν ε, είχα συνομιλίες με τόσους δημοσιογράφους που να λένε πόσο φοβούνται. Πόσο φοβούνται μήπως καταγραφούν οι απόψεις τους για θέματα όπως το NSA. Οι αποκαλύψη του Σνόντεν κατέστησαν σαφές ότι κάποιοι δημοσιογράφοι είχαν ε, παρακολούθηση στις ηλεκτρονικές τους επαφές. Και θεωρούσαν ότι η εμπλοκή τους σε τέτοια προγράμματα μπορεί να οδηγούσε και σε περισσότερη παρακολούθηση της ζωής τους. Κάποιοι δημοσιογράφοι μόνο είχαν πρόσβαση σε συγκεκριμένα έγγραφα και βρέθηκαν ε, απομονωμένοι, χωρίς θεσμική υποστήριξη. Οπότε πώς να κάνουν τη δουλειά τους. Για τα αποδεικτικά στοιχεία της παραβίασης ε, έγινε μια ερώτηση, αλλά και αυτό είναι κάτι που οι αρχές το καθορίζουν. Εμείς εκτός ε, κυβέρνησης δεν έχουμε στοιχεία για το πώς χρησιμοποιήθηκαν τελικά τα δεδομένα και πληροφορίες η κυβέρνηση. Κάποιες φορές δίνει θεωρητικά υποθετικά στοιχεία και δίνει έμφαση σε κάποια δεδομένα αποκρύπτοντας ε, κάποια που έχουν σχέση με τρομοκρατικές οργανώσεις. Οι απαντήσεις είναι κάπως ασαφείς. Στις Ηνωμένε Πολιτείε ε, είμαστε εξαρτημένοι από κάποια μέλη του Κογκρέσου, ιδίω η Ένωση μας, που οι άνθρωποι αυτοί έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες λόγω της, δημο... της κρατικής του λειτουργήματο. Αλλά υπάρχουν και πολλά ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων. Για το κατά πόσο βελτιώνουν την ασφάλεια και κατά πόσο ε, σέβονται την ε, αρχή της αναλογικότητας κατά τη συλλογή των τηλεφωνικών μεταδεδομένων όπως ονειμάστηκαν και πώς αυτό διακρίνεται από τα ουσιαστικά στοιχεία. Thank Ευχαριστώ. Για τον ε, κύριο Σνόντεν, νομίζω ότι με κάλεψε η συνάδελφος και φίλη και που είναι στο επόμενο πάνελ και θα διαβάσει ε, ε μία δήλωση για το Snowden ε, η Τζέσλιν Ράντακ, επομένως νομίζω ότι καλύπτω από τη δική της την απάντηση. Ρωτήθηκε ε, αυτή η κρίσιμη ερώτηση γιατί να συλλέγονται δεδομένα, για ποιο λόγο συλλέγονται αυτά τα δεδομένα. Να σας πω την άποψή μου. Τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται δημοσίως αποτελούν δημόσια γνώση, συνεισφέρουν προς αυτόν και αυτό είναι εξαιρετικό. Στοιχεία τα οποία συλλέγονται απορρίτως χρησιμοποιούνται για να αποκτήσει κάποιο μεγαλύτερη εξουσία και έλεγχο. Και αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο οι σύγχρονε δημοκρατικέ κυβερνήσει ανησυχούν ιδιαίτερα για αυτή τη μυστική συλλογή πληροφοριών. Διότι το θέμα είναι η εξουσία και ο έλεγχο. Η κυρία Σίπχολ ρώτησε γιατί αλλάζουν τα πράγματα στις ΗΠΑ Πολιτείες και νομίζω ότι τμήμα των απαντήσεων είναι ότι γίνεται ένας γενικευμένος δημόσιος διάλογος, αλλά επίσης ο Λευκός Οίκος ε, συνομιλεί με ηγέτες εδώ στην Ευρώπη και εκφράζεται μεγάλη ανησυχία μεταξύ των κυβερνήσεων για τις συνέπειες της παρακολούθησης των τηλεπικοινωνιών, διπλωματών, ε, εμπορικών ε, εταίρων ε, και άλλων ε, δημοσίων αξιωματούχων. Νομίζω ότι υπάρχει ένα όριο πέρα από το οποίο ε, αυτοί που βρίσκονται στα υψηλά οφήκια θεωρούν ότι δεν θα πρέπει να υπερβούμε. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι η απάντησή σας. Τέθηκε και μία σειρά από υπεροπτικές ερωτήσεις από τον κύριο Εμπρόνς για το τι ακριβώς κάνει η NSA. Προσπαθούμε όλοι να μάθουμε η δική μου οργάνωση ε, έχει αρκετές πηγές, ε, η ε, ACLU έχει επίσης πολλά στοιχεία, ο οργανισμός της CRAMP και η δική μας η EPIC και προσπαθούμε όλοι μαζί να αποκτήσουμε μια καλύτερη εικόνα. Για μένα, μεταξύ των πιο αποκαλυπτικών εγγράφων δεν ήταν μόνο τα εντάλματα τα οποία αποστάλησαν και ζητούσαν τις πληροφορίες, αλλά και οι δικαστικές αποφάσεις οι οποίες ε, εκδίδονται τώρα από τα δικαστήρια, οι οποίες περιλαμβάνουν πάρα πολλές λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησαν αυτά τα προγράμματα και σύμφωνα με τα δικαστήρια ε, διαπιστώθηκαν και πολλές παραβιάσεις και του συντάγματος ε, και του συνταγματικού δικαίου και νομοθεσίας εν γέννη και αυτά τα εξετάζουμε. Ρωτήθηκε επίσης πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς στις Ηνωμένε Πολιτείε τις διεθνείς ανησυχίε. Νομίζω ότι το κοινό στις Ηνωμένε δεν λαμβάνει υπόψη του ακόμα την παγκόσμια διάσταση των παρακολουθήσεων το NSA. Ο, η πρόεδρος της Βραζιλίας ε, αποφάσισε να μην συναντηθεί με τον πρόεδρο Ομπάμα για το θέμα αυτό ε, και είναι και θέμα σε εκλογέ σε άλλες χώρες αλλά νομίζω ότι ε, ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο σημείο το, στο οποίο ανησυχεί τους Αμερικανούς. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί ε, με τις διάφορες πολιτικές μάχες που δίνονται. Κάποιες φορές οι πολιτικοί δεν θέλουν να εκχωρήσουν κάποια άλλα τους δικαιώματα, τα οποία είναι πολύτιμα και αυτό το αντιλαμβάνομαι. Ε, οι αμερικανογερμανικές ε, σχέσεις είχαν και το θέμα αυτό της παραβίασης των προσωπικών δεδομένων και στην επιστολή μου ε, υπήρχε κάτι το οποίο άρεσε σε διαφόρους. Οι φίλοι δεν κατασκοπεύουν φίλους. Υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά μεταξύ της έρευνας για ε, κατασκόπους και ανθρώπους που αποτελούν απειλή για τη χώρα σου και ε, συστηματική συλλογή στοιχείων για συμμάχους, φίλους και συναδέλφους. Και νομίζω ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν περάσει αυτή τη διαχωριστική γραμμή. Σας ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να κατασκοπεύουμε μόνο ε, πιθανές απειλές εναντίον μιας χώρας. Νομίζω ότι ε, δεν νομίζω ότι θα προχωρήσει πολύ αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ για την συνεισφορά σας. Είμαι βέβαιη ότι η Επιτροπή μας θα μείνει σε επαφή μαζί σας και μπορεί να σας θέσουμε και κάποιες περαιτέρω ερωτήσεις οι οποίες μπορεί να προκύψουν στα πλαίσια των ερευνών μας. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τους δύο πάρα πολύ. Πριν περάσουμε στην επόμενη σειρά ομιλητών, θα ήθελα να πω το εξή. Έχουμε προσκαλέσει και τις Αμερικανικές Αρχές για να μας δώσουν στοιχεία, αλλά αρνήθηκαν. Λάβαμε κάποιες επιστολές, οι οποίες θα έλεγαν και σας παραθέτω εδώ. Λυπούμαστε, αλλά δεν μπορούμε να ενθαρρύνουμε επίσημη ε, συμμετοχή από πλευράς ΗΠΑ και να σας πω ότι στην προηγούμενη ε, ακρόαση είχαμε καλέσει τις Ολλανδικές αρχές οι οποίες αρνήθηκαν, είχα, έχουμε καλέσει και τις Βρετανικές αρχές για κάποια συνεδρίαση στο μέλλον και ακόμα περιμένουμε να, αποφασί, να απαντήσουν. Εάν κάποιος λοιπόν θέλει να επικρίνει τη σύνθεση και την ισορροπία εδώ στις ακροάσεις θα πρέπει να γνωρίζει ότι έχουμε καλέσει όλες τις πλευρές για να μας προσκομίσουν στοιχεία αλλά κάποιοι αρνήθηκαν. Κύριε Μορβάη έχετε κάτι διαδικαστικό. Ναι, θα ήθελα να ζητήσω τα αντίγραφα αυτών των επιστολών. Καλό θα ήταν να τα έχουμε όλοι, γιατί θα μπορούσαμε ίσω να τα δώσουμε και στι περιφερειέ μα στη συνέχεια. Είμαι βέβαιη ότι μπορούν να σας τα στείλει αυτά η γραμματεία. Δεν νομίζω να είναι απόρριτα. Και άλλωστε οποιοδήποτε απόρριτο στοιχείο δεν είναι πλέον μυστικό, είναι κοινό μυστικό γνωστό τη πάση. Ευχαριστώ. Να περάσουμε λοιπόν στον επόμενο γύρο μιλητών, να καλέσω εδώ στο πάνελ τους ομιλητές. Στο επόμενο τμήμα έχουμε τους whistleblowers, τις δραστηριότητες τους, αφενός και την ε, νομική προστασία αφετέρου, διότι όπως ακούστηκε και εδώ ε, από τους πρώτους ομιλητές, ο ρόλος τους είναι ζωτικός, διότι το επίπεδο διαφέανες που διαθέτουμε δεν ε, λειτουργεί αποτελεσματικά. Θα ακούσουμε λοιπόν τρεις μαρτυρίες. Πρώτα απ' όλα ο κύριος Ντρέγκ, ο οποίος είναι πρώην εργαζόμενος της NSA, μετά με τηλεδιάσκεψη την μαρτυρία του κυρίου Βίμπε, ο οποίος είναι και εκείνος αναλυτής της NSA. Θα μιλήσει μαζί μας μέσω τηλεδιάσκεψης από την Washington και μετά την κυρία Άννη Μάκεν. Ελπίζω ότι προφέρω σωστά το όνομά της. Ήταν ε, εργαζόμενη MF5. Sorry. I was instructed wrong. <laughs> I tried to get it right, sorry. Okay, we're going to uh, ask each of you to, uh, to do a 15-minute presentation. Θα έχουμε μια 15 λεπτή παρουσίαση, αλλά λόγω της τηλεδιάσκεψης θα σας ζητήσω να παραμείνετε εντός του χρόνου ομιλίας σας, γιατί θα έχουμε τεχνικά προβλήματα διαφορετικά. Καλώ ήρθατε στην Επιτροπή μα. Θα ζητήσω τον κύριο Τέικ να ξεκινήσει. Έχετε το λόγο για 15 λεπτά. Ευχαριστώ το Ευρωκοινοβούλιο και την Επιτροπή σα, που με καλέσατε να μιλήσω για αυτό το κρίσιμο θέμα σε αυτή την ακρόαση. Μιλάμε για τα προγράμματα των εθνικών ε, μυστικών υπηρεσιών και το τι γίνεται στι διάφορε χώρε σε σχέση με τον ιδιωτικό βίο ε, των πολιτών και στη δική μου χώρα και στη δική σα. Ε, Πολλές φορές οι κυβερνήσεις εμπλέκονται και με άλλες ξένες κυβερνήσεις, με τη ζωή των πολιτών σε άλλες χώρες, με κατασκοπία, με τις τηλεφωνικές υπηρεσίες και τηλεφωνικούς πάροχους άλλων χωρών και βεβαίως υπάρχει κάποιες φορές δυσκολία ή και διευκόλυνση παρακολούθησης της ζωής των πολιτών στην καθημερινή ζωή. Με συγχωρείτε να σας διακόψω για ένα δευτερόλεπτο. Οι διερμενείς θα σας ζητήσουν να Μιλήστε λίγο πιο αργά γιατί δεν μπορώ να σας παρακολουθήσω. Ήμουν ένας ε, ειδικό αποκρυπτογράφησης ε, και τα τελευταία χρόνια του ψυχρού πολέμου ε, είδαμε σε ευρωπαϊκά θέατρα να χρησιμοποιούνται ειδικοί κώδικες για να μπορέσουν να περάσουν μηνύματα από την Ανατολική Γερμανία. Οι κατάσκοποι έχουν συνηθίσει να μαθαίνουν τα πάντα. Αυτό είναι το μοντέλο που χρησιμοποιείται. Όμως ποτέ δεν φαντάζομαι ότι θα μπορούσαν ε, οι Αμερικανοί να χρησιμοποιήσουν εκείνο το εγχειρίδιο των κατασκόπων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου για να παρακολουθούν τη ζωή των πολιτών της χώρας τους και άλλων εκατομμυρίων εκτός ε, Αμερικής. Θέλουμε εμείς να είμαστε αντικείμενα ή υποκείμενα της παρακολούθησης των μυστικών υπηρεσιών, όλοι γίνονται καχύποπτοι, αλλά ο νόμος προστατεύει και τον ιδιωτικό βίο και την ελευθερία της έκφρασης. Οπότε, υπό το πρόσχημα ότι πρέπει να είμαστε όλοι ασφαλείς, ε, κάποιες φορές υπάρχει πουλή παρακολούθηση και συλλογή δεδομένων, με τεράστιο όγκο που αφορούν την καθημερινή μας ζωή. Το καθεστώς αυτό παρακολούθησης έχει γίνει ένα παγκόσμιο φαινόμενο, ένα σύστημα με πολλά πλοκάμια που έχει ξεπεράσει τα όρια της καταπολέμησης της θερμοκρατίας και των υπόλοιπων διακρατικών και διεθνών εγκληματικών ενεργειών. Η Επιτροπή σας πρέπει να κοιτάξει τι ακριβώς συμβαίνει με τις σκιές στο σύστημα της παρακολούθησης και της συλλογής δεδομένων, πώς παραβιάζονται τα δικαιώματα των πολιτών και πώς κάποιοι ε, καταλύουν περιοχές εθνικής κυριαρχίας με το σύστημα αυτό. Έτσι διαρριγνύονται σχέσεις εμπιστοσύνη μεταξύ εθνών και διακινδυνεύονται οι διπλωματικές μας σχέσεις και σε εμπορικά και οικονομικά ζητήματα. Ε, δεν μπορεί να χρησιμοποιείται η ασφάλεια ενός κράτους ως πρόσχημα για να περιέβαζονται ζωές πολιτών άλλων χωρών. Πολλές φορές οι απειλές λαμβάνουν υπερβολικές διαστάσεις και υπάρχει πρόσβαση στα δεδομένα του καθενός μας σε όλα τα επίπεδα χωρίς αυτό να αιτιολογείται. Υπάρχουν τεχνολογικά μέσα και πρωτόκολλα που επιτρέπουν σε πολίτες αλλά και ιδιωτικές εταιρείες οι ιδιώτες να αναπτύσσουν σχέσεις εμπιστοσύνης με τη θεωρία ότι τα δεδομένα τους και η ζωή τους προστατεύεται. Όταν αυτό όμως γίνεται αντικείμενο εμπορικό είναι δύσκολο να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη. Τίποτε δεν είναι τόσο σημαντικό όσο η κυριαρχία και η προστασία των πολιτών μας όταν δημιουργείται ένα τέτοιο τεράστιο σύστημα παρακολούθησης. Από τις τελευταίες αποκαλύψεις φάνηκε ότι σε βιομηχανικό πια επίπεδο, σε τεράστια ε, κλίμακα, η Αμερικανική κυβέρνηση παραβίασε τα συνταγματικά δικαιώματα των πολιτών παραβιάζοντας την ακαιρεότητα και τα θεμελιώδη ε, δικαιώματα επίσης ε, πολιτών εκτός Αμερικής. Το γνωρίζω γιατί ήμουν της μάρτυρας στην ε, δημιουργία του κράτους αυτού υπερβολικής παρακολούθησης ε, μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001. Ήμουν εκεί από τη γέννηση του συστήματος. Ήταν ένας ε, όταν δούλευα στα κρατικά ε, στις κρατικές υπηρεσίες και έβλεπα πως υπήρχε τεράστια και ανεμπόδιστη πρόσβαση σε ψηφιακά στοιχεία με οικονομικές συναλλαγές, email, τηλεφωνικές επικοινωνίες. Οι Ηνωμένε Πολιτείε για σκοπούς παρακολούθησης και άντλησης δεδομένων έγινε ένα κράτος ε, που παραβίαζε ε, την, ε, δικαιώματα των πολιτών και Οι πολίτες έχουν βρεθεί όμοιροι της κυβέρνησης, καθώς χρησιμοποιούνται τα στοιχεία τους, περίπου όπως γινόταν τη δεκαετία του 60 και του 70 τα μυστικά αυτά προγράμματα παρακολούθησης. Δημιουργήθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες γύρω από την ημερομηνία της 11 Σεπτεμβρίου μετά αποφάσεις των ανώτατων κλιμακίων της Αμερικανικής κυβέρνησης. Τέτοιες παρακαμπτήριοι και αδιέξοδα δεν χρειάζεται να υπήρχαν, διότι εναλλακτικέ νόμιμες ε, θα βρίσκονταν. Μπορούσε να παρακολουθηθεί ε, να παρακολουθούνται τα απαραίτητα δεδομένα χωρίς να παραβιάζεται το ιδιωτικό ε, βίος των πολιτών ταυτόχρονα. Εδώ λοιπόν πρέπει να πω ότι είναι πολύ σοβαρές οι ανησυχίες μας, το έχω θέσει σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παγκοσμίω και γι' αυτό ακριβώς Έγινα δότης για δύο έρευνες που οργανώθηκαν κατόπιν της 11 η Σεπτεμβρίου λόγω της υπέρμετρης και ανεξέλεγκτης καταγραφής και κατακράτησης δεδομένων από τις Εθνικές Μυστικές Υπηρεσίες των ΗΠΑ. Εδώ μιλάμε για πρόγραμμα συλλογής δεδομένων αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2005 που ήταν πολύ περισσότερο ενοχλητικό παρά χρήσιμο στην ε, τελική του έκβαση δεν χρησιμοποιήθηκαν οι νόμιμες εναλλακτικέ. Ακολούθησα όλους τους κανόνες που ίσχυσαν για τους ε, πληροφοριοδότες, ορκιζόμενος να υπερασπίζουμε πρώτα απ' όλα τα όσα ορίζει το Σύνταγμα. Και αυτήν την υποχρέωση την ανέφερα, την ανανέωσα το 2006, προκειμένου να εφαρμόσω όσα ορίζει το πρώτο άρθρο του Συντάγματος για την ελευθερία της έκφρασης και την μη παραβίαση της ε, ε, ιδιωτικής σφαίρας, με αντισυνταγματικές πρακτικές. Όμως, αντί να διορθωθούν αυτές οι παρανομίες, ε, ε, έγινα στόχος. Στόχος μιας τεράστιας ομοσπονδιακής έρευνας για πληροφοριοδότες, επειδή έδωσα πολλά στοιχεία, αποκάλυψα ε, το μυστικό αυτό πρόγραμμα μαζικής καταγραφής και έχασα κάθε δυνατότητα ε, κρατικής σταδιοδρομίας. Μπήκα σε μαύρο κατάλογο ενώ ταυτόχρονα ε, έπρεπε να καταβάλω τεράστια δικατικά, να καλύψω τις δικαστικές δαπάνες. Έχασα το σπίτι μου, μου ε, καταργήθηκαν οι τραπεζικοί μου λογαριασμοί και βεβαίως όλες μου οι οικονομίες και τα συνταξιδετικά μου. Αυτό ήταν μόνο η αρχή έτσι κι αλλιώς. Αυτό που έζησα ως πληροφοριοδότης είναι τελικά δίνει ένα μήνυμα πολύ ανατριχιαστικό. Η κυβέρνηση όταν αποφασίσει να κάνει κάτι θα το κάνει. Όταν ε, θέλει να ασκήσει την εξουσία της. Εδώ μιλάμε για νομικά αντίπεινα και για λογοκρισία. Ε, τα αντισυνταγματικές παρακαμπτήρια που χρησιμοποιήθηκαν μπορούν να δικαιολογηθούν από ασαφή και ατεκμηρίωτα στοιχεία για την εθνική ασφάλεια και την προάσπιση της. Αυτά χρησιμοποιεί η κυβέρνηση ως επιχειρήματα. Όμως ζούμε σε μια εποχή όπου ανταλλάσσουμε πληροφορίες που είναι σημαντικές για το δημόσιο συμφέρον, αλλά δεν υπονομεύουν απαραίτητα την εθνική ασφάλεια και κάποιες φορές θεωρούνται ποινικά κολάσιμες, ενώ καταγγέλνουν το αντίθετο οι δημοσιογράφοι και ο τύπος. Δεν είναι αυτό μια ανοιχτή δημοκρατική και ανοιχτό μια κοινωνία. Έκανα ό,τι μπορούσα. Έκανα ό,τι μπορούσα για να προασπιστώ τα αναλύωτα δικαιώματα των Αμερικανών πολιτών και την, ε, την, την κυριαρχία μάλλον του ατόμου. Η κυβέρνηση δεν είχε κανένα λόγο να κάνει όσα έκανε και αυτό δεν σταμάτησα να το φωνάζω. Ήταν απλώς ε, ένας τρόπος για να πάει στην αντίπερα όχθη, την λεγόμενη ανε, ανευθυνότητα, παράνομα, μονομερός, αυθαίρετα και υπογείως. Έτσι λοιπόν άρχισα να δίνω πληροφορίες διότι θεώρησα ότι η αδικία ήταν πραγματικά σοβαρή εντός και εκτός μυστικών υπηρεσιών της χώρας μας. Δέχτηκα σωματική, μάλλον ήμουν θύμα σωματικής παρακολούθησης και ηλεκτρονικής από το FBI ε, από το 2007 και δυόμιση χρόνια μετά κατηγορήθηκα για ομοσπονδιακά αδικήματα με ενδεχόμενο φυλάξης 35 ετών. Οι τεράστιες κατηγορίες τις οποίες, ε, των οποίων έπεσα θύμα από το Υπουργείο Δικαιοσύνη της ε, χώρας είναι ουσιαστικά το αποτέλεσμα ε, της 11 Σεπτεμβρίου 2001. Αυτό χρησιμοποιήθηκε ως πρόσχημα με παραβίαση του δικαιώματο ελευθερία τη έκφραση και τη ιδιωτική σφαίρα. Η κυβέρνηση βρήκε ό,τι μπορούσε ω στοιχείο εναντίον μου και έγινε εχθρό του κράτου. Έγινα ο πρώτο ε, whistleblower που διώχθηκε ποινικά ε, μετά από τον δρακόντιο, το δρακόντιο αυτό καθεστώ που ίσχυσε από την 11η Σεπτεμβρίου και μετά. Οι πληροφοριδότε να ονομάζονται, να μην θεωρούνται πια κατάσκοποι. Και τα στοιχεία που συλλέγονται είναι αντικείμενο επεξεργασία τελείω αφαίρετη, χωρί καμία συγκατάθεση των πολιτών για του οποίου έχουν συλλεγεί. Η παρακολούθηση της χώρας μας ε, για τη ζωή των πολιτών χωρίς καμία διαφάνεια ενώ οι ειδικοί φωνάζουν για το αντίθετο, είναι κάτι που πρέπει να απασχολήσει όλους τους πολίτες. Θα πρέπει να ανησυχούν πολύ για το μέλλον τους, ε, για το τι γίνεται όταν οι ελευθερίε του παραβιάζονται πλήρω στο όνομα τη εθνική ασφάλεια, χωρί όμω τη συγκατάθεσή του. Ο φόβο που προκαλεί η επίκληση απειλών που μπορεί να είναι και φανταστικέ δημιουργεί ένα κλίμα φόβου ε, και ουσιαστικά καταλήγει αιμονή το θέμα τη εθνική ασφάλεια. Και προσπαθεί φυσικά η κυβέρνηση να ελέγξει τη ζωή των πολιτών. Η δική μου δικαστική υπόθεση είναι κάτι που ξέφυγε από κάθε έλεγχο λόγω των πιέσεων της κυβέρνησης. Παραβιάζει κάθε νόμο του συντάγματος και ξεφεύγει και από τα όρια της χώρας. Οποιαδήποτε μορφή κυβέρνησης λαμβάνει τη μορφή ενός κράτους που παρακολουθεί σε ακραίο βαθμό τους πολίτες του, παίρνει τελείω άλλη μορφή και αυτό αναθεματίζει και εξωστρακίζει κάθε μορφή δημοκρατίας. Καμία τυραννίδα δεν είναι πιο σκληρή από αυτήν που κινείται στα παρασκήνια του νόμου και στα υπόγεια της δικαιοσύνης. Μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι η κυβέρνηση επέλεξε να κάνει εμένα και κάποιους άλλους στόχους της, ώστε να δημιουργήσει μια συνολικότερη εκστρατεία κατά των whistleblowers. Και η κυβέρνηση βεβαίως μπορεί να ισχυριστεί ό,τι θέλει κατά των συγκεκριμένων ατόμων ή πολιτών. Έχει λάβει τέτοιες διαστάσεις αυτή, αυτό το φαινόμενο που πρόσφατα φάνηκε και από την υπόθεση του κυρίου Σνόντεν τα προγράμματα μαζικής παρακολούθησης των ΗΠΑ σήμερα είναι από τα μεγαλύτερα που έχουν υπάρξει ποτέ και αποτελούν απειλή για τον οποιονδήποτε στον πλανήτη. Χωρίς προστασία και νόμιμη κάλυψη οι πολίτες δεν είναι ασφαλείς. Η NSA κάνει αυτό που επιδιώκει ανεξέλεγκτα, ανεμπόδιστα, μυστικά και χωρίς ε, κανέναν έλεγχο. Εάν όλες οι πληροφορίες περνάνε στα χέρια των μυστικών υπηρεσιών, καταλαβαίνουμε πόσο υπονομεύεται έτσι η καρδιά του δημοκρατικού καθεστώτος, εντός του οποίου υποτίθεται ότι πρέπει να λειτουργεί η κυβέρνηση. Όλοι οι άνθρωποι ουσιαστικά γίνονται κτήμα της κυβέρνησης, όπως συνέβαινε πάντοτε στην ιστορία σε παρόμοιες καταστάσεις. Ε, και το πρόσχημα ότι αυτά μπορεί να χρησιμεύσουν στο μέλλον ως στοιχεία δεν είναι αρκετό. Το βαρύ χέρι της ποινική δίωξη είναι η απάντηση σε όσους αντιστέκονται. Ε, υπάρχουν λοιπόν ε, Ανάλογε καταστάσει από τη δεκαετία του 70 που μα θυμίζουν το τι γίνεται σήμερα. Το καθεστώ Μακάρθη χρησιμοποιούσε τέτοια επιχειρήματα για να καταπιέζει του πολίτε και να απαγορεύει την ελευθερία τη έκφρασή του. Υπήρχε μια, ένα απόλυτα τυραννικό καθεστώ και κανεί δεν μπορούσε να αντισταθεί ακριβώ επειδή η κυβέρνηση κατέπνιγε οποιαδήποτε μορφή αντίστασης. Ε, ε, σήμερα πια τα πράγματα έχουν ξεφύγει από κάθε έλεγχο, διότι τεχνικά μέσα δίνουν απεριόριστε δυνατότητε. Θα πρέπει λοιπόν οι άνθρωποι στι ΗΠΑ και παντού να μην αποφεύγουν την, ε, τον αγώνα για την προσωπική του προστασία. Είναι θέμα δική του προστασία και όχι αυτό που ισχυρίζεται η κυβέρνηση ότι αυτή προστατεύει του πολίτε καταγράφοντα στοιχεία, στοιχεία του. Αφού συνθλίβει οποιονδήποτε προσπαθεί να καταγγείλει τις μεθόδους της. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει διαφάνεια και νομιμότητα στην κάλυψη των δικαιωμάτων των πολιτών εφόσον θέλουν να εκφραστούν ελεύθερα. Θα πρέπει να εκτίθενται οι κυβερνητικοί οι κυβερνητικές υπηρεσίες που διαπράττουν αυτές τις αδικίες. Ελπίζω ότι η Επιτροπή σας θα μπορέσει να προχωρήσει σε νομοθεσία ευρωπαϊκών διαστάσεων για να προσφέρει ανάλογη προστασία στους Ευρωπαίους πολίτες παρά τα τεχνολογικά μέσα που προσφέρονται που θα πρέπει να βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών παρά να την καταστρέφουν. Θα πρέπει εδώ να δούμε πώς η μαζική παρακολούθηση αποτελεί απειλή και πώς οι σχετικοί νόμοι δεν αρκούν για να προστατεύουν τους πολίτες. Τα δικά σας κάτι μέλη πώς προστατεύονται από το καθεστώς παρακολούθησης. Υπάρχει σαφής ανάγκη για πολιτικές που να προστατεύουν τους πολίτες από τις χώρες και από την πρόσβαση των ε, μυστικών υπηρεσιών άλλων χωρών στην ιδιωτική σφαίρα των πολιτών. Εδώ θα πρέπει να ε, λογοδοτήσουν όλες οι διακρατικές εταιρείε και οντότητες που ε, για λόγους εμπορικούς και τα συμφέροντά τους ε, δίνουν τα στοιχεία των πολιτών σε τρίτα μέρη. Η περίπτωση του πρίσμου είναι πολύ χαρακτηριστική. Βλέπουμε πως ε, κάποιοι κρατούνται όμοιροι ε, από την καταγραφή των δεδομένων τους. Με συγχωρείτε κύριε Ντρέικ. Οι διερμηνείς μου λένε ότι πρέπει να επιβραδύνετε λίγο. Αν μπορείτε να πληρώνετε σιγά σιγά. Δεδομένων των όσων συνέβησαν σε μένα προσωπικά δεν μπορώ παρά να τα επιβεβαιώσω όλα αυτά. Ε, εάν θέλουμε να το δούμε συνολικά, έπρεξα τυχερό. Δεν έζησα όσα συνέβησαν με το πρίσμ. Αλλά βλέπουμε ότι η εξουσία ε, την ε, ανυπακοή και την ατομική συνείδηση τα καταπνίγει σε αυτήν την περίοδο. Αυτό που χρειάζεται η ελεύθερη και ανοιχτή κοινωνία δεν είναι ένα ψηφιακό φράγμα γύρω μας, το οποίο να καταγράφει κάθε μα κίνηση. Αυτό είναι, είναι, καταλήγει στο να θέλουν ε, οι μυστικές υπηρεσίες να ξέρουμε τι σκεφτόμαστε και αισθανόμαστε, την πραγματική ουσία του ανθρώπου που είμαστε ο καθένας μας. Ευχαριστώ. Thank you Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη δήλωση. Έχουμε μία σύνδεση με τον κύριο Βίμπε ο οποίος βρίσκεται στη Washington. Μας ακούτε? Good afternoon to Europe. Hello, you Mr. Okay? <clears throat> Mr. Aguilar, members of the Committee on Civil Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να χαιρετήσω το, την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα που μπορώ να βρεθώ ε, από την Ουάσιγκτον, αλλά να πάρω το λόγο ενώπιόν σας. Πραγματικά θα ήθελα να πω ότι εμείς είμαστε η μόνη προστασία, μη η προστασία για τους ανθρώπους που προσπαθούν να προσπίσουν τη συμβολή της ελευθερίας ανά τον κόσμο. Βεβαίως πολλά άτομα έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στη διάρκεια της ιστορίας μας για να αλλάξει το Σύνταγμα των Ηνωμένων εδώ και έναν αιώνα. Και θα αναφερθώ εδώ στη τέταρτη τροπολογία του συντάγματος που προστατεύει αυτές τις ελευθερίες και βεβαίως υπάρχει για να διαπιστώσουμε ότι πολλές φορές παραβιάσεις της ε, ιδιωτικής σφαίρας, της ιδιωτικότητας και της προσωπικής ζωής έχουν κάποιους λόγους. Ο Μάικλ Χέιντον έλεγε ότι δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε αυτή την τέταρτη τροπολογία σε κάθε περίπτωση, αλλά βεβαίως θα πρέπει να υπάρχουν αρκετά βάσιμες υπόνοιες ότι υπάρχουν παράνομες πράξεις και παραβίαση κάποιων βασικών ε, Είναι πάρα πολύ σημαντικό εδώ να υπάρξει μια συνειδητοποίηση του τι συνέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Τα πράγματα άλλαξαν και βεβαίως ο Μαρκ Χέιντεν όταν πήρε το λόγο μπροστά στο Κογκρέσο διαπίστωσε ότι βεβαίως υπάρχουν πολλές περιπτώσεις να δεχθεί κανείς κάποιες τέτοιες ε, πιο βάσιμες ε, περιπτώσεις που μπορεί κανείς να επικαλεστεί αυτήν την τέταρτη τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος από ό,τι πριν. Και είδαμε ότι εδώ το Κογκρέσο υποχώρησε όταν βεβαίως διαπιστώσαμε κατόπιν ότι η NSA είχε αρχίσει να συλλέγει πληροφορίες επί Αμερικανών πολιτών, διαπιστώσαμε ότι τα πράγματα άλλαξαν πολύ και ότι δεν ήταν αυτός ο αρχικός σκοπός ούτε η πρόθεση του Κογκρέσου. Βεβαίως χάρη στον Σνόουντεν σήμερα γνωρίζουμε πράγματα τα οποία μας οδήγησαν σε κάποιες διαπιστώσεις. Ξέρουμε ότι ο Βίλιαμ Όντεν και ο Μπάμπι Ίμμεν, οι οποίοι εργαζόταν προηγουμένως στην NSA, σήμερα είναι στην σύνταξη, έχουν επικαλεστεί αυτές τις υποθέσεις και βεβαίως πρόσφατες αποφάσεις των Αμερικανικών δικαστηρίων θα έπρεπε να οδηγήσουν, αν είχαν αναδρομική ε, ισχύ, στην ε, προσφυγή κατά του Προέδρου Μπούς. Δεν θέλω εδώ να σας ε, υπενθυμίσω παρά κάποιες περιπτώσεις γερουσιαστών όπως του κυρίου Κέννη ο οποίο, όταν αναφέρθηκε σε αυτή την υπόθεση έλεγε ότι δεν θα μπορέσει να ελέγξει τον εαυτό του και τις αντιδράσει του. Γιατί ήταν τόσο εκνευρισμένος και οργισμένος ε, ο κ. Κέννη, καθότι στην προσπάθειά τους να προσπιστούν και να προστατεύσουν το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά όλων των εχθρών, εντός και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, παραβίασαν πολύ συγκεκριμένη νομοθεσία. Η NSA έχει σαν κύριο κανόνα ότι η πρώτη εντολή του NSA είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί κανείς χωρίς εντολή δικαστηρίου, δικαστική εντολή, να παρακολουθήσει Αμερικάνο υπήκο. Και πραγματικά πολύ σοβαρές προσωπικότητες και άνθρωποι που επί χρόνια εργαζόταν στην NSA ήδη από το 1978 αναφέρθηκαν στις περιπτώσεις παραβιάσεων όπως αυτές τις οποίες αναφέρθηκε ο Χέιντεν. Έλεγε, παραδείγματος χάρη, ότι κανείς δεν μπορεί παραβιάζοντας τον νόμο να κάνει πράγματα τα οποία είναι παράνομα επικαλούμενος την προστασία του συντάγματος ή της εθνικής ασφάλειας. Και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί κανείς παρά να δράσει εντός της νομοθεσίας ή να τροποποιήσει την νομοθεσία αν αυτό είναι απαραίτητο. Εάν δεν μπορεί να τροποποιήσει κάποιος την νομοθεσία, αλλά προσπαθεί μέσω των διαφόρων νομικών τεχνασμάτων εντός και εκτός των νομικών υπηρεσιών να παραβιάσει τα δικαιώματα των ε, Αμερικανών πολιτών, παρόλα αυτά αυτό θεωρείται παράνομο με την στήριξη και τη βοήθεια της σημερινής σύγχρονης τεχνολογίας δεν υπάρχει κανένας λόγος να παραβιάσει κανείς και να θυσιάσει την ελευθερία, την δημόσια ελευθερία έτσι ώστε να υπάρξει ασφάλεια και να αναλύσει κανείς προσωπικά δεδομένα. Θα σας δείξω εδώ σε αυτή τη διαφάνεια τον ορισμό του περιεχομένου. Ξέρετε ότι όσον αφορά την ηλεκτρονική παρακολούθηση, υπάρχουν δύο κατηγορίες ε, πληροφοριών. Τα μεταδεδομένα και το λεγόμενο περιεχόμενο, metadata και content. Με συγχωρείτε, θα ήθελα να σας διακόψω. Η παρουσίασή σας αυτή πρέπει να σας πω είναι στους φακέλους σας. Ναι, θα ήθελα απλώς να σας δώσω κάποια παραδείγματα περιεχομένου, content. Πρόκειται, παραδείγματος χάρη, για ένα έγγραφο όπως ένα ηλεκτρονικό μήνυμα, είτε μία τηλεφωνική διάσκεψη, είτε ένα τηλεφώνημα, είτε ένα αρχείο. Όταν χρησιμοποιεί κανείς, παραδείγματος χάρη, το τηλέφωνό του, έναν αριθμό και βλέπουμε ότι τα τηλέφωνα αυτούς των οποίων τηλεφωνείτε θα χαρακτηριστούν σαν μεταδεδομένα, όπως και το δικό σας τηλέφωνο. Το ίδιο μπορώ να πω και για κάθε είδους ε, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, στο facebook, στο twitter, όλα αυτά θεωρούνται μεταδεδομένα. Τα ονόματα επίσης. Οι πινακίδες ενός αυτοκινήτου, ο τίτλος μιας φωτογραφίας, το μέγεθος, τα δεδομένα, τα πιξέλ μιας φωτογραφίας. Όλα αυτά είναι παραδείγματα του τι είναι ένα μεταδεδομένο. Και ο τρόπος με τον οποίο παρακολουθούμε... Α, βλέπετε αυτήν την διαφάνεια και θα σας δώσω ένα παράδειγμα της απειλής. Στις Ηνωμένες Πολιτείες το περιεχόμενο μπορεί να μην αποκαλυφθεί, μπορεί να μην μπορεί συγγνώμη να αποκαλυφθεί χωρίς δικαστική εντολή. Παρ' όλα αυτά, τα μεταδεδομένα μπορούν να αλλαληθούν να εντοπιστούν χωρίς απολύτως καμία προηγούμενη άδεια από καμία αρχή. Τα μεταδεδομένα λοιπόν, από τη στιγμή που κάποιος ας πούμε ακουμπάει ένα σύστημα ηλεκτρονικό πληροφοριών, αφήνει ένα ε, σημάδι, αφήνει ένα αποτύπωμα. Αυτά όλα τα σημάδια, τα αποτυπώματα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συλλογής όλων αυτών που αποφασίζουν να μας παρακολουθήσουν. Υπάρχουν λοιπόν διάφορες βάσεις δεδομένων με όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία μπορούν να παρουσιαστούν με μια χρονολογική σειρά, αν θέλετε, ορολογιακή σειρά. Παρακολουθούμε λοιπόν από τις 6 το πρωί κάποιον, από τις 6 το πρωί μέχρι τις 9 ε, το βράδυ και βλέπετε εδώ όλες τις ηλεκτρονικές συναλλαγές τις οποίες συμμετέχει και τι αποτυπώματα αφήνει αυτός ο άνθρωπος. Εδώ βλέπετε ποια μπορεί να είναι η παράνομη χρήση αυτών των προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών. Πρόκειται για την υπηρεσία των ειδικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών για τα ναρκωτικά. Και εδώ βλέπετε τους κανόνες τους οποίους υπόκειται αυτή η υπηρεσία και βλέπουμε ότι οι πληροφορίες NSA βεβαίως χρησιμοποιούνται και από άλλες υπηρεσίες κυβερνητικές των Ηνωμένων Πολιτειών έτσι ώστε να μπορέσουν να διεκπαιρεώσουν τις αποστολές τους. Και δεν είναι πολύ ενδιαφέρον διότι πρόκειται για παράνομες δια... δραστηριότητες κάποιων ε, οι οποίοι πολλούν ναρκωτικά. Στην δεύτερη ε, αυτή διαφάνεια όσον αφορά την παράνομη χρήση αυτών των προσωπικών δεδομένων βλέπετε ότι εδώ κρύβεται, δεν αποκαλύπτεται τουλάχιστον η πηγή αυτών των δεδομένων και προσωπιών. Και αυτό που θέλει εδώ να κάνει το αμερικανικό δικαστικό σύστημα είναι να αποκρύψει κάθε πιθανή πηγή, τον εντοπισμό πηγής από την οποία προέρχονται αυτά τα προσωπικά δεδομένα. Να καλύψει λοιπόν αυτή την πηγή και να παρουσιάσει αυτές τις πληροφορίες σαν να είναι πληροφορίες οι οποίες απορρέουν από μια κανονική τυπική έρευνα παραδείγματος χάρη του FBI. Στις Ηνωμένε Πολιτείες καταλαβαίνετε ότι η υπόθεση Smith vs. Merlin του 79 προϋποθέτει ότι για να υπάρξει εκτεταμένη και μαζική συλλογή τηλεφωνικών μεταδεδομένων χρειάζεται δικαστική εντολή. Εδώ πρόκειται για μια υπόθεση μιας κλοπής ο διαρρήκτης κάλεσε, τηλεφώνησε στο θύμα και χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα αυτής της τηλεφωνικής συνδιαλλαγής, την οποία μάλιστα παρενόχλησε ε, το θύμα, στο δικαστήριο. Και εδώ πραγματικά είναι τελείως παράλογο σε τέτοιες περιπτώσεις να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα δεδομένα. Αυτή η υπόθεση θα πρέπει να επανεξεταστεί. Το 79 βεβαίως ο δικαστής, καθότι δεν υπήρχαν οι τεχνολογικές δυνατότητες που έχουμε σήμερα, δεν μπορούσε να διανοηθεί τις επιπτώσεις που μπορούσε να έχει μια τέτοια υπόθεση και μια τέτοια απόφαση. Σήμερα που διαθέτουμε όλα αυτά τα ηλεκτρονικά δίκτυα και τα αποτυπώματα και τα σημάδια που αφήνει οποιαδήποτε ηλεκτρονική συνδιαλλαγή, όπως ε, χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών δικτύων πιστοτικών καρτών κτλ. Σήμερα βεβαίως υπάρχει η βασική αρχή της προστασίας της ιδιωτικότητας, της προσωπικής ζωής, των προσωπικών δεδομένων. Και κανείς δεν μπορεί να παραβιάσει αυτές τις θεμελιώδεις ελευθερίες, εκτός αν υπάρχει βάσιμη υποψία ή απόδειξη ότι οι δραστηριότητες αυτού του ανθρώπου αποτελούν απειλή για την δημόσια ασφάλεια. Και δεν ξέρω ποια είναι ακριβώς η αντίστοιχη περίπτωση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά τουλάχιστον από ό,τι ξέρω πρόκειται για μια παρόμοια περίπτωση σαν αυτή που ισχύει στις ΗΠΑ. Χρειάζονται βάσιμες πληροφορίες και όχι απλώς κάποια υπόνοια ή μη επιστημονική ε, έρευνα που οδήγησε σε ένα τέτοιο συμπάρασμα. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας δείξω ότι υπάρχουν δύο επίπεδα διαχωρισμού της ανάλυσης και των δεδομένων. Η απειλή εδώ στην ιδιωτική ζωή και στα προσωπικά δεδομένα είναι τα ηλεκτρονικά συστήματα. Τα εργαλεία αυτά, τα οποία όμως την ίδια ώρα, ταυτόχρονα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προστατεύσουν τα προσωπικά δεδομένα. Η ανάλυση οδηγεί στην παραβίαση της προσωπικής, των προσωπικών δεδομένων. Βλέπετε εδώ, έχουμε έναν ύποπτο, ο John Doe, ο οποίος ζει στην Καλιφόρνια. Είναι ένας ύποπτος είναι ο κακός, είναι τρομοκράτης ας πούμε, ο οποίος έρχεται σε επαφή με τον άλλο ύποπτο, ο οποίος είναι με κίτρινο χρώμα και όλες οι πληροφορίες με κίτρινο χρώμα είναι οι πληροφορίες οι οποίες κανονικά προστατεύονται. Και βεβαίως κανονικά η ανάλυση δεν θα πρέπει να τις αποκωδικοποιήσει. Θα πρέπει δηλαδή να παραμείνουν υπόκρυπτα ανάλυση χωρίς να αποκαλυφθούν τα οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία και προσωπικά δεδομένα αυτού του υπόπτου. Δεν υπάρχει ανάγκη όλα αυτά τα στοιχεία να αναλυθούν, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για αθώους. Βλέπετε εδώ ότι αυτός ο οποίος καλείται να αναλύσει αυτές τις πληροφορίες μπορεί να αναλύσει όλα τα στοιχεία που αφορούν τον Τζον Ντο. Αν ο ύποπτος με κίτρινο χρώμα στη διαφάνειά μας αποδειχθεί ότι εμπλέκεται σε κάποια ποινική πράξη, σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να θεωρήσουμε ότι και τα δικά του προσωπικά δεδομένα πρέπει ή μπορούν να αποκαλυφθούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάμε σε ένα δικαστήριο, γιατί τα κριτήρια τα οποία θα θεωρήσει βάσιμα ο, το δικαστήριο, ο δικαστής για να υπάρξει αποκάλυψη αυτών των στοιχείων είναι μία σειρά, αν θέλετε, κανόνων και κριτηρίων που θα πρέπει να έχουν καθοριστεί βεβαίως από το δικαστήριο, από τη δικαστική αρχή και κατόπιν εμείς βάσει αυτών των κανόνων η υπηρεσία παρακολούθησης μπορεί να πάρει την απόφαση σε δευτερόλεπτα αν ναι ή όχι πρέπει να αποκαλυφθούν αυτά τα στοιχεία. Και με αυτόν τον τόπο προστατεύουμε τους αθώους Αμερικανούς πολίτες. Ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά πρέπει να ολοκληρώσετε. Ναι, ναι, τελείωσα. Δυστυχώς ε, πρέπει να παρακολουθώ και το χρόνο ομιλία σας. Ε, αν μπορείτε να ολοκληρώσετε και μετά να μπορέσετε να προσθέσετε ίσως κάποια στοιχεία ε, στις ερωτήσεις που θα σας τεθούν. Ε, ναι, ολοκληρώνω γιατί αυτό ήταν το τελευταίο μου σχόλιο. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ε, ε, Ήρθα σε δύσκολη θέση τώρα. Λοιπόν, προτείνω να θέσουμε ερωτήσει προς τον κύριο Βίντεο αμέσω ε, και να μην περιμένουμε το τέλος τη συνεδρίαση, γιατί έχουμε αυτή τη σύνδεση μέσω βίντεο και προτείνω να περιορίσουμε τις ερωτήσεις ε, στον εισηγητή και στους κοιόδη εισηγητέ. Κύριε Μωράς, δεν έχετε ερωτήσεις, ωραία. Ο κύριος Βος από το ΕΛΚ. Ε, θα γίνουν ερωτήσεις στα αγγλικά. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, σας παρακαλώ πέστε μου το. Ωραία, σας ευχαριστώ. Μπορώ να θέσω ερωτήσεις στα γερμανικά. Είπατε ότι σε σχέση με την ανάλυση των δεδομένων και την εκτίμηση με ενδιαφέρει ιδιαίτερα αν η αξιολόγηση, η εκτίμηση αυτών των δεδομένων γίνεται μόνο για την αξιολόγηση κάποιων κινδύνων, είτε αυτή η εκτίμηση γίνεται και πολιτικά και με επιστημονικό τρόπο. Μπορείτε να απαντήσετε αυτή την ερώτηση. Ναι. Στις Ηνωμένε Πολιτείε η χάρτα του NSA του ε, εξουσιοδοτή να ερευνά θέματα ε, πληροφοριών οποιοδήποτε ε, οποιασδήποτε μορφής υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για ξένους στόχους. Αυτό βασικά περιγράφεται στη χάρτα. Τώρα, το τι γίνεται με το πώς εφαρμόζεται στην πραγματικότητα είναι ξεχωριστές συμφωνίες με διάφορες χώρες ανά τον κόσμο και συνήθως αυτές οι σχέσεις καθορίζονται από εταιρικές σχέσεις και συμπράξεις με ε, οργανισμούς πληροφοριών ε, που εδράζουν στα Ηνωμένα Έθνη και κάποιους άλλους όχι. Υπάρχουν διάφορες διακλαδώσεις και διάφορες μορφές ε, συνεργασίας, είτε είναι ευρύτερε είτε στενότερες, ανάλογα με τις συμφωνίες αυτές. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενη ερώτηση από τον κύριο Άλπρεχτ από τους Πρασίνους. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να μου πείτε σε ποιο βαθμό προβλέπετε να γίνεται εκ των προτέρων διατήρηση των μεταδοδημένων και αν αυτό αφορά και πρόσβαση σε βάσει δεδομένων ε, επιχειρήσεων που βρίσκονται στο εξωτερικό ε, από τον NSA. Εξαιρετική ερώτησή σας και να σας πω το εξή. Στο σημερινό κόσμο δεν έχει τόσο σημασία πού βρίσκονται τα δεδομένα, διότι αυτή τη στιγμή είναι συνδεδεμένα με το παγκόσμιο διαδίκτυο κατά κάποιον οποιονδήποτε τρόπο υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης από κάποιο οργανισμό ή από κάποια υπηρεσία και ο μόνος παράγοντας ο οποίος δρά ως ανασταλτικός παράγοντας είναι ε, η δυνατότητα μέσω λογισμικού να προστατεύονται ή να κωδικοποιούνται ε, και να μην υπάρχει πρόσβαση στο πρωτόκολλο. Ο μόνος τρόπος λοιπόν να προστατεύονται τα δεδομένα οπουδήποτε βρίσκονται είναι να είναι πολύ υψηλή η κωδικοποίηση και ο κλειδάριθμος για την αποκωδικοποίηση να μην βρίσκεται στα, χέρια του οργανισμού παρακολούθησης πληροφοριών αλλά ε, στα χέρια ενός δικαστηρίου ή κάποιον εξάρτητου φορέα ο οποίος θα διασφαλίζει ότι η αποκωδικοποίηση και οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται για την αποκωδικοποίηση δεν είναι διαθέσιμοι σε κανέναν για να τους χρησιμοποιούν και να το δοκούν. Τώρα, εάν πρέπει τα δεδομένα να βρίσκονται σε κάποιον ε, ε χώρο για να προστατεύονται θα πρέπει να προστατεύονται και από το hacking και, και επομένως θα πρέπει να χρησιμοποιείται η κωδικοποίηση ως φραγμός. Στις ε, διαφάνειες που σας έδειξα, στην τελευταία εικόνα με τη σύνδεση που γίνεται με τις τελείες, δεν χρειάζεται να δίνονται δεδομένα τα οποία δεν έχουν σχέση με εγκληματική ή τρομοκρατική δραστηριότητα. Θα πρέπει να, ε, γίνεται, να δίνεται ένταλμα από το δικαστήριο και να λαμβάνονται τα στοιχεία αναπερίπτωση. Εμείς αυτή την νομοθεσία θα θέλαμε για αυτές τις περιπτώσεις. Σας ευχαριστούμε. Δεν είναι κανείς εδώ σε μέρους των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Δημοκρατών. Η κυρία Έρστ. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ σύντομα είπατε ότι επίτηδες αποκρύπτονται, καλύπτονται οι πηγές έτσι ώστε να μην μπορεί κανείς να ανατρέξει και να δει πώς προέκυψαν αυτές οι πληροφορίες. Μπορείτε να μου πείτε ποιες είναι οι συνέπειες αυτού που μας είπατε με λίγο περισσότερες λεπτομέρειες. Um, yes. Uh, ναι. Όταν γίνεται παρακολούθηση από τις υπηρεσίες πληροφοριών, και κάνουν αυτό το οποίο θα επιθυμούσαμε όλοι να κάνουν, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να προστατεύονται οι πηγές τους και οι μέθοδοί τους. Αυτά είναι τα δύο στοιχεία τα οποία πρέπει να προστατεύονται ώστε να μπορούν να φυλάσσονται τα μυστικά. Οι πηγές και οι μέθοδοι. Εάν όμως τα στοιχεία δεν χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιούνται εντός ε, της χάρτας του οργανισμού, εκτός συγγνώμη, της χάρτας του οργανισμού και στις Ηνωμένε Πολιτείες υπήρχε μια παραδοσιακή διαχωριστική γραμμή μεταξύ των πληροφοριών και της εφαρμογής της νομοθεσίας και μάλιστα αυτή η διαχωριστική γραμμή υπήρχε επί τούτου ώστε να μην είμαστε ένα μεγάλο αστυνομούμενο κράτος το οποίο καταπιέζει και καταχράζεται στοιχεία. Και δυστυχώς αυτό βλέπουμε. Έχουμε φτάσει πλέον σε ένα αστυνομούμενο κράτος όπου παρακολουθούνται οι πάντες και δίνονται πληροφορίες σε διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες. Έχουμε πλέον ένα παράδειγμα το οποίο ε, έχουν συλλέξει νομικοί και έχετε και δύο διαφάνειες οι οποίες αναφέρονται στο τμήμα ειδικών υπηρεσιών της ε, υπηρεσίας ε, καταπολέμησης των ναρκωτικών που αναφέρονται σε αυτό ακριβώς που συζητάμε. Πώς επηρεάζεται τώρα ο πολίτης. Μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο και να μην γνωρίζει ότι κατηγορείται με βάση στοιχεία τα οποία πραγματικά δεν δόθηκε έγκριση από την κυβέρνησή σας για να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία. Δηλαδή η κυβέρνηση δρά εκτός κανόνων που εσείς ως πολίτης σέβεστε και ουσιαστικά ε, είναι και τμήμα της ζωής σας. Αυτό λοιπόν είναι ακριβώς αυτή η απειλή, η δραστηριότητα η οποία μπορεί να υπονομεύσει πολλές από τις πολιτικές ελευθερίες στον τομέα αυτό. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Μορβά ήθελε να κάνει μια ερώτηση, επειδή δεν είναι σκιώδη ηχιάτρια ή δυνατόν αν μπορεί να είναι πολύ σύντομη. Ως ε, πρώην υπάλληλο της NSA, τι απαντάτε σε αυτούς που λένε ότι ναι, συλλέγουμε μεν όλα αυτά τα στοιχεία, αλλά τα χρειαζόμαστε για λόγους εθνικής ασφάλειας, θέλουμε να καταπολεμήσουμε τους τρομοκράτες με αυτή τη συλλογή στοιχείων. Και δεύτερη ερώτηση, ε, θα ήθελα να το ακούσω και από εσά παρά το γεγονός ότι και εγώ αυτό πρεσβεύω. Εξ όσων γνωρίζετε, από πού συλλέγονται τα στοιχεία κάποιων σαν αυτόν που συλλεγονται τα στοιχεια καποιον σαν εσείς στο παράδειγμα στη διαφάνεια Ποιος χρησιμοποιεί αυτά τα στοιχεία και για ποιο σκοπό. Είναι προφανές ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν για τα καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ποιος χρησιμοποίησε λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία ζητήθηκαν από την NSA και ποιος ήταν ο σκοπός της συλλογή τους. Ναι. Ένα οργανισμό που κάνει ηλεκτρονικέ παρακολουθήσει για ένομου λόγου, δεν χρειάζεται όλα τα στοιχεία. Χρειάζεται απλώς πρόσβαση σε κάποια από τα στοιχεία, οπουδήποτε και αν βρίσκονται. Και πάλι όμως όλο αυτό βασίζεται στην πιθανή αιτία, στο στοιχείο της πιθανής αιτίας. Η διαδικασία λοιπόν ε, στόχο έχει να παρισφρήσει σε όλο τον κόσμο των δεδομένων, των μεταδεδομένων και του περιεχομένου. Και ο στόχος θα πρέπει να είναι πάντα για όλους όσους ε, βρίσκονται πιο κοντά σε εγκληματική δραστηριότητα, όταν δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο δράστης και απλώς αναζητούμε αποδείξεις εγκληματικής δραστηριότητας, παραδείγματος χάρη, ιστοσελίδε ε, τζιχαντιστών, ε, κάποιοι οι οποίοι συμμετέχουν σε ριζοσπαστικές οργανώσεις, κάποιοι οι οποίοι συζητούν ή συνομιλούν για την αγοραπολισία ναρκωτικών και αντίστοιχα τέτοια πράγματα στο διαδίκτυο. Ε, γίνεται λοιπόν αναζήτηση σε δημοσίως διαθέσιμα δεδομένα. Από εκεί ξεκινούμε. Αν όμως δεν υπάρχει κάποια αφετηρία, όπως ε, σας έδειξα στο παράδειγμα μου προηγουμένως, δεν χρειάζεστε όλα τα δεδομένα του κόσμου για να αναζητήσετε αυτές τις λίγες σχέσεις που έχει ο πιθανός δράστης με τους υπολείπους ανά τον κόσμο και εκεί θα πρέπει να επικεντρωθείτε όταν κάνετε την ανάλυση των πληροφοριών σας. Δεν χρειάζεστε δηλαδή όλα τα στοιχεία εκ των προτέρων για να επιτύχει, επιτύχει η αποστολή σας. Χρειάζεστε απλώς τα σχετικά στοιχεία και να υπάρχουν ένα-δύο διαχωριστικές γραμμές από την αρχική σας πληροφορία. Παραδείγματος χάρη αυτόν τον ανώνυμο ύποπτο που είχαμε ε, στα στοιχεία. Είπατε, πού είναι τα στοιχεία για τον Bob. Θα μπορεί να βρίσκονται σε κάποιους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών, σε, υπηρεσίες, σε εταιρείες τηλεπικοινωνιών, μπορεί να βρίσκονται και στον κόσμο του εμπορίου φανταστείτε, στοιχεία τα οποία περνούν ε, από τους διάβλους του διαδικτύου. Όλα αυτά μπορούμε να τα λάβουμε μέσω δικαστικού εντάλματος, το οποίο θα έχει ζητήσει κάποια νομική αρχή, όπως για παράδειγμα ένας δικαστής, ή ε, Μέσω λογισμικού το οποίο καθορίζει ένας δικαστής σε ένα δικαστήριο. Δεν χρειάζεται να τα πάρουμε όλα, να τα έχουμε σε μια μεγάλη βάση δεδομένων και να ελπίζω ότι μια μέρα μπορεί να τα χρειαστείτε. Αυτό δεν είναι απαραίτητο. Λυπάμαι κυρία Μορβάη, αλλά δεν έχουμε άλλο χρόνο, καθυστερούμε και θα ήθελα πραγματικά να θέσω και εγώ μια ερώτηση εξ ονόματος των φιλελευθέρων και μετά θα περάσουμε στον επόμενο γύρο ερωτήσεων. Δύο ερωτήσεις. Αναφερθήκατε στο ήθο εσεί στο τέλο τη παρέμβασή σα, έγινε μια αναφορά από τον κύριο Γκρέι και στο Σύνταγμα και φαντάζομαι ότι η κυρία ε, Μέισον αργότερα θα αναφερθεί σε κάτι αντίστοιχο. Εσείς ξεκινήσατε να εργάζεστε στην NSA πιστεύοντας ότι όλα γίνονται σε ένα συγκεκριμένο συνταγματικό πλαίσιο. Τι σας έκανε να στραφείτε προς τα έξω, να επικρίνετε την NSA και να δώσετε πληροφορίες για αυτά τα οποία γίνονταν. Και ε, ποια είναι γενικότερα η αίσθηση. Έχουν και άλλοι αμφιβολίες, θέλουν και άλλοι να επικρίνουν την NSA και θεωρούν ότι μπορούν με ασφάλεια να ε, διαρρεύσουν πληροφορίες. ε, λέτε ότι κανονικά θα έπρεπε να τα αναλαμβάνουν όλα τα δικαστήρια, αλλά δεν αναφέρεστε σίγουρα σε ένα δικαστήριο το οποίο δεν λειτουργεί αποτελεσματικά. Για την πρώτη σας ερώτηση, γιατί επέκρινα εγώ, γιατί έγινα εγώ whistleblower πληροφοριοδότης. Έγινα για δύο λόγους. Υπήρξα μάρτυρας διαφθοράς, κακοδιαχείρισης εντός της NSA, ε, και σε σε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ε, πληροφοριών. Ένα διέρευσε και στα ε, ε, ειδήσει, το λέγανε Trailwazer και στον καιρό μου κάποιοι από εμά στο κτίριο ξέραμε ότι θα αποτύχει αυτό το πρόγραμμα διότι δεν ήταν καλά οργανωμένα αυτή εξ αρχής. Ε, και οι προϋποθέσεις επί των οποίων έγινε ήταν λαθασμένες. Πολύ συχνά γίνεται ε, αυτό σε οργανισμούς όπως τον NSA, οι καλές ιδέες παραγωνίζονται ε, εις βάρος κάποιων άλλων που εξυπηρετούν εμπορικά συμφέροντα και δυστυχώς αυτό το υποβοηθούν κάποιοι στο Κογκρόεσο οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε αυτά τα επιχειρηματικά συγχέροντα. Πολλά λοιπόν τα προβλήματα διαφθοράς προκαλούνται από τις ίδιες μας τις κυβερνήσεις. Και ο άλλος λόγος ο οποίος επέκρινα είναι γιατί ο κύριος Μπένι, ο συνάδελφό μου, ε, ε, έλαβε πληροφορίες ότι η NSA παρανόμως συνέλεγε στοιχεία και εξέταζε στοιχεία τα οποία δεν είχε εξουσιοδότηση να εξετάζει. Πιο συγκεκριμένα στοιχεία ε, Αμερικανών πολιτών. Ποια λοιπόν είναι η δεύτερη ερώτησή σας και πάλι συγγνώμη. Ρώτησα αν νιώθουν ελεύθεροι οι υπόλοιποι και θεωρούν ότι θα μπορούσαν με ασφάλεια να επικρίνουν τα όσα γίνονται στην NSA ε, και ρώτησα και κάτι για τα δικαστήρια. Όχι, δεν νιώθουν ασφαλείς. Ε, μπορεί κάποιοι ε, να ήθελαν να μιλήσουν και αυτοί, αλλά επειδή έχουν θέσει εργασίας και εξαρτώνται από την κυβέρνηση για το εισόδημά τους και την ευημερία τους, φοβούνται να μιλήσουν είναι μια φρικτή μορφή καταπίεσης αυτή και ελευθερίας των πληροφοριών, αλλά είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι θα ήθελαν να δώσουν πληροφορίες. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις από πλευρά μας. Θα συνεχίσουμε γιατί έχουμε καθυστερήσει λίγο. Η τελευταία μιλήτρια σε αυτό το τμήμα είναι η κυρία Μάσον, πρώην υπάλληλος της MI5. Σας ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσετε εδώ. Ευχαριστώ την Επιτροπή σας. Θα μιλήσω για τις μυστικές υπηρεσίες στον Ηνωμένο Βασίλειο και τις νομικούς περιορισμούς, καθώς και το τι γίνεται με τους πληθωροειδότες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης υπάρχουν και κάποιες συστάσεις, τις οποίες θα ήθελα να σας τις υποβάλω, ώστε να έχουμε και ένα αντικείμενο συζήτησης ε, σε λίγο. Για όσους ε, ενημερωτιέστε πώς είμαστε οργανωμένοι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είμαστε διαφορετικοί από τις Ηνωμένες στην στη διοργάνωσή μας και οι μυστικές υπηρεσίες δημιουργήθηκαν πριν από 100 χρόνια. Τα μέλη του Κοινοβουλίου μάλιστα δεν είχαν δικαίωμα να θέτουν ερωτήματα ως τώρα για να ξέρουν ε, τι συμβαίνει με τις μυστικές υπηρεσίες. Το 1970 ξεκίνησε το πρώτο νομοσχέδιο και η πρώτη νομηθήκη διάταξη για να ε, μην υπάρξει διαρροή πληροφοριών προς την κυβέρνηση, όπου δεν κανείς ε, καταδικαζόταν μάλιστα για δίκημα παραβίασης αυτού του νόμου, μπορούσε να δεχτεί και 40 κάθριξη. Τη δεκαετία του 80 υπήρξαν αυτά σκάνδαλα με πληροφοριοδότες, whistleblowers, και ε, έτσι προβλέφθηκαν νόμοι για να προβλέψουν τις εξελίξεις των όσων θέλω να θίξω σήμερα. Πρώτα απ' όλα, ο νόμος για το, κυβερνητικό απόρριτο, για το κρατικό απόρριτο ε, ανανεώθηκε. Και από το 1980 ε, άλλαξε η διάταξη για το ότι δεν μπορεί το δημόσιο συμφέρον να αντίκειται με την ε, αποκάλυψη πληροφοριών. Εάν κάποιος μιλήσει για τη δουλειά του εκτός υπηρεσίας ε, κρατικής στην οποία δουλεύει, θεωρείται ότι παραβιάζει τον νόμο. Επίσης, από το δεκαετία του 1990 ξεκίνησε άλλη νομοθετική κίνηση για να καλυφθεί και η περίπτωση του κυβερνητικού απορρίτου και το ίδιο και ο επόμενος νόμος που έθεσε τις κρατικές μυστικές υπηρεσίες στην ίδια κατηγορία με τους πληροφοριοδότες. Ε, Κοινοβουλευτική Επιτροπή που έπρεπε να έχει συνολική εποπτεία του έργου των μυστικών υπηρεσιών ανέλαβε την παρακολούθηση αυτή τη δουλειά. Όμω ω σήμερα αυτή η βουλευτική Επιτροπή για τι Μυστικέ Υπηρεσίε παραμένει σχετικά αδρανή και ανώδυνη, διότι είναι πολύ περιορισμένε οι αρμοδιότητέ τη και τα σκάνδαλα τη τελευταία 20 ετία δεν μπόρεσαν να διαλευκανθούν. Ε, κάλεσαν μέλη των μυστικών υπηρεσιών, ε, απίθυναν ε, κατηγορίε εναντίον του και ζήτησαν να γίνουν έρευνε για τι παραβιάσει του απορρίτου, αλλά Συνολικά αυτή είναι η κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι ειρωνικό να το συζητάμε τώρα, διότι είναι κάπως ε, ένοχη η Βρετανία, αν δούμε τι έγινε με την υπόθεση Σνόντεν. Θα ήθελα λοιπόν για το MI5 από το 1990 ε, να πω ότι εκεί εργάζομαι και ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα από νομικές άποψεις όταν ξεκίνησα. Ήταν μια άλλη εποχή. Ε, ήταν πολύ διαφορετικά τα τεχνολογικά συστήματα και ξαφνικά βρεθήκαμε σε μια τελείως νέα κατάσταση όταν ε, οι μυστικές υπηρεσίες πήραν πλέον ε, νέες διαστάσεις. Πολλά έχουν αλλάξει και έχουν πάει και πολύ άσχημα στα χρόνια που εργάζομαι στο MI5. Ε, θέσαμε πολλές από τις ανησυχίες μας και το ίδιο και οι συνάδελφοί μας. Και μάλιστα πολλοί παρετήθηκαν, αλλά μας είπαν να το να μην λέμε τίποτα και να ακολουθούμε τις εντολές που μας δίνουν ε, εκτός των μυστικών υπηρεσιών. Ο David Σέλλορ και εγώ λοιπόν, εγώ τον βοήθησα, αποφασίσαμε να αρχίσουμε να αποκαλύπτουμε πληροφορίες για μια σειρά από αδικήματα που είχαν να διαπραχθεί. Και αυτό κλιμακώθηκε με τα χρόνια στο MI5. Μιλάμε για αδικήματα υπουργών, ανθρώπους που θα έπρεπε να προσπίζονται πρώτα τα δικαιώματα των πολιτών. Ε, Επίσης, αδικήματα κατά αριστερό, αριστερών στα φρονήματα δημοσιογράφων, άνθρωποι που φυλακίζονταν, αλλά μπορεί να ήταν αθώοι, αλλά παραμποδοζόταν η εκδίκαση της υπόθεσής τους. Το MI5 επίση, η υπηρεσία MI5 ε, πολλές φορές είπε ψέματα και στην κυβέρνηση και αυτό ε, ήταν για μας καθοριστικό και γι' αυτό παρατηθήκαμε. Ε, επίση με τη χρηματοδότηση τρομοκρατική ε, ενέργεια στη Συρία για την ενδεχόμενη τηλεφωνία του Καντάφη το 1996 ξέρουμε ότι έχασαν τη ζωή τους ε, αθώοι άνθρωποι γιατί απέτυχε αυτή η απόπειρα. Ξέραμε ότι τέτοια πράγματα είναι σοβαρά δικήματα και από το 1990 με την ε, νομοθετική πράξη που επέτρεπε την αποκάλυψη πληροφοριών αποφασίσαμε να τα δημοσιοποιήσουμε όλα αυτά. Αρχίσαμε να κρυβόμαστε για χρόνια στη Γαλλία Ζήσαμε στη Γαλλία εξόριστη τρία χρόνια συνολικά, γιατί το MI5 ήθελε να μας διώξει. Ε, δύο προσπάθειες έγιναν όταν ε, το Ηνωμένο Βασίλειο ζήτησε την έκδοσή μας από τη Γαλλία το 1998 και μετά, ε, άλλον ένα χρόνο μετά, το Ηνωμένο Βασίλειο ε, θέλησε να μας δικάσει για άλλη κατηγορία, για την παραβίαση του νόμου για το, μυστικό, για το κρατικό απόρριτο. Ήταν ε, φυσικά μια μεγάλη αναστάτωση στις ζωές μας όλη αυτή η εμπειρία με το να χάσουμε τη δουλειά μας, να αλλάξουμε ζωή. Ο Ντέιβιν πήγε φυλακή, εγώ συνελήφθη, ο αδερφός του συνελήφθη επίσης, ε, οι καλύτεροι του φίλοι, δημοσιογράφοι που είχαν σχέση με αυτή την υπόθεση γιατί τόλμησαν να αποκαλύψουν ε, στοιχεία. Ήταν πολύ χρήσιμο το μάθημα αυτό γιατί βλέπουμε πόσο ζούμε σε ένα καθεστώ μόνιμη παρακολούθηση. Όταν δεν μπορεί κανεί να έχει ιδιωτικέ συνομιλίε στο τηλέφωνο ένα στέλνει email χωρί να παρακολουθείτε. Ακόμα και στην, στην, στο χώρο, τον ιδιωτικότερο χώρο του σπιτιού του δεν μπορεί κανείς να έχει μια ανενόχλητη ζωή. Χρειάστηκε λοιπόν να ζήσουμε από αυτό το καθεστώς παρακολούθησης επί σειρά ετών. Αυτό που ήταν ενδιαφέρον στην υπόθεσή μας ήταν να δούμε και πώ ε, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που θα έπρεπε να, να υπερασπίζονται την αποκάλυψη στοιχείων. Πολλέ φορέ και αυτά παρακολουθούνταν παρανόμω. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, μάλιστα, ασκούνταν πιέσει κατά των δημοσιογράφων, ε, απειλέ και το ίδιο βλέπουμε ότι έγινε και στην υπόθεση του Σνόντεν. Αυτό με επιταγές, με εντολές που δεν μπορούσε κανείς ούτε να τις ε, συζητήσει καν. Ε, υπήρχαν μάλιστα κυβερνητικές κινήσεις που λειτουργούν σαν τέτοιου είδους εντολές υπήρχαν ανάλογες νομοθετικές προβλέψεις, εντάλματα κατά των δημοσιογράφων. Ε, ακόμη και για την υπόθεση Σνόντεν είδαμε να ακολουθούνται τέτοιε τακτικέ. Έπειτα το πρόβλημα δεν είναι μόνο να είναι κανεί πληροφοριοδότη όπου μπορεί να δεχτεί ποινικέ διώξει. Ένα δημοσιογράφο μπορεί να διωχθεί βάσει του άρθρου 5 και της πράξης του 1989, εάν θεωρηθεί ότι διαπράττει δίκημα κατά της εθνικής ασφάλειας, αναφέροντας στοιχεία που του έδωσαν πληροφοριοδότες. Αυτό ε, μπορεί να οδηγήσει σε δύο εξανθρώπων όπως έγινε τώρα πρόσφατα στη Ρωσία λόγω χάρη, εκτός Ηνωμένου Βασιλείου. Υπάρχει η Επιτροπή για τις Μυστικές Υπηρεσίες, η ISU όπως την ανέφερα προηγουμένως, αλλά όπως είπα δεν έχουν, δυνατό, δεν έχουν αρμοδιότητες, δεν έχουν εξουσία. Πολλές υποθέσεις της τελευταίας δεκαετίας έδειξαν ότι αυτή η Επιτροπή ε, άφησε πολλούς ανθρώπους ε, να φύγουν ενώ έλεγαν ε, ψέματα στην ε, υπόθεση που διερευνά του. Το θέμα είναι λοιπόν υπάρχει κάποια δημοκρατική, δημοκρατικός έλεγχος όλων αυτών των παρακολουθήσεων. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα κρατικό ένταλμα λόγω χάρη για τους ανθρώπους που αφήσουν να διώξουν οι μυστικές υπηρεσίες. Όμως, ουσιαστικά παρουσιάζεται μόνο η περίληψη μιας περίληψης της περίληψης της περίληψης των στοιχείων που έχουν κεντρώσει οι μυστικές υπηρεσίες. Είναι πολύ δύσκολο αυτό που θα εκδώσει το ένταλμα να καταλάβει αν τεκμηριώνεται η υπόθεση και αν μπορεί να προσφύγει και στην ε, αρμόδια επιτροπή. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και νομίζω ότι το είδαμε και με τον DCHQ την ε, τεχνική παρακολούθηση στέμπλε. Εδώ είδαμε ότι προφανώς είναι παράνομο, ότι προφανώς παραβλέπεται η νομοθεσία, όμως φαίνεται να υπάρχει νομική ασάφεια εδώ. Ένα ένταλμα που μπορεί να καλύπτει εκατοντάδες ε, εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια συνομιλίες. Και αυτό επί σειρά μηνών. Φυσικά αυτό μπορεί να θεωρηθεί αποτελεσματική παρακολούθηση γιατί είναι σημαντικό λοιπόν να υπάρχουν whistleblowers και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν υπάρχει ένα τέτοιο δικαίωμα κατοχυρωμένο στο Σύνταγμα. Ούτε έχουμε γραπτό Σύνταγμα στη... στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ουσιαστικά από την άποψη των μυστικών υπηρεσιών είμαστε λιγότερο προστατευμένη κοινωνία στο δυτικό κόσμο. Είναι πολύ στενό μια κοινοτροπία μα. Δηλαδή, εάν κανεί πει, το να μην, ε, πει στους δημοσιογράφου να μην αμφισβητήσουν τι. Ε, Κρατικέ αποφάσεις μπορεί να τους ε, χειραγωγήσει. Το είδαμε τι έγινε με το MI5 και το MI6, ε, υποθέσεις βασανιστήριων την τελευταία δεκαετία από τον 11 Σεπτεμβρίου του 2001. Ήταν αντιδιοντολογικό και αποτελεσματικό όπως κρίθηκε από τους ε, ειδικού να προσφύγει κανεί τη μεθόδο των, βασανιστήριων. Αυτό το είδαμε και στην περίπτωση τη Βόρεια Ιρλανδία. Όμω τα μαθήματα αυτά δυστυχώ δεν έδωσαν καρπού νομοθετικού. Υπήρξε λοιπόν ηθική εκτραχύλυνση και γι' αυτό ε, μπόρεσαν οι υπεύθυνοι των μυστικών υπηρεσιών να καταφύγουν μέχρι και σε βασανιστήρια. Είναι σημαντικός λοιπόν ο ρόλος των πληροφοριοδοτών εδώ. Άλλωστε, δεν είναι μια υπόθεση που αφορά μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο. Βλέπουμε τι γίνεται στι ΗΠΑ ε, με την πράξη κατά τη κατασκοπία που έχει χρησιμοποιηθεί πολλέ φορέ ω πρόσχημα για να ασκηθούν ε, διώξει κατά των πληροφοριδωτών. Αυτό ξεκίνησε από το 1989 και δεν είναι κάτι που αφορά αποκλειστικά του whistleblowers, αλλά έχει ουσιαστικά καταλήξει να επιφυλάσσει την ίδια μεταχείριση που επιφυλάσσεται στου ε, πραγματικού κατασκόπου. Και ενώ υπήρξε συμφωνία για την προστασία κάποιων πληροφοριοδοτών, τελικά εκδόθηκαν στη Ρωσία. Στη Ρωσία βάσει του νόμου αυτού που έχει χρησιμοποιηθεί επανειλημμένω για να διώκονται οι πληροφοριοδότε τη ΗΠΑ. Είναι υποκρισία αυτό και είναι μάλιστα μια υποκρισία που μα αφήνει άναυδου. Τι γίνεται όμω με το κράτο αυτό που όλο ένα γίνεται και πιο ελεγκτικό, ε, πιο παρεμβατικό τι είδαμε να γίνεται με την υπόθεση Snowden και με τη διάδοση και άλλων αμφισβητούμενων ενεργειών ανά τον κόσμο. Δηλαδή η CIA και οι δράσεις της, η, η δολοφονία, υπόπτων για τρομοκρατικές ενέργειες από τις υπηρεσίε υπηρεσίες των Αμερικανών ή η εισβολή σε κυρίαρχα κράτη με ε, πρόσχημα τις πληροφορία των μυστικών υπηρεσιών, όπως έγινε στο Ιράκ. Όλα αυτά ε, δείχνουν πρόδειλα ότι υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερη δημοκρατία, λογοδοσία και διαφάνεια. Αυτές οι δύο πτυχές πρέπει να συνδυαστούν για να ελπίζουμε σε μια δικαι... κάποιο είδους δικαιοσύνη στο μέλλον. Ποιες είναι οι συστάσεις τώρα που θα ήθελα να εκφράσω, ε, να διατυπώσω για τη συζήτησή μας. Εάν δούμε την νομική προστασία των πληροφοριωτών ένα στοιχείο που ειδικά θα έπρεπε να ισχύσει για το Βασίλειο είναι ότι χρειάζεται Πραγματικός κοινοβουλευτικός έλεγχος, επί της ουσίας όμως. Δηλαδή να υπάρξει κοινοβουλευτική επιτροπή που να ασκεί εξουσία, να μην διορίζεται από τον Πρωθυπουργό όμως και να έχει συνολικά νομοθετικές αρμοδιότητες ώστε να μπορεί να προστατεύσει τους πληροφοριοδότες, να έχουν και μια νομική οδό που να καταφύγουν. Και όχι να εκτίθενται απλώς Επίσης, η Επιτροπή αυτή του Κοινοβουλίου θα πρέπει να χαίρει τη εμπιστοσύνη των πληροφοριωτών, να ξέρουν ότι θα έχουν αποτελεσματική και επί της πράξης ε, διερεύνηση των κατηγοριών που μπορεί να εκφράσουν. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνεται ολοκληρωμένη έρευνα με πληροφορίες που συλλέγονται και από τις δύο πλευράς, με αντιπαραβολή και στοιχεία για ενδεχόμενα δικήματα που θα πρέπει να τιμωρούνται εφόσον διαλευκανθούν. Επίσης θα πρότεινα ειδικά στο Ηνωμένο Βασίλειο να υπάρξει νομικός ορισμός του τι αποτελεί η εθνική ασφάλεια, διότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στην νομοθεσία μας. Και θα πρέπει να προστατεύσουμε την ε, εθνική ασφάλεια προφανώ, να τη συνδυάσουμε με τα εθνικά συμφέροντα. Αυτό δεν σημαίνει όμω ότι πρέπει να, το, να κλείνουμε τα στόματα των πληροφοριδιωτών εφόσον ε, καταγγέλουν παράνομε ενέργειε. Υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Χρειάζεται λοιπόν νομικό ορισμό και μια κοινή κατανόηση ότι για να προστατευτεί η εθνική ασφάλεια πρέπει να προστατεύεται και ακαιρεότητα και η μελλοντική ύπαρξη των εθνικών κρατών. Αυτό λοιπόν που θέλουμε δεν είναι να βγούμε στους δρόμους, αλλά σίγουρα όχι να διακινδυνεύει και η εθνική ασφάλεια των, ενός κράτους με την παραβίαση του δυτικού βίου των πολιτών. Επίσης, η έκθεση Έσελον, εδώ και, μια, εδώ και μια δεκαετία, πρέπει να την αναθεωρήσουμε. Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία τότε για την Ευρώπη, για να δημιουργήσει τις δικές της υποδομές επικοινωνίας, να ξεφύγει από την ε, ε, πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ και τη Γερμανία. Και να υπάρξει πραγματική αρρωγή σε όσου τη χρειάζονται. Επίση, να βεβαιωθούμε ότι οι ΗΠΑ ε, συμμορφώνονται με την Ευρωπαϊκή Χάρτα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Πολύ σύντομα, για να ολοκληρώσω ναι. κιόλα, χρειαζόμαστε πολιτικέ και για την τεχνολογία, για τεχνολογικά μέσα, ώστε να μπορούμε να προστατευτούμε ένα, εάν ένα κράτο θέλει να παραβιάσει την ιδιωτική μα ζωή. Λόγου χάρη, εάν δεν μπορούμε να προστατευτούμε στο δίκτυο τηλεπικοινωνιών, τότε θα πρέπει ως μεμονωμένοι πολίτες να μπορούμε να λάβουμε κάποια μέτρα. Να ξεφύγουμε από τα software που ελέγχουν οι εταιρείε των Ηνωμένων Πολιτειών και ε, κατ' επέκταση ελέγχουν και τη ζωή μας. Γιατί τα κάναμε όλα αυτά ω πληροφοριώτε όμω, Γιατί χρειαζόμαστε ελεύθερα μέσα μαζική ενημέρωση, ελεύθερο διαδίκτυο. Αυτό δεν το έχουμε. Εάν δεν μπορεί κανεί να γράψει, να μιλήσει, να συζητήσει και να ξέρει ότι ο ιδιωτικό του βίο γίνεται σεβαστό, η ιδιωτική του σφαίρα γίνεται σεβαστή, τότε πού πηγαίνει η Δύση. Ε, η βασική κοινωνική λειτουργία τη ιδιωτικότητα τη επικοινωνία μα δεν είναι απλώ για να μπορούμε να λέμε ανοησίε και να περνάμε την ώρα μα. Όταν κανείς έχει την αίσθηση ότι παρακολουθείται συνεχώς, κάπου βέβαια προς αυτό τίνει. Όμως η ιδιωτικότητα, η ιδιωτική σφαίρα, οι ιδιωτικές συνομιλίες είναι το θεμέλιο και η ασπίδα κατά των παρεμβατικών ε, κρατών που παρακολουθούν τους πολίτες τους και γίνονται τυραννικά. Είδαμε τι έγινε με την Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα. Εδώ το πολιτικό σύστημα υπονομεύει το μέλλον των πολιτών αντί να προστατεύει και να διασφαλίζει την ιδιωτική τους σφαίρα. Ω τελικό λοιπόν σχόλιο θα ήθελα να πω ότι αν δεν υπάρχει ισορροπία μεταξύ ιδιωτική σφαίρα και ε, ε, ασφάλεια, αυτό που χρησιμοποιούν ω επιχείρημα οι μυστικέ υπηρεσίε, τότε υπάρχει πρόβλημα. Αυτή την ισορροπία πρέπει να εξεύρουμε μεταξύ ιδιωτικότητα και ασφάλεια. Και νομίζω ότι αντί για διχοτόμηση και αντιπαραβολή των δύο θεμάτων, πρέπει να αποφασίσουμε ότι και τα δύο τα χρειαζόμαστε και πρέπει να προστατεύονται και να συνδυάζονται. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι τώρα μπορούμε να θέσουμε τις ερωτήσεις στην κυρία Μάρσον, στον κύριο Drake, όπως και προηγουμένως. Θα ακολουθηθεί η διαδικασία. Είμαστε όμως πολύ, πολύ καθυστερημένοι. Θα ήθελα να πω στον εισηγητή ότι τα 10 λεπτά που έχετε επισήμως θα περιοριστούν σε ένα. Γλιτώσαμε 10 λεπτά, ωραία. Και θα ήθελα να σας προετοιμάσω, εσάς που θα πάρετε το λόγο κατόπιν, να είστε πιο σύντομοι από ό,τι αρχικά είχατε σκεφτεί να είστε. Γιατί πραγματικά έχουμε την υποχρέωση να τελειώσουμε στις 6.30 λόγω των διερμηνέων. Κύριε Μωράης, ναι, δεν θα κάνω τα συμπεράσματα δεν θα σας τα παρουσιάσω όπως ήθελα, αλλά πραγματικά όλες αυτές οι παρουσιάσεις ήταν εξαιρετικά χρήσιμες. Αυτό που τελικά πρέπει να κάνουμε στην έκθεση είναι να καταλάβουμε και ε, αν θέλετε από ιδεολογικής φιλοσοφικής απόψεως αλλά και στην πράξη τι αντιμετωπίζουν αυτοί οι whistleblowers, αυτοί οι άνθρωποι που προειδοποιούν αποκαλύπτοντας πληροφορίες. Γιατί ουσιαστικά πρέπει να τους δώσουμε κάποια στοιχεία και πρέπει εμάς να μας εξηγήσετε ακριβώς πώς έχει η κατάσταση όσον αφορά τις δυνατότητες που έχουν σε σχέση με τις Αμερικανικές αρχές. Πώς παραδείγματο κάποιον που εργάζεται στην NSA και βλέπει κάτι το οποίο δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Οποιουσδήποτε λοιπόν που θέλει να προειδοποιήσει και να αποκαλύψει ορισμένα πράγματα, ποια είναι η θέση του. Και το ίδιο αυτό θα ήθελα να αναρωτηθώ και για την Ευρώπη. Εγώ γνωρίζω τι γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στην δική μου χώρα δεν υπάρχει θέμα γραπτού συντάγματος, αλλά δεν αλλάζει τίποτα, καθότι δεν τηρούνται οι διαδικασίες όπως έχουν θεσπιστεί. Το ένα κράτος μέλος λοιπόν μετά το άλλο θα πρέπει να εξετάσουμε τις δυνατότητες, γιατί εδώ παραδείγματο χάρη διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει κοινοβουλευτικός έλεγχος. Δεν υπάρχει αρκετή και ικανοποιητική προστασία. Ποια θα ήταν λοιπόν η δική σας σύσταση όσον αφορά την ενίσχυση αυτής της προστασίας αυτών που θέλουν να προειδοποιήσουν. Σας παρακαλώ πολύ λέει η Πρόεδρος, μην ξεπεράσετε τα δύο λεπτά. Μπορείτε όμως να μιλήσετε και πιο λίγο από δύο λεπτά. Φώστην, θα μιλήσω γερμανικά πάλι. Βάλτε τα ακουστικά σας. Προσπαθούμε όλοι να βρούμε την ισορροπία μεταξύ της ασφάλειας, της προστασίας, της ιδιωτικής σφαίρας και ζωής. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, αυτή η εκτενής, η μαζική παρακολούθηση μας οδήγησε σε στοιχεία τα οποία τελικά συλλέγονται αδιάκριτα και εν μέρη χρησιμοποιούνται χωρίς τις άδειες οι οποίες προαπαιτούνται. Αυτά τα στοιχεία, αυτά τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία μπορούν να μπουν στην κατηγορία του πολιτι... της πολιτικής κατασκοπίας, αλλά και της επιστημονικής και βιομηχανικής κατασκοπίας. Κατά πόσο και ποιο είναι το ποσοστό αυτών των δραστηριοτήτων που σας φαίνεται επικίνδυνο Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ και παίρνετε το λόγο. Για μας αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η πρώτη μου ερώτηση είναι η εξής. Ποια είναι η κλίμακα, όπως εσείς την αξιολογείτε, για την μη αποκάλυψη στοιχείων. Ο κύριος Βίμπε αλλά και εσείς κύριε Ντρέικ ήσασταν ε, στην NSA. Ε, Εργαστήκατε σε αυτήν την ε, υπηρεσία. Ξέρω λοιπόν ότι μπορείτε να μας εξηγήσετε ακριβώς το τι συμβαίνει εκ των έσω. Επίσης μιλήσατε και για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Πώς αυτό μπορεί να γίνει αποτελεσματικά. Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν έχετε λοιπόν να μας δώσετε κάποιες ε, ιδέες, κάποιες συστάσεις, αλλά μιλήσατε και για κάτι άλλο που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, τι μπορούμε να κάνουμε όσον αφορά την προστασία των δεδομένων και την προστασία αυτών που θέλουν να ξεκινήσουν την αποκάλυψη στοιχείων και να προειδοποιήσουν την κοινή γνώμη. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν πραγματικά να σας ευχαριστήσω που είστε σήμερα εδώ. Είναι πολύ σημαντικό για μας. Και έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι πώς μπορεί να γίνει αυτός ο κοινοβουλευτικός έλεγχος. Μιλήσατε για αυτόν, ε, κυρία και θα ήθελα να μας πείτε σε εθνικό επίπεδο τι μπορούμε να κάνουμε για να είναι αποτελεσματικός αυτός ο κοινοβουλευτικός έλεγχος. Και δεύτερον, τι μπορούμε να κάνουμε νομοθετικά για να ενισχυθεί η προστασία αυτών των whistleblowers. Διάβασα κάποια από αυτά που λέτε. Διάβασα τις συστάσεις σας. Ναι, τα βρίσκω πολύ χρήσιμα αυτά που λέτε, αλλά συγκεκριμένα για την ε, νομοθετική προστασία των whistleblowers. Τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να αλλάξει ουσιαστικά η κατάσταση σημερινή. Ε, um, Ευχαριστώ κυρία Ernst. Η τελευταία ερώτηση είναι δική μου, είμαι σκιώδης της ε, Άλτε των Φιλελεύθερων. Μιλήσατε για πόλεμο κατά των whistleblowers. Εγώ θα έλεγα πόλεμος κατά της δημοκρατίας. Γιατί αν δεν υπάρχει διαφάνεια, δεν υπάρχουν μηχανισμοί διαφάνειας οι οποίοι να λειτουργούν. Οι whistleblowers είναι οι μόνοι που έχουν παραμείνει ζωντανοί για να μάθουμε το τι συμβαίνει. Όσο τρελό και αν φαίνεται, Έχουμε την εντύπωση ότι οι μυστικές υπηρεσίες λειτουργούν κρυφά και ανεξέλεγκτα, τελείως ανεξέλεγκτα. Οι ερωτήσεις μου λοιπόν είναι οι εξής. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι εδώ, σε αυτό το κοινοβούλιο, οι οποίοι αποκαλούν τους whistleblowers εγκληματίες, οι οποίοι θα πρέπει να καταδικαστούν. Δεν είναι όμως σήμερα εδώ όλοι αυτοί. Θεώρησαν ότι δεν ήταν χρήσιμο να έρθουν. Και καταλαβαίνετε ότι όλοι αυτοί πρεσβεύουν ότι αυτά τα συστήματα εκτεταμένης ηλεκτρονικής παρακολούθησης υπάρχουν για να μας προστατεύσουν. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν να αντικρούσουμε αυτές τις ιδέες και πώς είναι δυνατόν το Κογκρέσο και άλλα νομοθετικά σώματα, άλλα κοινοβούλια να δέχονται, ενώ είμαστε δημοκρατικά πολιτεύματα, να αφήνουν αυτές τις υπηρεσίες να λειτουργούν ανεξέλεγκτες και γιατί τα κοινοβούλια δεν κάνουν το καθήκον τους και δεν ασκούν κοινοβουλευτικό έλεγχο σε αυτές τις μυστικές υπηρεσίες. Κύριε Drake, έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Όσον αφορά την προστασία των πληροφοριοδοτών, των whistleblowers, να σας πω αυτά τα οποία, ε, ε, να σας παραπέμψω σε αυτά που θα πούν οι προηγούμενοι, εγώ να σας πω ότι ήμουν τελείως εκτοθυμένος, οποιαδήποτε νομοθεσία δεν ε, ε, λήφθη υπόψη και δεν είχα και καμία δυνατότητα να προσφύγω στο δικαστήριο ή να εφεσιβάλω κάποια απόφαση. Έχω πολλά να πω, αλλά δεν θα τα πω για το θέμα αυτό. Όσον αφορά τώρα το θέμα της διατήρησης των δεδομένων και το κράτος δικαίου, βάσει Αμερικανικής νομοθεσίας και του τετάρτου άρθρου του συντάγματος ε, πρέπει να υπάρχει πιθανή αιτία Και δεν έχει σημασία. Αυτό που συνέβη είναι ότι έγιναν όλα με πάσα μυστικότητα και ε, αποφασίστηκε βάση του θέματος να κατασχεθούν πρώτα τα στοιχεία και να εκδώσουν τα εντάλματα αργότερα. Το πού έγιναν ε, οι έρευνες και πού βρίσκονταν αυτά τα στοιχεία ε, που θέλουμε να κατασχέσουμε έχει μεγάλη σημασία. Τώρα, για τη βιομηχανική, ε, χρηματοοικονομική και άλλη μορφή κατασκοπίας νομίζω ότι όλα τα στοιχεία τα οποία αποκαλύπτονται στον τύπο αποτελούν πολύ σημαντικές αποδείξεις που δείχνουν ότι χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες αυτές ε, ανάλογα με την ε, πρόσβαση που έχουμε και για άλλους λόγους. Αυτά ήταν ένα από τα μεγάλα καθόδη ζητήματα Υποτίθεται ότι υπάρχουν ισχυρισμοί ότι χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες αυτές για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή άλλης εγκληματικής δραστηριότητας, αλλά όταν έχει κάποιος ε, τέτοιες πληροφορίες γιατί άλλο θα μπορούσε να τις χρησιμοποιήσει. Εγώ θα μπορούσα να προσθέσω εδώ και για πολιτικούς λόγους. Όσον αφορά τώρα την κλίμακα, εγώ έμεινα μέχρι το 2008 στην NSA ε, γνώριζα για το πρόγραμμα ε, Πρίσμα, το οποίο το είχε δημιουργήσει η Αμερικανική κυβέρνηση για να δει τι είχε αν γίνει τα προηγούμενα δύο χρόνια σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα, αλλά η μυστική ερμηνεία ήταν να δίνεται πρόσβαση παρανόμως για όλα όσα γίνονταν τα προηγούμενα 4-5 χρόνια. Υπήρχε πρόσβαση χωρίς καμία έγκριση σε ε, ε, στοιχεία τα οποία δεν θα έπρεπε να λαμβάνονται και υπήρξε και μια ρήτρα το 2006 για να δοθεί πρόσβαση σε πολύ μεγάλο αριθμό δεδομένων και σε τηλεφωνικά μητρώα ε, από τις βασικές επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών. Για μένα όλα όσα αποκάλυψε λοιπόν ο ο Σνόντεν απλώς αποδεικνύουν πόσο μεγάλης κλίμακας είναι η παρακολούθηση πλέον. Όσον αφορά την εποπτεία και τον έλεγχο, ε, εμείς αστείευουμε βέβαια εδώ, αλλά έχουμε επιτροπές οι οποίες δεν κάνουν κανέναν έλεγχο. Είναι όλοι μπλεγμένοι, ελάχιστοι γερουσιαστές ή βουλευτές μπορούν πραγματικά να πούν ότι είναι αθώοι και το άλλο καθόδε ζήτημα είναι ότι διακυβεύονται πάρα πολύ μεγάλα κονδύλια εδώ, επιχειρήσεις, ιδιωτικές επιχειρήσεις ε, σε συνδυασμό με την κυβέρνηση ε, και πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη βιομηχανία η παρακολούθηση. Δεν έχουμε μόνο επιχειρήσεις που παρακολουθούν στοιχεία και τα πολλούν, αλλά γίνεται παρακολούθηση για να δίνονται πληροφορίες και στις κυβερνήσεις και πραγματικά ε, πιστέψτε με δεν γίνονται σε καμία περίπτωση νομίμως αυτές οι διαδικασίες. στην ουσία αυτό το οποίο διακυβεύεται εδώ είναι τα ίδια τα θεμέλια της δημοκρατίας και κάτι πρέπει να γίνει. Όταν υπάρχει μυστική νομοθεσία, μυστικά στοιχεία, μυστικές απόψεις, ε, τότε η ίδια η δημοκρατία παραλύει και φυσικά ε, η ιστορία μας δείχνει και η ιστορία λειτουργεί χρησμοδός για το μέλλον μας δείχνει ότι χρειαζόμαστε στοιχεία για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε την κυριαρχία ε, των κρατών αλλά κυρίως ε, και την αξιοπρέπεια και την, το ίδιο το άτομο. Εδώ αντικαθίσταται το κράτος δικαίου και αυτός είναι ο μεγάλος καταλήτης από μορφές απολυτερχικής μεταχείρισης και εγώ το είδα αυτό, η διεισόμαση τα τελευταία 6 χρόνια και το δείχνει και η ιστορία ε, τι ακριβώς γίνεται όταν ζει κάποιος σε απολυταρχικά και φασιστικά καθεστώτα. Ευχαριστώ κυρία Προσπαθήσω να είμαι πολύ πολύ σύντομη. Φαίνεται ότι πολλά θέματα προκύπτουν σε πολλές από τις ερωτήσεις και επαναλαμβάνονται. Η προστασία των whistleblowers. Τι πρέπει να κάνουμε για να προστατεύσουμε στο μέλλον ε, ανθρώπους που θα αποφασίσουν να αποκαλύψουν κάποιες πληροφορίες και ιδιαίτερα στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Σαφώς και εδώ χρειάζεται για όλες τις χώρες μου τις χώρες μας στην Ευρώπη μία πρώτη έρευνα κοινοβουλευτική η οποία να επιτρέπει να εντοπιστούν και να τεθούν υπό αυτά τα άτομα. Η συγκεκριμένη προστασία των whistleblowers, παραδείγματο χάρη στο Ηνωμένο Βασίλειο, ήδη από το 1998 υπάρχει μέσω του Disclosure Act η δυνατότητα μια τέτοια προστασίας. Βεβαίως, βεβαίως αποκλείονται από αυτές τις περιπτώσεις οι μυστικέ υπηρεσίες, οι υπηρεσίες πληροφοριών. Μήπω θα πρέπει να τους ε, ενσωματώσουμε. Αυτό θα ήταν μια περίπτωση. Επίσης, ακόμα και οι υπηρεσίες κατασκοπια υπάρχουν τριών ειδών, αν θέλετε, ε, διαβαθμίσει ε, πληροφοριών. Υπάρχουν ε, οι ευαίσθητες πληροφορίες, οι ευαίσθητες ε, τεχνικές πληροφορίες, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε, παραδείγματο χάρη, να χρησιμοποιήσουμε κάποιες πληροφορίες που προκύπτουν από τηλεφωνικές συνδιαλέξεις σε μία υπόθεση στο δικαστήριο. Καταλαβαίνετε ότι σήμερα με τα κινητά τηλέφωνα και τις δυνατότητες παρακολούθησης που υπάρχουν τη νέα τεχνολογία, αυτό είναι γελίο. Γι' αυτό και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση των τεχνικών δυνατοτήτων και φυσικά να επιληφθούν τα κοινοβούλια και οι κοινοβουλευτικές ε, επιτροπές όλων αυτών των διαδικασιών και ήδη από το Ηνωμένο Βασίλειο στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 1998 και από το συγκεκριμένο αυτό νομοθετικό κείμενο το οποίο επιτρέπει κάποιες αποκαλύψεις έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ τα πράγματα που θα πρέπει και αυτό να αναθεωρηθεί. Τώρα, αυτό ήταν σε εθνικό επίπεδο, τι πρέπει να κάνει η κάθε ε, χώρα, το κάθε κοινοβούλιο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα προσφυγής κάποιου whistleblower από τη στιγμή που δεν θα μπορέσει να τύχει της ε, κατάλληλης προστασίας στη χώρα του, σε εθνικό επίπεδο, σε κάποιο όργανο, σε κάποιο θεσμό, κάποια επιτροπή, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία να μπορεί να επιληφθεί της υπόθεσής του. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε σήμερα είναι ότι σήμερα από τη μία έχουμε την ε, ελευθερία λόγου, τον τύπο, τα διαδίκτυα, τα ηλεκτρονικά δίκτυα και την επικοινωνία και από την άλλη τα τελευταία 10-15 χρόνια έχουμε μία ενδυνάμωση της ασφάλειας και μία παρακολούθηση της προσωπικής μας ζωής, μία παρακολούθηση του τι κάνουμε, με ποιον συναντιόμαστε, με ποιον επικοινωνούμε, έτσι ώστε να υπάρξει μία ενίσχυση της ασφάλειας. Αυτό που εμείς πρέπει εδώ να πούμε συλλογικά και εκτεταμένα είναι ότι κάπου θα πρέπει να σταματήσει και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση χωρίς να αρνηθούμε βεβαίως το διαδίκτυο και τις δυνατότητες που μας παρέχει να προστατεύσουμε την προσωπική μας ζωή και ιδιαίτερα αυτό μπορεί να το κάνει στην Ευρώπη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μου είπατε ότι κάποιοι εδώ θεωρούν ότι καλά κάνουν οι μυστικές υπηρεσίες και ορθώς υπάρχει και μας προστατεύει αυτό το σύστημα παρακολουθήσης. Κρίμα που δεν είναι σήμερα εδώ, γιατί θα ήθελα να τους ακούσω, γιατί πραγματικά με ενδιαφέρει ιδιαίτερα να ε, δω τι επιχειρήματα έχουν αυτοί οι άνθρωποι όταν τους ε, ενημερώνουμε για το τι σημαντικά στοιχεία μας αποκάλυψαν αυτοί οι whistleblowers, πόσες ζωές σώθηκαν χάρη σε αυτούς. Εν πάση περιπτώσει, σε καμία περίπτωση εγώ δεν θέλω να προστατεύσουμε κάθε είδους ε, πληροφορίες, είτε πληροφορίες που ανήκουν στην κατασκοπία, παράνομη κατασκοπία, ε, είτε άλλου είδους τέτοιες αποκαλύψεις. Όσον αφορά τώρα το 1996 και την ε, περίπτωση αυτών οι οποίοι ανήκαν στον MI6, Γνωρίζουμε σήμερα ότι ήταν μπλεγμένη σε εγκληματική οργάνωση, ότι βρισκόταν πολύ κοντά στην Αλκάιντα. Βεβαίως, ξέρετε ότι από την άλλη πλευρά έχουμε αποκαλύψεις. Θυμάστε την περίπτωση του ελικόπτερου που πυροβόλησε παιδιά σήμερα ο πιλότος αυτού του ελικόπτερου δεν είναι στη φυλακή. Συνεχίζει να είναι ελεύθερος γιατί εργαζόταν για μια κρατική υπηρεσία. Νομίζω ότι αυτό ήταν ε, για να επικροτηθεί το έργο σας. Έχουμε πολλά κοινά, εσείς στη δουλειά σας και εμείς στην Επιτροπή μας, οπότε τώρα πολύ γρήγορα θα περάσουμε στο τελευταίο μας τμήμα της ε, συζήτησης. Όχι, έχουμε μια τελευταία ερώτηση, κυρία Μορβάη. Αλλά η κυρία Μορβάη θα είστε πάρα πολύ σύντομη, γιατί ο κύριος Μπρόντς είχε ζητήσει το λόγο πρώτος. η μαρτυρία του κυρίου Ντρέικ ότι το 2011 ήταν ε, αυτό που ξεκίνησε τη χινοστιβάδα, ας το πούμε έτσι. Αυτό που οδήγησε σε αυτές τις φρικαλαιότητες ήταν ότι δόθηκε το πρόσχημα για την παρακολουθήση. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι οι εργαζόμενοι της NSA και άλλων πρακτορείων επιθυμούν ε, επιθυμούσαν την παρακολούθηση πριν βρουν το ανάλογο πρόσχημα. Διότι ξέρετε ότι δεχτήκατε διώξεις, διότι αποκαλύπτοντας τις ενέργειες της NSA. Είδατε να χρησιμοποιούνται για ευρύτερους πολιτικούς ε, σκοπούς που να μην έχουν σχέση με την παρακολούθηση αυτή καθεαυτή. Η κυρία Μάκεν μας είπε πολλά για τη χρήση των δεδομένων. Πώς πιστεύετε ότι χρησιμοποιούνται στην περίπτωση των Υπουργείων και των δημοσιογράφων Ο κύριος Χέικ έδειξε προθυμένη να συνεννοηθεί με τις μυστικές υπηρεσίες. Μπορώ να ρωτήσω λοιπόν τελείως επιφυλακτικά. Αυτό το έκανε αυτόβουλα, διότι κάποιες από τις δράσεις του μπορεί να θεωρηθούν το λιγότερο αμφισβητούμενες, αμφισβητήσιμες μάλλον. Για τις μυστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων βλέπουμε ότι χρησιμοποιούν τις πληροφορίες για πολλούς σκοπούς ασχέτως ασφάλειας. Υπάρχει γραφειοκρατικό ενδιαφέρον να προστατευτούν θερμικά συμφέροντα των υπηρεσιών ή υπάρχει μια ευρύτερη ατζέντα και ποιανού είναι αυτή η ατζέντα. Και επίσης, τι θα γίνει εάν κάποιος ε, τύραννος έρθει στην εξουσία. Η κυβέρνηση μπορεί να χρησιμοποιήσει και να παρακάμψει κάθε μέσο πολιτικούς, ε, πολιτικής πυθός. Και αν θέλει να λάβει κάποιο μέρος, απλώς θα το κάνει. Ευχαριστούμε. Κυρία Μόρβα, παρακαλώ να είστε όσο το δυνατόν πιο σύντομη. Δεν ξέρω γιατί εγώ πρέπει να είμαι σύντομη και συντομότερη από τους ε, υπόλοιπους. Ε, μα δεν υπάρχουν και άλλα μέλη τη Επιτροπή εδώ και δεν βλέπω γιατί εγώ πρέπει να κάνω έκουση, κυρία Πρόεδρε. Γιατί όλοι είχαν δύο λεπτά, πάντα Πρόεδρο. Όχι, όλοι είχαν δύο λεπτά και τόσο θέλω και εγώ. Τέλο πάντων, ο... μετά τι αποκαλύψεις, ο ήλιο συνεχίζει να ανατέλει καθημερινά. Το ίδιο και μετά τον ε, κύριο Σνόντεν. Αλλά πιο συγκεκριμένα αναφέρατε, κυρία Ντρέικ, την στάζη και τους πράκτορες της ΤΑΖΗ καθώς και το έργο τους για τη συλλογή δεδομένων. Σε αυτή τη χρονική περίοδο δεν ξέρω ποιοι συμφωνούν. Ο εθνικοσοσιαλισμός, ο κομμουνισμός ήταν ένα είδος δημοκρατικ... δικτατορίας. Και αυτά ήταν τα μέσα της δικτατορίας για να πετύχουν τους σκοπούς τους. Ε, εδώ ε, υπάρχει πολιτική αποδοχή στο σημείο αυτό, όμως μια δικτατορία βλέπετε να υπάρχει σήμερα. Είναι μια τέτοια δήλωση λιγότερο πολιτικός ορθή. Δεν μπορούμε να μιλάμε για δικτατορία πλέον. Και ποιοι είναι οι δικτάτορες. Είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε. Είναι οι πολυεθνικές εταιρείες, οι τραπεζίτες που χέρι-χέρι διαπλέκονται με την πολιτική εξουσία. Βλέπουμε το 99% της εξουσίας να βρίσκεται στα χέρια λίγων. Είπατε ότι όλα ξεκίνησαν με την 11η Σεπτεμβρίου. Όμως, η ανάγκη για ευρύτερη παρακολούθηση ξεκίνησε τη στιγμή που συνέβη αυτό το γεγονός. Πώς εξηγείται αυτή την παράλληλη πορεία. Και γιατί να περνάμε όλες αυτές τις δυσκολίες και τα προκειμένου να σώσουμε τελικά την ελευθερία. Αυτός είναι ο μόνος στόχος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κύριε Ντρέικ, θέλετε να ξεκινήσετε. Να ξεκινήσω από το τέλος. Για όσα λέει το Σύνταγμα, ξεκίνησε πριν από μια 20 ετία ως πείραμα όλη αυτή η διαδικασία. Και για τις δύο πλευρές του Ατλαντικού όμως. Εγώ δεν πήρα όρκο μυστικότητας αλλά ούτε και να διαπράττω παράνομες πράξεις και να παραβιάζω την ακαιρεότητα της ιδιωτικής σφαίρας των πολιτών. Είναι θεμελιώδη σημασία στο γιατί άρχισα να αποκαλύπτω πληροφορίες. Κάτι που έκαναν κι άλλοι συναδελφοί μου άλλωστε. Διότι πέρασαν μια κρίση συνείδησης. Κρίση συνείδησης και αυτό το επέλεξα για το μέλλον. Όχι εγώ, άλλοι. Δεν μπορούσα να μένω απαθής και να βλέπω ο τρόπος ζωής μου να ε, υποβαθμίζεται ηθικώς κάτι που είχα αποφασίσει από μια 40 ετία. Τώρα αυτό που στάζει και αν υπάρχει δικτατορία. Ναι, είναι πολύ ισχυρά τα εταιρικά συμφέροντα, πολύ ε, πιεστικά τα πρωτόκολλα, αλλά με το είδο τεχνολογικών μέσων που διαθέτουμε. Δεν χρειάζεται και πολύ ένα κράτο παρακολούθησης να πετυχαίνει του σκοπού του. Μπορούν να βρουν ό,τι στοιχείο θέλουν για τον οποιονδήποτε να πάσα στιγμή. Και για το άλλο ερώτημα, για την NSA. Η NSA ε, εκτέθηκε στο διαδίκτυο, γιατί θεώρησε το διαδίκτυο είναι ελεύθερο και ανοιχτό για όλους. Αυτό βεβαίω άλλαξε δραματικά τα χρόνια πριν την 11η Σεπτεμβρίου. Να πω σύντομα ότι κατά την προεδρική μετάβαση του George Bush ε, στις αρχές του 2000 η δράση της NSA δημοσιευόταν στο ίντερνετ. Ήδη με το τέταρτο άρθρο του συντάγματο έψαχναν τρόπου βέβαια να γίνουν ακόμη πιο πιεστικοί στην παρακολούθησή του και προέκυψε 11 Σεπτεμβρίου. Κάτι μα λέει αυτό και μπορεί να υπάρξει και διασύνδεση μεταξύ των γεγονότων. αλλά νομίζω ότι συνολικά έχω απαντήσει λίγο πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μαξόν. Ενδιαφέρουσε ερωτήσεις και θα μπορούσα να απαντήσω με τις ώρες ε, στην καθεμιά, αλλά θα προσπαθήσω να τα συνοψίσω. Οι Βρετανοί πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι ε, είναι δεσμευμένοι από την ε, μυστικότητα που πρέπει να τηρούν. Ακόμα και αν υπουργό εσωτερικών ή εξωτερικών που είναι υπεύθυνοι για το MI5 και MI6 αντίστοιχα, δεν μπορούν να δουν τις πληροφορίες και τα αρχεία ε, που συγκεντρώνουν αυτές τις μυστικές υπηρεσίες. Δεν ξέρουν τι στοιχεία έχουν συγκεντρωθεί εναντίον του. Και μπορούμε να φανταστούμε ότι οι πολιτικοί μπορεί να έχουν τα μικρά του ένοχα μυστικά και ότι θα ήθελαν πολύ να τα απαλείψουν. Οι δημοσιογράφοι λένε ακριβώ το αντίθετο, ότι επειδή δεν ξέρουν τι θα γίνει ή τι μπορεί να υπάρχει εναντίον του, φοβούνται ακόμη περισσότερο. Και αυτό είναι και ο λόγο που η προηγούμενη κυβέρνηση των λιγοτικών ήθελε να ελέγξει την ε, ε, κοινότητα των μυστικών υπηρεσιών το αν ε, κοιτάζουν την, ε, και επηρεάζουν την ευρύτερη πολιτική διαδικασία. Ναι, αυτό συνέβη και με μυστικού ε, αστυνομικού, οι οποίοι ήθελαν να διαχωρίσουν το αστυνομικό του έργο από το καταστροπικό στι αρχέ τη δεκαετία του 1990. Και στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν υπάρχει ε, πρόβλημα μετακίνηση στο Βρετανικό δίκαιο από ένα δίκημα σε άλλο. Δηλαδή οι μυστικοί αστυνομικοί διερευνούσαν την ε, εξτρεμιστική δράση που η Βρετανική κυβέρνηση αυθαίρετα είχε θεωρήσει εξτρεμιστές ή ενδεχόμενου τρομοκράτε μόνο και μόνο επειδή είχαν καταλάβει ένα χώρο αγατήκητο στο κέντρο της πόλης και κατοικούσαν εκεί. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη ευθερεσία και αυτό είναι πραγματικός κίνδυνο για τη δημοκρατία τώρα. Γιατί ε, διτηρούν την εξουσία τους. Ε, είναι επειδή έτσι έχουν δουλειά. Υπήρχε το MI5, είχαν ελεύθερο χρόνο όλοι αυτές τις μυστικές υπηρεσίες, δεν υπήρχαν προβλήματα, τους βρήκαν την ε, τρομοκρατία, την Αλκάιντα. Αλλά ποιε είναι οι πραγματικέ απειλέ στην εθνική μα ασφάλεια, στην εθνική μα ε, ακαιρεότητα. Πώ μπορούμε από αυτέ να προστατευτούμε καλύτερα. Αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα. Αν οι μαε 5 ήταν ε, σωστοί ε, ή δεν έκαναν καλά τη δουλειά του, θα πρέπει απλώ να φύγουν και να βρεθούν άλλοι αξιότεροι. Αυτό είναι η λύση και πρέπει να εργάζονται και υπό τους όρους από του οποίους εργάζεται η αστυνομία. Η MI5 ε, παρακολουθεί τρομοκρατικές ομάδες, οι ομάδες που έτσι έχουν θεωρηθεί, κάνοντας αστυνομικό έργο και χωρίς αυτό τι έχει ζητηθεί. Και για το αν ζούμε σε μια δικτατορία. Να σα πω, θα μιλήσω με το παράθυμα του Λένιν για το τι είναι ο φασισμό και ποια είναι η πραγματική ουσία του φασισμού. Είναι η διαπλοκή του κράτου με του επιχειρηματίε. Οι ομάδες πίεσης μπορεί να επηρεάσουν την καθοριστική νομοθεσία ακόμη και στα υψηλότερα θεσμικά όργανα, όπως η περσινή πράξη για την ε, καταπολέμηση της αντιδημοκρατικής εταιρική δράσης. Οι ακτιβιστές άσκησαν πιέσεις, αναμενόταν υπογραφή και φυσικά αυτό αποτελεί παρέμβαση στα πράγματα του κράτους. Και αυτό μας πάει πάλι στα στα, στις προειδοποιήσεις ε, της ιστορίας. Ο Eisenhower το 1946 προειδοποιούσε την, ε, για την παρέμβαση της βιομηχανίας στην ελευθερία του τύπου. Αυτό λοιπόν δείχνει πόσο περίπλοκο είναι το φαινόμενο και η διαπλοκή κράτους με μυστικές υπηρεσίες. Στον πόλεμο οι μυστικές υπηρεσίες, οι μυστικές πληροφορίες είναι κάτι που όντω οδηγεί σε μορφή συνεργασίας που δεν θα είχαμε φανταστεί και μάλιστα πολύ στενές. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Κλείνουμε τώρα αυτήν την, αυτό το τμήμα τη ε, συζήτησή μας. Θα περάσουμε στο τελευταίο τμήμα να καλέσω τώρα τους ομιλητές μας στο Προεδρείο και ζητώ συγγνώμη γιατί εσείς θα πρέπει να μιλήσετε πολύ σύντομα. Θα σα τους ε, συντομεύσουμε. Θα ζητήσω να μιλήσετε ο καθένα σα από 10 λεπτά και μετά θα έχουμε μόνο 10 λεπτά για ερωταπαντήσει. Θέλω να είσαστε τάχιστοι. Εάν μπορούν οι διερμηνείς να μας δώσουν και λίγα παραπάνω λεπτά επίσης, ώστε να παρατείνουμε κάπως τη συνεδρίαση. Αυτό θα μας βοηθούσε πολύ. Καλώς ορίσατε. Έχουμε δύο μιλητές από με κυβερνητικές οργανώσεις πολύ δραστήριες στον τομέα των πληροφοριοδοτών. Ο κύριος ε, Ραντέκ είναι ο πρώτος ε, ε, ομιλητής υπεύθυνο ε, για το πρόγραμμα κυβερνητικής λογοδοσίας ο οποίος έχει αναλάβει έξι προϋποθέσεις εκ των οποίων και ο ίδιος και ο Τζον Ντεβιτ Ντεβιτ, με συγχωρείτε ε, υπεύθυνο για τη Transparency International για θέματα πληροφοριωτών. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα κυρία Ρόντεκ να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που μου δίνει το λόγο. σε αυτήν την πάρα πολύ σημαντική ε, συνεδρίαση εδώ σήμερα και βεβαίως ελπίζω ότι μετά τις αποκαλύψεις του Edward Snowden θα χρησιμοποιηθούν όλες αυτές οι περιπτώσεις για να ενδυναμώσουμε την προστασία αυτών που τολμούν να αποκαλύψουν τόσο σημαντικές πληροφορίες και ότι πραγματικά το κοινό θα μπορεί να μην βασίζεται μόνο στις ε, πληροφορίες ε, που του αποκαλύπτουν, οι οποίες δεν είναι ποτέ πλήρης, οι διάφοροι εργαζόμενοι στις κρατικές υπηρεσίες και στις ε, υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ το πρόγραμμα για την εθνική προστασία, προστασία των πολιτικών ελευθεριών, συμπεριλαμβάνει πολλές ε, περιπτώσεις σαν και αυτή του Edward Snowden και σαν υπεύθυνη για την προάσπιση αυτών των επιθέσεων λαμβάνουμε υπόψη μας όλες τις υποθέσεις από το πρώτο στάδιο όταν υπάρχει κατάχρηση ή παράνομη δράση. Το 2010 για πρώτη φορά γνώρισα για πρώτη φορά την υπηρεσία των ε, μυστικών υπηρεσιών και την NSA. Ακούσατε τον William, Drake και ήταν ο πρώτος με τον οποίο είχα ε, επαφή από αυτήν την ε, υπηρεσία. Μετά την 11η ε, Σεπτεμβρίου έμαθα και κατάφερα να γνωρίσω εκ των έσω ότι πραγματικά η κυβέρνηση Μπούς είχε αποφασίσει να είναι πάρα πολύ σκληρή με όλους αυτούς οι οποίοι έμπαιναν στην κατηγορία των whistleblowers και αποφάσιζαν να αποκαλύψουν σημαντικές πληροφορίες για να διαφυλάξουν το κοινό καλό. Αυτό έφτανε μέχρι και να κινδυνεύσει η ζωή τους. Όταν ανέλαβε ο πρόεδρος Ομπάμα και συνειδητοποίησα ότι η ποινικοποίηση της αποκάλυψης της αλήθειας ξεπέρασε ένα ακόμα στάδιο, συνειδητοποίησα ότι είχαμε περάσει από την άλλη όχθη ε, του ποταμού και ότι πραγματικά δεν υπήρχε περίπτωση να προστατεύσει κανείς τους whistleblowers από τη στιγμή που είδαμε ότι άρχισαν να καταδικάζονται σαν κατάσκοποι. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι μετά από ένα χρόνο διακυβέρνησης Ομπάμα περισσότεροι άνθρωποι μπήκαν στην κατηγορία της κατασκοπίας, ενώ ήταν whistleblowers, άνθρωποι που ήθελαν να αποκαλύψουν σημαντικές πληροφορίες στο κοινό. Είδαμε ότι πολλές οργανώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν σήμερα με την αποκάλυψη πληροφοριών να στηρίξουν και να προστατεύσουν τους whistleblowers και ο Julian Assange και ο ίδιος όπως ξέρετε βρίσκεται υπό μια τέτοια διαδικασία και ο οποίος ε, φυλακίστηκε οικειοθελώς στην ε, πρεσβεία του Ισημερινού στη Μεγάλη Βρετανία. Έχει ξεκινήσει μια ολόκληρη διαδικασία συλλογής στοιχείων για όλες αυτές τις διαδικασίες Γνωρίζουμε σήμερα ότι δημοσιογράφοι αλλά και άλλοι οι οποίοι εργάζονται για την προάσπιση των δικαιωμάτων των whistleblowers έχουν συλλέξει στοιχεία όσον αφορά την προστασία τους με σκοπό να αποκαλύψουμε όλες αυτές τις παράνομες διαδικασίες οι οποίες συμπεριλαμβάνουν βεβαίως παράνομη παρακολούθηση, σε απαράδεκτο βαθμό της προσωπικής ζωής ε, ιδιωτών, αλλά και βασανιστήρια και εγκλήματα πολέμου. Το ερώτημα είναι εδώ αν θα ανοίξει ένας πόλεμος κατά αυτών των υπηρεσιών και ξέρουμε ότι οι περισσότεροι οι οποίοι βρίσκονται και εργάζονται σε αυτές τις υπηρεσίες, με αυτές τις παράνομες πρακτικές, καλούνται να επιλέξουν μεταξύ της ελευθερίας συνείδησης και της ε, εργασίας τους, τη θέση τους στην κοινωνία. Σήμερα οι whistleblowers καλούνται να επιλέξουν μεταξύ της ζωής τους και της τυφλής υπακοής στην υπηρεσία. Οι αποκαλύψεις πολλές φορές δεν έχουν σαν αντικείμενο την παρακολούθηση, την ηλεκτρονική παρακολούθηση, αλλά και την προσαγωγή τους και αυτό βεβαίως καθαρά και μόνο διότι έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Υπάρχουν πολλοί Αμερικάνοι πολίτες οι οποίοι σήμερα παρακολουθούνται. Δημοσιογράφοι, πολιτικοί, απλοί πολίτες, επαγγελματίες, γιατί παρακολούνται. Διότι ζούμε σε έναν κόσμο ηλεκτρονικό που η τεχνολογία σήμερα πάρα πολύ εύκολα επιτρέπει την ηλεκτρονική παρακολούθηση και την συλλογή στοιχείων. Και βεβαίως δεν χρειάζεται κανείς να εργάζεται στον κυβερνοχώρο και να είναι ειδικό του κυβερνοχώρου για να μπορέσει να κατασκοπεύσει, να παρακολουθήσει παράνομα αθώους πολίτες. Σήμερα οι Ηνωμένε Πολιτείε από την 11η Σεπτεμβρίου δαπανούν δισεκατομμύρια για την ηλεκτρονική παρακολούθηση των πολιτών. Και ένας άνθρωπος κατάφερε να αποκαλύψει στοιχεία που αφορούν την πιο ισχυρή μυστική υπηρεσία στον κόσμο. Και με τις συγκλονιστικές αυτές αποκαλύψεις μπόρεσαν δημοσιογράφοι παντού στον κόσμο να δημοσιεύσουν τις πληροφορίες του Edward Snowden, ο οποίος πραγματικά κινδύνεψε την ίδια του τη ζωή, διακινδύνευσε την ίδια του τη ζωή, αποκαλύπτοντας στην κοινή γνώμη αυτές τις πληροφορίες και τις παράνομες διαδικασίες, οι οποίες συνεχιζόταν εδώ και χρόνια. Η προστασία της προσωπικής ζωής, των προσωπικών δεδομένων και η δυνατότητα να διαδοθούν αυτές οι περιπτώσεις είναι κάτι που θα πρέπει όλοι να το στηρίξουμε και ελπίζω ότι αυτές οι έρευνες θα συνεχιστούν καθότι έχουμε νέα στοιχεία που αποκαλύπτονται. Όπως είπε ο πρόεδρος Λίκων πριν από 150 χρόνια, χειρότερα από τους προδότες είναι αυτοί οι οποίοι κρύπτονται πίσω από την ειρήνη, από την προστασία των πολιτών και συνεχίζουν να οδηγούν τον λαό τους στην λάσπη. Θεωρούμε πραγματικά ότι η δημιουργία ενός κράτους παρακολούθησης, παράνομης παρακολούθησης, είναι κάτι που θα πρέπει να σταματήσει. Και ελπίζω ότι αυτά που σας είπα σήμερα εδώ θα σας βοηθήσουν να κάνουμε ένα βήμα προς την ελευθερία. Η επιλογή της ελευθερίας έναντι της ασφάλειας είναι μια λανθασμένη επιλογή. Μπορούμε κάλλιστα να ζήσουμε με ασφάλεια και ελευθερία και δεν χρειάζεται να επικαλούμαστε τις παράνομες δραστηριότητες της NSA για να οδηγηθούμε προς την ελευθερία. Υπάρχουν νόμιμες διαδικασίες οι οποίες δεν είναι απαραίτητο να περνούν μέσα από το δαπανηρό και παράνομο πρόγραμμα παρακολούθησης της NSA. Ο κύριος Σνόντεν θα ήθελε πολύ να είναι παρόν σήμερα εδώ. Αλλά δυστυχώς για λόγους ε, απαράδεκτους δεν μπορεί. Αλλά πραγματικά ο Julian Assange, το Wikileaks, που πραγματικά τον ε, στήριξαν, τον βοήθησαν, τον βοήθησαν να περάσει στη Ρωσία, να κρυφτεί, του έδωσαν άσυλο και προστασία. Και πρόκειται πραγματικά για ανθρώπους που τον 21ο αιώνα μας βοήθησαν να στηρίξουμε την ελευθερία. Είναι οι θεματοφύλακες του κυρίου Σνόιδεν τον βοήθησαν να περάσει με ασφάλεια σε αυτό το δύσκολο ταξίδι. Για να προστατευθούν και οι δικές σας ελευθερίες και η δική μου ελευθερία, πραγματικά θα πρέπει να στηρίξουμε τις προσπάθειες του Τζούλιαν, της Σάρα και του Έντουαρτ, τα παραδείγματα που έδωσαν και αυτοί και άλλοι whistleblower, που πραγματικά μας καθοδηγούν. Of Αυτά είπε ο Edward Snowden και ευχαριστούμε πολύ την Κοινοβουλευτική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αποφάσισε να οργανώσει αυτή την ακρόαση για τους whistleblowers, για την προστασία της προσωπικής ζωής. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις και πραγματικά η ελευθερία μας εξαρτάται από τη δημιουργικότητα που θα δείξουμε έτσι ώστε να ξεπεράσουμε αυτές τις παράνομες δραστηριότητες. Και η δημιουργικότητα, όπως ξέρετε, είναι το αποτέλεσμα της περιέργειας. Και η περιέργεια είναι το αποτέλεσμα της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας της. Θα ήθελα λοιπόν πραγματικά να σας πω ότι πρέπει να βρούμε μια εξισορροπημένη προσέγγιση μεταξύ των συμφερόντων ε, των κρατικών αρχών και των υπηρεσιών για έρευνα και διερεύνηση, αλλά και της προστασίας της προσωπικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων. Δεν μπορεί να υπάρξει δημόσια συζήτηση χωρίς να υπάρχει γνώση. Και στη χώρα μου, κάποιος που βρίσκεται στη δική μου θέση, σαν νομικός και σαν ε, ειδικό ε, ο οποίος ε, υπερασπίζεται τέτοιου είδους υποθέσεις, έχει σαν αποτέλεσμα η δράση μου να αναγκαστώ να εγκαταλείψω τη χώρα μου. Αυτό βεβαίως είναι κάτι το οποίο με οδήγησε στην πολύ προσεκτική εξέταση όλων αυτών των whistleblowers, όλων αυτών που εργαζόταν στην NSA και που σήμερα βρίσκονται υπό διωγμό. Δεν είμαστε οι μόνοι βεβαίως που αναλαμβάνουμε τέτοιες υποθέσεις. Υπάρχουν πολλές υποθέσεις σήμερα οι οποίες θα πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά. Τα σύγχρονα προβλήματα απαιτούν βεβαίως σύγχρονες λύσεις και η εθνική ασφάλεια θα πρέπει να προστατευτεί με κάθε τρόπο, αλλά θα πρέπει και το κοινό να γνωρίζει ποιοι το κυβερνούν με ποιον τρόπο. Και αυτό προϋποθέτει ότι όλες αυτές οι υπηρεσίες πληροφοριών δεν λειτουργούν ανεξέλεγκτα, δεν είναι αυτοκυβερνόματα σώματα. Με τέτοιου είδους ακροάσεις νομίζω ότι μπορούμε να διαπιστώσουμε τι γίνεται. Έχετε όλοι μου, όλες μου τις ευχαριστίες και την αναγνώρισή μου για αυτά που κάνετε. Σας ευχαριστώ πολύ, Edward Snowden. Σας ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστούμε που μας διαβιβάσατε το μήνυμά του. Να περάσουμε κατευθείαν στον ε, κύριο Ντέβιτ από την ε, Transparency International της Ιρλανδίας. Ευχαριστώ κύριο Πρόεδρε και να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Είναι τιμή να βρίσκομαι εδώ μαζί με τη Τζέσλιν και με άλλους ανθρώπους που θαυμάζω απεριόριστα. Ως πρώην δημόσιο υπάλληλος και εγώ θεωρώ ότι είμαι ιδιαίτερα τυχερός διότι ποτέ δεν χρειάστηκε να ε, αντιμετωπίσω προβλήματα με τη συνείδησή μου και να έχω ηθικούς φραγμούς όπως ε, η, ε, ο Τόμας, η Άννη και άλλοι. Δυστυχώς οι πληροφοριοδότες βρίσκονται στη λανθασμένη θέση, στη λανθασμένη στιγμή. Υπάρχουν διαβλή που επιτρέπουν ε, σε αυτούς τους ανθρώπους που αναγκάζονται να επιλέξουν ε, πότε να σιωπούν ή αν πρέπει να μιλήσουν για να μπορέσουν να προασπίσουν το δημόσιο συμφέρον. Επίσης να σας πω ότι εγώ μπόρεσα να υποστηρίξω ανθρώπους οι οποίοι υπερασπίζονται αυτά τα δικαιώματα και ε, προσπαθούν να προστατεύσουν τα θεμελιώδη δικαιώματα και τον κώδικα δεοντολογίας τους. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθούμε να παρέχουμε νομική προστασία σε πληροφοριοδότες εδώ και 20 χρόνια. Πρόσφατα υπήρξε και νομοθεσία για τα θέματα αυτά και σύντομα θα δημοσιεύσουμε και μία έκθεση ε, για τα στοιχεία που έχουμε για τους whistleblowers στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης βοηθούμε, έχουμε γραμμές βοήθεια σε 15 χώρες και ε, μέχρι τώρα έχουμε πάνω από χίλιους πελάτες παγκοσμίως. Η Transparency Ireland ξεκίνησε την πρώτη γραμμή βοήθειας για θύματα διαφθοράς και whistleblowers στην Δυτική Ευρώπη και είμαστε η πρώτη γραμμή βοήθειας στη Δυτική Ευρώπη που ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια. Έχουμε γραμμές ε, τώρα πλέον στην Τσεχική Δημοκρατία, στη Ρουμανία, στο Λουξεμβούργο και θα πρέπει να πω ότι γίνεται πάρα πολύ σημαντική δουλειά και στο Ηνωμένο Βασίλειο γιατί έχουν προχωρήσει και το θεματολόγιο για νομοθεσία για τα θέματα αυτά, όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και ε, αλλού. Προσπαθούμε λοιπόν να ε, δούμε τι γίνεται, διότι υπάρχει αυτή η προϋπόθεση ότι γίνεται για να μας προστατεύσουν από την τρομοκρατία και από επιθέσεις και πολλές φορές συζητώνται το πώς ε, πληροφορίες συλλέγονται. Υπάρχουν αρκετές πληροφορίες οι οποίες δεν έχουν δημοσιευθεί για διαφόρους πληροφοριοδίτες. Θα γνωρίζετε ίσως την περίπτωση του Frank Level που μίλησε για μια υπόθεση της ε, Δανίας και της υπηρεσίας πληροφοριών για την ε, εισβολή στο Ιράκ ε, και επίσης και τις διάφορες υποθέσεις που συζητήσαμε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στην Ιρλανδία δεν υπάρχει δημόσια αντιπαράθεση ε, εδώ και 40 χρόνια, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν κάποιοι ισχυρισμοί για τα ε, ονείρα και ε, κάποιες πληροφορίες οι οποίες ήρθαν στην επιφάνεια το 1972. Αλλά έχουμε διάφορες συμπεριφορές στις δημόσιες υπηρεσίες που είναι αντίστοιχες με τους πληροφοριοδότες, τους whistleblowers στις υπηρεσίες πληροφορίας στο Ταμείο Κοινωνικής Πρόνοιας στην Ιρλανδία ε, μαθεύτηκε κάποια στιγμή ότι διαβιβάζονται πληροφορίες για τους ε, ε ασθενείς και μαθαίστηκε επίσης ότι η Ιρλανδική Ανθινομία ε, χρησιμοποιούσε ε, στοιχεία και έδινε στοιχεία σε μέλη οικογενείας ή σε άλλους αστυνομικούς. Επίσης υπάρχουν κάποια θύματα τα οποία Ε, απολύθηκαν, όπως για παράδειγμα μια δημοσιογράφος η οποία έδωσε κάποια στοιχεία για τον επικεφαλής της αστυνομίας, ο οποίος ε, είχε ε, συμμετοχή σε αντίστοιχες υποθέσεις. Η πίεση για τους whistleblowers είναι πάρα πολύ μεγάλη. Οι πληροφορίες μπορεί να είναι πολύτιμες όπως και κάθε άλλο δημόσιο αγαθό. Το θέμα είναι τι γίνεται με ε, δημοσίους υπαλλήλους, δημοσίους αξιωματούχους όταν ε, αναγκάζονται να ε, διαχειριστούν δημόσια περιουσία, συμπεριλαμβανόμενες και πληροφορίες και να πρέπει να συλλέγονται και μπορεί να υπάρχει και κατάχρηση για προσωπικά δεδομένα ή για αρχεία πολιτών. Ορισμένες φορές οι πληροφοριοδότες υποχρεούνται να δώσουν στοιχεία για κακοδιαχείριση. Οι whistleblowers όμως δεν είναι μόνοι τους. Υπάρχουν ελάχιστες δικλείδες ασφαλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρά το γεγονός ότι ε, βάσει των στοιχείων που υπάρχουν από την Ένωση για πιστοποιημένους ε, ελεγκτές απάτης, ε, τα περισσότερα στοιχεία δίνονται από whistleblowers. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι οι whistleblowers βοηθούν να εντοπίζονται κάποιες τέτοιες περιπτώσεις, ε, πολλές φορές ε, βοηθούν και να μην υπάρχουν τέτοια περιστατικά, διότι αν το γνωρίζουν ότι μπορεί κάποιος να διαρρεύσει τις πληροφορίες, μπορεί να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα και κάποιοι οι οποίοι θα μπορούσαν ίσως να ε, ε, διαπράξουν απάτη δεν το κάνουν. Υπάρχει και η Disclosure Act του 1998 μετά από μια σειρά από διάφορες αποτυχίες όπου μια περίπτωση ας πούμε όπου χάθηκαν 193 δολιές, ε, ε, ζωές συγγνώμη, ε, ή μια άλλη περίπτωση στην οποία είχαμε 500 ε, θύματα ε, τραυματισμού και 25 θανάτους θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να διαβιβάζονται διάφορες επικίνδυνες πρακτικές οι οποίες δεν ε, κοινοποιούνται καταλήλως και θα πρέπει να γίνονται γνωστές. Η Ιρλανδία είναι μία από τις λίγες περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δίνει πλήρη μέτρα και συνεχή ε, βοήθεια σε whistleblowers και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Ε, δεν προστατεύονται όμως οι whistleblowers ακόμα και στο Ηνωμένο Βασίλειο στις υπηρεσίες πληροφοριών. Ε, οι whistleblowers από κάποιους τομείς όπως για παράδειγμα στον τομέα της υγείας ή της ε, φροντίδας παιδιών ε, δίνονται κάποιες πληροφορίες, μπορούν να γίνουν καταγγελίες για απάτη ή για κακομεταχείριση παιδιών. Μπορεί κάποιο να είναι σε θέση, για παράδειγμα, να καταγγείλει κάποια περιστατικά διαφθοράς. Η διαφθορά θεωρείται ως ιδωροδικία στο δημόσιο τομέα, δημόσιο αξιωματούχο. Μπορεί να μην προστατεύονται εάν δώσουν στοιχεία για κάποιες ε, προσωπικές πληροφορίες ή προσωπικά δεδομένα. Αυτό γίνεται για παράδειγμα με τις πληροφορίες τις οποίες ε, χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες πληροφοριών ε, με λάθος τρόπο ή με παράνομο τρόπο. Επιτρέπεται να ε, καταγγέλλεται κάποιος από τους whistleblowers, όπως για παράδειγμα το αφεντικό τους ή ένας αστυνομικός, αλλά δεν προστατεύονται εάν για παράδειγμα καταγγείλουν το λάθος άτομο. Αυτοί οι περιορισμοί δεν βοηθούν την ε, δημοσίευση αυτών των πληροφοριών και ε, οι πολίτες δεν νιώθουν ασφαλείς και δεν νιώθουν ότι θα μπορούσαν να καταγγείλουν αυτά τα περιστατικά. Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν κατάλληλη αλλαγή στην νομοθεσία και θεωρούμε ότι θα πρέπει να ε, το λάβετε υπόψη αυτό όταν θα κάνετε οποιαδήποτε επίσημη πρόταση για νομοθεσία για το whistleblowing στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση στα κράτη-μέλη. Υπάρχουν τρεις βασικές αρχές τις οποίες θεωρώ ότι θα πρέπει να λάβετε υπόψη. Καταρχάς, η νομοθεσία αυτή θα πρέπει να προστατεύει όλους τους εργαζομένους, ακόμα και αυτοί που εργάζονται σε υπηρεσίες πληροφοριών ή σε υπηρεσίες άμυνας, καθώς επίσης εργολάβους, εκπαιδευόμενους, εργαζόμενους, εργοδότες, οι οποίοι θα πρέπει να προστατεύονται και από κάποιες επίσημες διαδικασίες, όπως για παράδειγμα την απόλυσή τους, αλλά και αναπίσημες διαδικασίες, όπως παρενόχληση. Ε, θα πρέπει επίσης να καταγγέλουν ε, ε, τη διαφθορά και να δίνεται τη δυνατότητα στους whistleblowers όχι μόνο να καταγγέλουν τη διαφθορά ή την απάτη, αλλά και αμέλεια, ε, παράβαση καθήκοντος, ε, η παραβίαση της αρχής της εμπιστευτικότητας, για παράδειγμα προσωπικών δεδομένων πολιτών. Και επίσης, θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλοι διάβλοι μέσω των οποίων θα μπορούν να καταγγέλλονται αυτές οι πληροφορίες και θα μπορούν ίσως να κάνουν και εσωτερική καταγγελία αλλά να έχουν και τη δυνατότητα να κάνουν και καταγγελία σε κάποιον εξωτερικά. Εάν οι πληροφορίες ε, είτε θα αποκρυφθούν είτε θεωρείται ότι δεν θα αναλάβει κανείς δράσεις ε, ή είναι ε, οι πληροφορίες δημοσίου συμφέροντος οι οποίες θα πρέπει να δοθούν ευρύτερα οι αρχές αυτές ε, σε μεγάλο βαθμό βασίζονται σε εμπειρία που έχουμε από whistleblowers και διάφορα περιστατικά να τον κόσμο. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να κάνουν εσωτερική καταγγελία ή ε, στα Υπουργεία Εσωτερικών. Αυτό λοιπόν που θεωρούμε ότι είναι αποτυχία των δημοκρατικών θεσμών είναι να μπορέσουν να τηρήσουν τις αρχές επί των οποίων έχουν θεμελιωθεί τα συστήματα ε, των υπηρεσιών πληροφοριών και οι σχετικές έρευνες που έχουν γίνει καταδεικνύουν ότι θα πρέπει να γίνεται κατάλληλη αξιολόγηση και να ελέγχεται ε, κατά πόσον δεσμεύονται για το κράτος δικαίου και να υπάρχει ανάλογη λογοδεσία. Οι πληροφορίες οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες, ε, ναι μεν θα πρέπει να λαμβάνονται, αλλά θα πρέπει και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να έχουν την ελευθερία να δημοσιοποιούν αυτές τις πληροφορίες. Ε, όπως έχουμε δει και στη χώρα μου και στην Ευρώπη θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον το οποίο θα είναι κατάλληλο ώστε να μπορεί κάποιος ελεύθερα να λένε την αλήθεια για να μπορούν να πατάξουν αυτούς που έχουν την εξουσία παρανόμω. Ευχαριστώ και να ζητήσω συγγνώμη και από τους δυο σας ε, γιατί σας ε, πιέσαμε λίγο. Υπάρχουν άλλοι εκτός από τον εισηγητή και τους κοιόδης που θέλουν το λόγο, κυρία Μορβάη, ο κύριος Μπρόνς, κυρία Σίπολ. Όλοι από ένα λεπτό. Θα ακούσουμε όλες τις ερωτήσεις. Ένα λεπτό, αλλά αυστηρότατα. Παρακαλώ να κοιτάτε τα ρολόγια σας. Κύριε Σιγητά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρίως ε, τον Γκέσλι ε, και τον Στίβεν και τον Τζον. Μιλήσατε για την ε, καλύτερη έκφραση των ανθρώπων που έχουν πράγματα να πούν ε, να δούμε περισσότερους διάβλους. Πώς ε, θα αντικατοπτριστεί αυτό στην έκθεσή μας, θα το, έκθεσή μου θα το δούμε. Αλλά στις Ηνωμένε Πολιτείε υπάρχουν επίσημοι διάβλοι για να εκφραστούν ε, οι πληροφοριοδότες και εσωτερικώς. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το εξή. Ο κύριο Σνόντεν αυτά που έκανε, τα έκανε διότι η εσωτερική διάρθρωση για τους πληροφοριοδότες δεν είναι πια ευστοχή τι ε, μπορείτε να μας πείτε γι' αυτό. Γι' αυτό έπρεπε να πει αυτά που είπε με τέτοιο δραματικό τρόπο. Και αν εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουμε να αποφύγουμε τέτοιου είδους καταστάσεις, τι θα συστήνατε. Ε, υπάρχουν ε, άλλες νομοθετικές πράξεις, όπως αυτή του Τζον Ντέβιτ που είναι άστοχες πλέον. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό. Έχετε ε, ξεφύγατε κατά 9 δευτερόλεπτα, αλλά αυτό δεν είναι προνόμιο. Έχετε 60 δευτερόλεπτα, κύριε Φως. Στα γερμανικά. Πολύ ενδιαφέροντα μας είπατε. Το ερώτημά μου έχει να κάνει με αυτό που είπε και ο συνάδελφος οι αποκαλύψεις, το λεγόμενο whistleblowing, ε, Η μόνη δυνατότητα έκφρασης είναι μέσω του τύπου ή υπάρχουν και άλλοι ανεξάρτητοι φορείς όπως ένας ombudsman που να μπορούσε να δεχτεί τις πληροφορίες χωρίς να εκτίθεται μάλιστα ο πληροφοριδότης σε κίνδυνο. Ε, διερωτώ με λοιπόν. Η Υπάρχει κάποιος τρόπος να δώσουν τις πληροφορίες στους πληροφοριοδότες χωρίς να εκτεθούν. Μας γλιτώσαμε 60 δευτερόλεπτα από τον επόμενο εισηγητή γιατί αποσιάζει η κυρία Ένστ. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομο αυτό. Θα ήθελα να επανέλθω και εγώ στο θέμα της προστασίας των ε, πληροφοριοδοτών για την έλλειψη πλήρως προστασίας μάλλον. Πώς θα έπρεπε να αντιλαμβανόμαστε τους πληροφοριοδότες. Γίνονται αντιληπτοί και τους βλέπουν οι άλλοι σαν προδότες, σαν παράνομους. Πώς αντιμετωπίζονται και μπορείτε να μας πείτε κάπως ξεκάθαρα εσείς πώς νομίζετε πρέπει να προστατεύονται αυτοί οι πληροφοριοδότες, τι κανόνες θα πρέπει να ισχύουν. Ευχαριστούμε κύριε Μορβάη, κύριος Μπρόνς και μετά έχω και εγώ μια ερώτηση. Κύριε Μορβάη, ευχαριστώ πολύ. Είναι πραγματικά συγκινητικό να ακούει κανείς το προσωπικό μήνυμα του κυρίου Σνόντεν ε, προς εμάς, αλλά προφανώς το ευχόμαστε ότι καλύτερο και είμαστε ευγνώμονες. Ελπίζω τουλάχιστον οι περισσότεροι είπε ε, ότι στην πρώτη του συνέντευξη μάλιστα ε, αυτό που φοβάται περισσότερο δεν είναι το Γκουαντάναμο και αυτό μου φάνηκε και περίεργο. Ούτε τις διώξεις, ούτε τις ποινές, αλλά την πιθανότητα αυτά που αποκάλυψε να μην ε, έχουν κανέναν αντίκτυπο. Αυτό το βρήκα πολύ ενδιαφέρον, διότι δείχνει πόσο έχει ενεργό συμμετοχή σε όλη αυτή τη διαδικασία. Πώς ε, βλέπετε την κατάστασή του σε αυτή τη χρονική περίοδο με τις ως τώρα συνέπειες. Ως δικηγόρος τι νομίζετε, τι πιστεύετε για το προσωπικό μέλλον του κυρίου Σνόντεν. Τι θα του συμβεί. Κάνουμε τίποτε ουσιαστικό για να προστατεύσουμε τα δικαιώματά του. Ευχαριστούμε κύριε Μπρόντσο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να είναι προστατευμένη από τα επικριτικά σχόλια σε ό,τι αφορά την προστασία των πληροφοριοδοτών. Υπάρχουν εργαζόμενοι που τους προστατεύουν υπηρεσιακές τους καταστάσεις ε, και αυτό ισχύει και για το με τον κανονισμό του 2004. Όμως ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέλησε υπάλληλό τη ε, μέσα στην ίδια χρονιά κιόλας γιατί κατηγορήθηκε για, πληροφοριοδο πληροφοριοδότης. Με η κυρία Ανδρέα Σεν, η οποία όταν έγινε μέλος αυτού του σώματος, ε, είχε αρκετές δυσκολίες στην αρχή. Βλέπουμε ότι ήδη έχουμε και άλλα περιστατικά με κατοίκον έρευνες και μάλιστα τελείως παρανόμες χωρίς ένταλμα, χωρίς να υπάρχει καν αιτιολόγηση. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει οργανωμένη συνωμοσία, αλλά υπάρχει διαρκώς η εντύπωση ότι διάφορες οργανώσεις, ιδίως οι μεστικές υπηρεσίες, ακολουθούν ε, τις ε, δικές τους ε, ατζέντες τα τελευταία χρόνια και οι κυβερνήσεις δυσκολεύουν να δράσουν κατά των πληροφοριωτών. Οι συντάκτες των ε, ε, νομοσχεδίων αυτών δεν ε, λαμβάνουν επαρκή μέρημνα για να προστατεύσουν ε, τις κυβερνήσεις, τους νομοθέτες που τελικά δεν καταφέρνουν να δώσουν τη σωστή προστασία. Πώς θα μπορέσει να... Ευχαριστώ. Εγώ θα κάνω την τελευταία ερώτηση, ιδιαίτερα όσον αφορά αυτό που είπε η κυρία Ρόντεκ για την προστασία των δημοσιογράφων και όλων των ε, υπολείπων ε, ατόμων που αποφασίζουν να, να αποκαλύψουν πληροφορίες. Τι έχετε να πείτε για τις υπόλοιπες κατηγορίες πληροφοριοδοτών. Κοιτάξτε, εγώ σαν νομικός, ναι, νιώθω ασφαλής, καθότι γνωρίζω τι διαδικασίες πρέπει να ακολουθήσω. Αλλά σε καμία περίπτωση όταν με παίρνουν τηλέφωνο οι πελάτες δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με ηλεκτρονικό τρόπο, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μετά από το τηλέφωνο, του συναντώ, μιλάμε, προσέχουμε, Όλες οι χρηματικές ε, συναλλαγές γίνονται χωρίς να περάσουμε από κανένα ηλεκτρονικό μέσο. Καταλαβαίνετε ότι χρησιμοποιούμε μεθόδους ε, εμπόρων ναρκωτικών. Τώρα, τι λύσεις, τι λύσεις μπορεί να προτείνω. Καταρχήν, πιστεύω ότι χρειάζεται μια μεταρρύθμιση αποτελεσματική και βεβαίως όσον αφορά το Protection Enhancement Act χρειάζονται κριτήρια που να μην βασίζονται μόνο στην εθνική ασφάλεια, αλλά χρειάζονται κάποιοι μηχανισμοί οι οποίοι θα επιτρέπουν στο μέλος στο μέλλον, συγγνώμη, τους whistleblowers να ξεκινήσουν κάποιες διαδικασίες προστασίας. Και βεβαίως εδώ προκύπτει το ερώτημα και εδώ υπάρχει η οδηγία 19 στην οποία είπε ο πρόεδρος ότι μπορεί να προστατεύσει τον Edward Snowden. Όχι, αυτό δεν ισχύει σε καμία περίπτωση, καθότι η οδηγία αυτή 19 δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην περίπτωση του Snowden. Από ό,τι φαίνεται, ο τύπος είναι ο μόνος τρόπος να βγουν προς τα έξω όλα αυτά τα μηνύματα. Αλλά, αλλά, Σήμερα τα αποδεικτικά στοιχεία αυτά δεν μπορούν μονίμως να περνούν από τον τύπο. Ο κύριος Σνόντεν θέλει σήμερα να ακολουθήσει μια νόμιμη διαδικασία, μια επίσημη διαδικασία και να βρεθεί αντιμέτωπος με κάποιο φορέα κρατικό, κυβερνητικό, με τον οποίο να μπορέσει να παρουσιάσει όλα του τα επιχειρήματα. Ναι, όντως χρειάζεται μια μεταρρύθμιση, πρέπει να βρεθούν τρόποι να αλλάξει η κατάσταση. Στην αρχική του δήλωση ο κύριος Νόντεν είπε ότι θα είναι πάρα πολύ κρίμα αν μετά από όλα αυτά δεν γίνει τίποτα, δεν αλλάξει τίποτα. Η σημερινή ακρόση, παραδείγματο χάρη. Και ξέρω ότι είναι μια ολόκληρη σειρά ακροάσεων που έχετε οργανώσει, μου δίνει μεγάλη ελπίδα. Μεγάλη ελπίδα. Τώρα, το μέλλον. Το μέλλον ε, του κυρίου Σνό δεν εξαρτάται από την ε, βούληση κάποιων ε, υπερδυνάμεων να δεχτούν ότι εδώ υπάρχει μια πολιτική δίωξη η οποία βασίζεται στις πολιτικές του πεπιθήσεις. Δεν πρόκειται λοιπόν εδώ για προστασία εγκληματία και αυτά που προσάπτουν στον κύριο Σνόδεν σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να μπουν σε καμία διαδικασία προσαγωγής ποινική. Οι πράξεις του δεν είναι εγκληματικές πράξεις. Είναι απλώς η έκφραση ελευθερίας και η βούληση να ζήσει ελεύθερα στη χώρα. Και όπως ξέρετε Το πιο σημαντικό σήμερα είναι να χαρακτηριστεί σαν whistleblower ο κύριος Σνόντεν και όχι σαν προδότης και σαν κατάσκοπος. Σήμερα βεβαίως βλέπουμε να επικρατούν ε, στερεότυπα, να επικρατούν προκαταλήψεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ επικίνδυνες και για τη χώρα μας, αλλά και για όλο τον κόσμο. Πολύ σύντομα, γιατί δεν θέλω να καθυστερήσουμε άλλο, γιατί ήδη έχουμε περάσει ε, το χρόνο μας, έχουμε υπερβεί το χρόνο. Μήπως θα μπορούσατε να διευκρινίσετε λίγο καλύτερα το τελευταίο αυτό που είπατε για να απαντήσετε και στην ερώτηση της κυρίας Έρνστ. Αν ε, χρησιμοποιήσει όλες τις επίσημους διάβλους ε, που του επιτρέπονται, αυτό σημαίνει ότι αυτόματα θα ισχύουν νόμοι κατά της αντακατασκοπίας και τρομοκρατίας απολύτως. Εάν είχε περάσει από τους επίσημους διάβλους, ε, μπορώ να σας διαβεβαιώσω, διότι εκπροσωπούσα και τον Τόμες Ντρέικ, ο οποίος μίλησε προηγουμένως, επειδή είχε πάει ε, στους επίσημους ε, διάβλους της NSA, σε ένα γενικό επιθεωρητή και σε δύο μέλη της Γερουσίας και έκανε αποκαλύψεις, όχι μόνο δεν έγινε τίποτα, αλλά και το Υπουργείο Άμυνας δεν ναι, μεν θεώρησε ότι υπήρχαν λόγοι για τις καταγγελίες τους, αλλά έκανε αμέσως απόρριτη την έκθεση ώστε να μην τη δει κανένα και μετά έδωσε το όνομα και του Τόμας και, σε άλλους, ε, και άλλων δύο πληροδοτών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για να ε, ε, τους δικάσουν. Ουσιαστικά οι άνθρωποι που έπρεπε λοιπόν να τους προστατεύσουν ε, τους πέταξαν στα σκουπίδια. Λοιπόν, ο, ο Σνόντιν επειδή είδε τι έγινε με τον William Μπένι, με την Τζέλσι Μάνινγκ και είδε ότι όταν πήγαν από τους επίσημους διάβλους βρέθηκαν ε, κατηγορούμενοι για κατασκοπία, ε, γνώριζε πάρα πολύ καλά τι θα μπορούσε να συμβεί και στην περίπτωσή του. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Ντέβιτ. Τέσσερις ερωτήσεις μου ετέθησαν. Με ρώτησαν ε, τι θα μπορούσε να υπάρξει στην ομοθεσία ώστε ε, να προστατεύονται οι whistleblowers ε, των υπηρεσιών πληροφοριών. Καταρχάς, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υπεραμεινθούν του αυτού τους ενώπιον του δικαστηρίου, θα πρέπει ε, να υπάρχει διασφάλιση ότι δεν θα απολυθούν ή δεν θα τους παρενοχλήσουν άλλοι εργαζόμενοι και ότι θα απολαμβάνουν άλλα τα δικαιώματα των υπολείπων εργαζομένων. Θα πρέπει επίσης ε, να υπάρχει δυνατότητα υπεράσπισης ε, κατά ε, ποινικών διαδικασιών και να αποδεικνύεται ότι όντως έχουν δράσει βάσει της νομοθεσίας. Και υπάρχουν αυτές οι ρήτρες ασφαλείας στην Ιρλανδική νομοθεσία. Παρέχεται ασυλία αρκεί να έχει τηρηθεί η νομοθεσία. Επίσης, και αυτό είναι σημαντικό, θα πρέπει οι whistleblowers να γνωρίζουν ότι οι πληροφορίες που παρέχουν ε, είναι πληροφορίες επί των οποίων θα υπάρξει δράση. Ε, βάσει αρκετών ε, φορέων έρευνας, ένας από τους βασικούς ανασταλτικούς παράγοντες που δεν επιτρέπουν στους whistleblowers να δώσουν πληροφορίες είναι και ο λόγος για τον οποίο δεν αποκαλύπτουν τα στοιχεία είναι γιατί φοβούνται ότι δεν θα γίνει τίποτα και θα πρέπει να υπάρχει νομική υποχρέωση για όσους λαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες να τις εκμεταλλεύονται. Ο κύριος Βος ρώτησε κατά πόσον οι πληροφορίες θα πρέπει να διαβιβάζονται εσωτερικώς. Απολύτως ε, ναι είναι η απάντηση στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία όπως και σε άλλες χώρες του κόσμου, στη Νέα Ζηλανδία και στην Νότια Αφρική υπάρχει μέρημνα ώστε οι εργαζόμενοι να καταγγέλουν εσωτερικά κάποιες πληροφορίες πρέπει να λογοδοτούν στο διευθυντή τους ή στον εργοδότη τους εκτός αν θεωρούν ότι υπάρχει κάποιος λόγος, υπάρχει κάτι δημοσίου συμφέροντος εντός κάποιου οργανισμού ε, ή σε κάποιο μέλος του κοινοβουλίου θα πρέπει να καταγγέλλονται εκεί ή σε κάποιο δημοσιογράφο. Ξέρω ότι είναι ρητορική ερώτηση της κυρίας Έρνστ αλλά συμφωνώ μαζί σας απόλυτα και με τα όσα είπε Τζέλσιν. Δεν νομίζω ότι είναι ήρωες αυτοί οι άνθρωποι ε, και το να τους να, να λέμε ότι είναι ήρωες ή προδότες δεν βοηθά σίγουρα τα όσα λένε. Ξέρω ότι ήταν η ρητορική ερώτηση σας. Από νομικής πλευράς όμως ρωτάω. Δεν βοηθα σιγουρα οσα λενε ξερω οτι ηταν η ρητορικη ερωτηση σας απο νομικης πλευρας ομως ρωταω δεν να ξέρω από νομικής απόψεως πώς το καλύπτεται. Ο, ο whistleblower πώς καλύπτεται, με ποια νομική βάση. Είναι σαφής η ερώτηση. Εξαρτάται από το ποιος ε, ε ξεκινά την ιστορία. Πρέπει να μπορούμε να τους βοηθήσουμε και χρειάζονται νομική προστασία. και επίσης σε διεθνούς και διαπεριφερειακούς οργανισμούς χρειάζονται προστασία whistleblowers, όχι μόνο σε εθνικές υπηρεσίες. Υπήρχε και κάποια άλλη ερώτηση, ζητή, συγγνώμη κυρία Σίπχολ, δεν τη θυμάμαι μπορείτε να είστε βέβαιος ότι θα υπάρξει δράση από πλευρά κυβερνήσεων για την προστασία των whistleblowers, ιδία στην ε, περίπτωση των μυστικών υπηρεσιών, διότι μπορεί να συμμετέχουν ή να μην είναι διατεθειμένοι να αποκαλύψουν τα όσα συμβαίνει. Νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτάται ε, τι θα ζητήσει ε, η πολιτεία. αν οι πολιτικοί θεωρούν ότι δεν υπάρχει ανάγκη για αυτόν, σίγουρα θα το αποκρύψουν. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές μας που ήταν εδώ σήμερα. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και για τις αποδείξεις και τα στοιχεία που μας δώσετε. Η Πρόεδρος ευχαριστεί και τους Διερμηνείς για την καθυστέρηση και να ευχαριστήσω και το κοινό γιατί ήταν τόσο υπομονητικό και έμεινε εδώ μέχρι τέλους. Ολοκληρώνω τη σημερινή συνεδρίαση. Ευχαριστώ στο επανειδή.